So, Καθίστε παρακαλώ στις θέσεις σας. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στη ε, συνεδρίαση μας τον Αντιπρόεδρο και Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό, τον κύριο Χωακίν Αλμούνια. Καλώς ήρθατε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είσαστε στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Δεν είσαστε τακτικός επισκέπτης, ε, αλλά έχετε ξανάρθει και το γνωρίζετε ότι ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα σε σχέση με τις επιπτώσεις στους καταναλωτές της ε, αρμοδιότητάς σας για τον ανταγωνισμό για θέμα για το οποίο θα μας μιλήσετε και γνωρίζουμε ιδιαίτερα όσον αφορά την ανακοίνωση σε σχέση με την οικονομία. Υπάρχει αναφορά σε θέματα ανταγωνισμού που μας ενδιαφέρουν άμεσα και για, για το λιανικό εμπόριο που μας απασχολεί και αυτό πάλι εδώ εντάσσεται και ενδιαφερόμαστε να μας πείτε τι έχετε υπόψη για το πρόγραμμα εργασίας σας και ίσως θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το ρυθμό εργασίας μας ώστε να συντονιστούμε καλύτερα. Καλώς ήρθατε. Με ιδιαίτερη χαρά σας δίνω τον λόγο. Ανοίγει ο πίνακας αγορητών για συναδέλφους που θα ήθελαν να παρέμβουν με ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ εσάς μέλη αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πράγματι να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Χάρμπορ για την ευγενική πρόσκληση να προσέλθω. Ως Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό για πρώτη φορά έχω την ευκαιρία αυτό το αξίωμα μου να προσφωνήσω τα μέλη της Επιτροπής σας και να εκθέσω τις απόψεις μου και με ιδιαίτερη ευχαρίστηση το κάνω. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για το οικονομικό παρασκήνιο και οικονομικά στοιχεία φυσικά δεν είναι ενθαρρυντικά τα μαντάτα για την οικονομία. Θα έχουμε μια ήπια ύφεση τους επόμενους μήνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύνολο του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει στάσιμο σε χαμηλά επίπεδα. Και βλέπουμε ότι αυτό έχει τον αντίκτυπό του στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι ιδιαίτερα είναι ανεργοί και πλήττονται από την ανεργία και αυτό είναι κάτι το οποίο πλήττει γενικότερα και τους εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ύφεση. Μετά από πέντε χρόνια η επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη είναι η πιο επίγουσα προτεραιότητα για όλους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε αποτελεσματικά μέτρα για να σταθεροποιήσει μια ενδυνάμει ολέθρια κατάσταση το 2007-2008. Τότε φυσικά η αντίδραση ήταν η σταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού τομέα. Τα προηγούμενα δύο χρόνια κατεδείχθη ότι οι ισολογισμοί στο δημόσιο ήταν πραγματικά είχαν δημιουργήσει μια ανέφικτη, πολύ δύσκολη κατάσταση, κατάσταση και για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση ελήφθησαν ριζοσπαστικά μέτρα για τη δημοσιονομική εξυγίανση και τον ισοσχερισμό και για τη διασφάλιση της νομισματικής ένωσης. Ε, και σε σχέση με τη δημοσιονομική διαχείριση υποστηρίζουμε στον τομέα του ευρώ όλες αυτές τις προσπάθειες. Όλα αυτά ήταν αναγκαία μέτρα αλλά επέβαλαν σημαντικές περικοπές στις κυβερνητικές δαπάνες την στιγμή που η μόχλευση σε σχέση με την εξωτερική και εσωτερική ζήτηση είναι πολύ χαμηλότερη και όλοι σχεδόν έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα χρειάζεται λιτότητα, αλλά η λιτότητα δεν αρκεί, δεν επαρκεί. Η επιτυχία των πολιτικών μας εξαρτάται από την ικανότητα της Ευρώπης να επιστρέψει στην πραγματική αυθεντική ανάπτυξη οικονομικά. Το ερώτημα είναι από πού θα προέλθει αυτή η ανάπτυξη. Δεν ε, είναι δυνατόν να έχουμε ακριβέ πολιτικέ με δαπάνε δημόσιε τεράστιε, αλλά υπάρχουν εναλλακτικέ λύσει. Μία από τι πιο αποτελεσματικέ δυνατότητε για την αύξηση τη ε, ε, οικονομικής μας ε, δύναμης ε, είναι πολύ λίγο δαπανηρή. Η ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, σε αυτό αναφέρομαι, που είναι το στοιχείο το οποίο δεν έχουμε εκμεταλλευτεί επαρκώς και είναι ο κινητήρας για ανάπτυξη. Πρέπει να ολοκληρωθεί, είναι μια ενιαίες αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, Τεράστι, τεράστιος αριθμός επιχειρηματιών συναθρίζεται σε αυτό το πλαίσιο Τίποτα δεν θα έδινε μεγαλύτερη ανάπτυξη από την ολοκληρωμένη αυτή οικονομική, ας το πω έτσι, πραγματικότητα σε ένα μέσο για να το εκμεταλλευτούμε, για να σημειωθεί ανάκαμψη. Σήμερα θα σας αναφέρω πώς μπορεί η πολιτική ανταγωνισμού να απελευθερώσει αυτό το ε, δυναμικό, να το απελευθερώσει ώστε μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να στραφεί στην πορεία της ανάπτυξης. Όταν έχουμε <clears throat> αποφάσεις για τον ανταγωνισμό που αντανακλώνται στις, ε, στους τίτλους εφημερίδων ή μπορεί να είναι απαγόρευση κάποιων συγχωνεύσεων, ε, συμπράξεων κτλ. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι προσπάθειές μας για τέτοιου είδους ε, αποφάσεις οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και βοηθούν τα δημόσια κονδύλια να χρησιμοποιούνται καλύτερα. Όλα αυτά λυθεύουν βέβαια, αλλά υπάρχουν και περισσότερα στοιχεία. Η πολιτική ανταγωνισμού έχει ευρύτερε συνέπειε για την οικονομία. Συχνά παραπληρωματικά ή συμπληρωματικά δρά στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντί της επίτευξης των οικονομικών στόχων. Μέσω ρυθμίσεων εσείς, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες, μπορείτε να άρετε τα εμπόδια, τα προσκόμματα και τους φραγμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτές οι πολιτικές δεν θα ήταν αποτελεσματικές αν επιτρεπόταν στις εταιρείε να κάνουν ό,τι θέλουν και να παρακάμπτουν αυτές τις ρυθμιστικές διατάξεις και ε, ρυθμίσεις. Το βλέπουμε αυτό συχνά, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μια διαθρωτική επιδείνωση σε κάποια εταιρεία ή όταν ανταγωνιστικά έχουν κάποιους ε, νέους ανταγωνιστές απέναντί τους. Έχουν μια αντίδραση που μπορεί πραγματικά να αποβεί εις βάρος ε, καινοτόμων ε, κερδοφόρων επιχειρήσεων και μπορεί να είναι ευλαπτική σε, στο τμήμα ολόκληρων βιομηχανιών, βιομηχανικών κύκλων. Γι' αυτό πρέπει να αντισταθούμε έναντι εκείνων που θέλουν να συστήσουν η ποιότερη πολιτική για τον ανταγωνισμό. Δεν θα έπρεπε να περιορίζονται οι προσπάθειές μας για αποτελεσματικές αγορές. Δεν πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα να υπονομευθεί η ανάκαμψη. Αντίθετα, πρέπει να εντείνουμε τον αγώνα κατά των πολιτικών που βαίνουν κατά του ανταγωνισμού και να έχουμε ένα πλαίσιο αυστηρό. Τώρα θα ήθελα να καταδείξω με κάποια συγκεκριμένα χειροπιαστά παραδείγματα πώς ε, το έργο μας αυτό μπορεί να προχωρήσει και να βοηθήσει. Ας ξεκινήσουμε με την αρχή της κρίσης στον χρηματοοικονομικό τομέα. Αν θέλουμε να προαγάγει την οικονομική ανάπτυξη η πολιτική ανταγωνισμού, πρέπει να βελτιώσει την, προσπέλαση, την προσπελασιμότητα ε, στου τομεί εκείνου που είναι θεμελιώδει για την προώθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι οικονομικέ υπηρεσίε είναι το καύσιμο της, ε, του κινητήρα της οικονομικής μηχανής για να δουλεύει σωστά. Αυτός είναι καθώς λόγος να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην αγορά και για τις υπηρεσίες αυτές. Παράδειγμα, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών είναι υποαναπτυγμένες στην Ευρώπη. Οι λόγοι για αυτό είναι διάφοροι και διάχυτοι. Όμως έχουμε και την, τις, τους δισταγμούς πολλών χρηματοοικονομικών ε, θεσμών να εγκαταλείψουν πρακτικές του παρελθόντος. Τον προηγούμενο Σεπτέμβριο 2011 ξεκίνησε μια εξέταση σε σχέση με το ε, Ευρωπαϊκό Σώμα Πληρωμών για να εξετάσουμε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τις πληρωμές στο διαδίκτυο ηλεκτρονικά. Ιδιαίτερα ανησυχούμε η, διάθεση, η διαδικασία τυποποίησης δεν είναι αρκετά ανοιχτή και ανοιχτά διαφανής και μπορεί κάποιες υπηρεσίες να αποκλείονται ή κάποιοι πάροχοι υπηρεσιών να αποκλείονται από την αγορά. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα είναι απόλυτα ανοιχτές αυτές οι διεργασίες γιατί τους συμμετέχοντες στην αγορά ώστε να μπορούν να αντλήσουν ωφέλη η αγορά υπηρεσιών και στις πληρωμές ε, έχουμε, βλέπουμε ότι βρίσκεται όπως και άλλα πεδία ε, χωλένων. Από τον συνάδελφο Μπαρνιέ ξεκινήσαμε μια προσπάθεια πράσινου βιβλίου να δούμε τι είναι εκείνα τα οποία παρακολύουν την ολοκλήρωση των αγορών πληρωμών στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα καθορίσουν το εύρο και τις ρυθμιστικές εκείνες παρεμβάσεις και προτάσεις που θα γίνουν. Και σας ενθαρρύνω εσάς Πρόεδρε να συμμετάσχετε σε αυτές τις διαδικασίες διαβούλευση. Χρειαζόμαστε ένα μείγμα ρυθμιστικών πολιτικών και πολιτικής ε, συμμόρφωσης για τα θέματα ανταγωνισμού, ώστε να πάψουν οι αρνητικές πρακτικές και να ανοίξουν ε, οι πανευρωπαϊκές διεργασίες πληρωμών σε όλους όσους εμπλέκονται οικονομικά στην Ευρώπη. Η πολιτική ανταγωνισμού θέλει να προωθήσει την ανάπτυξη και να ε, επιταχύνει τις διαδικασίες. Οι αγορές ε, θα πρέπει να είναι έτσι πιο δυναμικές ε, και πιο φιλικές στους χρήστες όταν εκείνοι εμπλέκονται και θέλουν να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά. Δεν θέλουμε να έχουμε τεράστιους μηχανισμούς ή γίγαντες που θα προστατεύονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο ή στο εθνικό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι ποτέ αυτό το πρότυπο ήταν επιτυχές, έστω και στο παρελθόν. Ιδιαίτερα σήμερα δεν, ε, μπορεί, δεν προσάδει σε μια τεχνολογική επανάσταση ένα τέτοιο πρότυπο με ταχύτατες αλλαγές, ελαστικότητα και αποτελεσματικότητα που απαιτούνται. Να υπενθυμίσω την πρόσφατη απαγορά, απαγόρευση με μεταξύ της ε, ε, γερμανικής τραπέζας και του και τις ε, επιχείρηση ε, που απαγορεύτηκε να συγχωνευτεί. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο απαγορευτικούς όρους και από πλευράς ε, όρων επιτοκίων. Οι δύο εταιρείε θα κατήχαν πάνω από 90% της αγοράς. Το αντίτιμο της δημιουργίας ενός ευρωπαίου πρωταθλητή δεν μπορεί να είναι η δημιουργία ενός μονοπωλίου που θα υπαγορεύει στους άλλους τους όρους συναλλαγών και λειτουργίας τους δεν θα υπήρχε καμία αποτελεσματικότητα σε μια τέτοια συγχώνευση. Καμία επιτυχία που δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί μέσω τεχνολογικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των άλλων εμπλεκόμενων στην αγορά. Το μονοπόλιο θα ήταν ιδιαίτερα επωφελές για τους μεριδιούχους, αλλά θα έπλητε εκατομμύρια καταναλωτές. Με την απαγόρευση διασφαλίσαμε την επιβίωση αποτελεσματικών παικτών στην αγορά που θα μπορούσαν να αποβούν προς όφελος των καταναλωτών. Ιδιαίτερα πιστεύω ότι έχοντας διαφορετικούς παίκτες στο παιχνίδι θα συνεισφέρει οι αγορές να είναι πιο αποτελεσματικές και διαφανείς. Καμιά φορά η ύπαρξη Μεγάλο αριθμό, όμως ε, παικτών δεν διασφαλίζει υψηλό βαθμό ανταγωνισμού χωρίς αυστηρή εφαρμογή κανονισμών και διατάξεων. Γι' αυτό συμφωνήσαμε να υπάρχει εξέταση των μέτρων antitrust αντί κατά των καρτέλ και μονοπωλίων σε αυτό το πεδίο. Ιδιαίτερα όσον αφορά και τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και τις, ε, τους ε, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τράπεζες κτλ. Ανησυχία μας, μέλημά μας είναι ότι εταιρείε ε, οι οποίες θα έχουν ε, παραβεί τέτοιου ε, κανόνες θα πρέπει να τιμωρούνται έχοντας υπόψη τον μεγάλο όγκο των ε, συναλλαγών στα παραγωγά και τον κέριο ρόλο που διαδραματίζουν αυτά τα προϊόντα στην διαχείριση κινδύνων, οποιαδήποτε χειραγώγηση θα μπορούσε να συνεπάγεται τεράστιο κόστος εις βάρος της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και οι μέτρα και μέσα πολιτικής ε, για τον ανταγωνισμό πρέπει να δράσουν προληπτικά να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Όπως προανέφερα, η καινοτομία είναι πηγή ανάπτυξης και ανταγωνισμού και ιδιαίτερα όσον αφορά την καινοτομία, αμέσω σκεφτόμαστε την ψηφιακή οικονομία. Πώς μπορεί η πολιτική των ανταγωνισμό να βοηθήσει ώστε η ψηφιακή ατζέντα να επιτευχθεί και η καινοτομία στις δράσεις να επιτευχθεί όσον αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020. Πολλές φορές έχω εκφράσει την απογοήτευσή μου, διότι χωλένουμε στην ψηφιακή επανάσταση στην Ευρώπη. Η συνάδελφός μου Νέλη Κρούς επαναλαμβάνει αυτές τις ιδέες επανειλημμένα έχει προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να άρει τις στενοπούς και τα εμπόδια που υπάρχουν στην Ευρώπη που καθυστερούν την ανάπτυξη αυτού που θα έπρεπε να είναι το επίκεντρο στην Ευρώπη η καινοτομία και ανάπτυξη. Αλλά ας ξεκινήσω από την, από αρχή. Η απελευθέρωση του τομέα, τομέα τηλεπικοινωνιών το 1990 παραμένει μία από τις επιτυχείς ιστορίες της Ευρώπης. Όμως δεν θα έπρεπε να υπεκφεύγει των ελέγχων όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Τα οικονομικά ωφέλη από αυτή την απελευθέρωση, την ε, απελευθεροποίηση πρέπει να διασφαλιστούν σε σχέση με την, το πρόστιμο 127 εκατομμυρίων που επευλήθη ε, σε μια τέτοια περίπτωση στην Πολωνία έχουμε και άλλες ε, ε, διακριβώσεις που γίνονται για τέτοιες παραβάσεις και παραβιάσεις που αφορούν στη Σλοβακία, Ισπανία, Πορτογαλία τέτοιους παρόχους υπηρεσιών στα θέματα της τηλεπικοινωνίας. Πρέπει να προχωρήσουμε, να επιτευχθούν οι στόχοι στην τηλεπικοινωνία. Δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί αυτό το φάσμα και όσον αφορά το όφελος ούτε σήμερα ούτε για τις επόμενες γενναίες. Η πρόσβαση είναι σημαντική υπόθεση και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές. Γι' αυτό επιτηρούμε τις, τα, τις ε, διεργασίες και έχουμε αναπτύξει νέες ε, διεργασίες ε, για όλα αυτά. Έχουμε ήδη ανακοινώσει προς όλους αυτούς ότι θα διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να δρουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εγκυμονεί κινδύνους η δράση τους εις βάρος των άλλων. Οι τεχνολογίες, οι μελλοντικές τεχνολογίες θα πρέπει να μπορέσουν να ανοίξουν τις ε, κλειστές θύρες ε, και να δράσουν σωστά. Όμως ε, θα υπάρχει πειρασμός για εκείνους που έχουν πριτανεύοντα ρόλο στις αγορές. Κι όμως οι αγορές είναι το δυνατόν πιο καινοτόμες όταν είναι πιο ανοιχτές και διαφανείς. Γι' αυτό η πολιτική ανταγωνισμού θέλει να περιορίσει τον ρόλο του δεσπόζοντος ε, ε, στην αγορά, της ε, πριτανεύουσας θέσης κάποιων στην αγορά. Η απόφαση που ελήφθη πέρσι είναι μια σημαντική, ένα σημαντικό ρώσιμο. Είπαμε ότι τα προϊόντα της νέας εταιρείας θα συνεχίσουν να είναι στην αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Η διαλειτουργικότητα συνδέεται στενά σε σχέση με τη χρήση κατάχρηση παραβίαση των ευρεσιτεχνιών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακολουθούμε σε σχέση με τις εξελίξεις και τις ευρεσιτεχνίες της εξελίξης. Είναι σαφές για μένα ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε ρυθμιστικά όταν ε, χρησιμοποιούνται ευρεσιτεχνίες στρατηγικά για να τροχοπεδηθούν ε, οι ανταγωνιστές κάποιων. Αυτό θα ήταν εις βάρος αυτού του συστήματος ευαισθητεχνιών που πρέπει να είναι κίνητρο και όχι τροχοπέδι. Αυτό είναι η διαδικασία που ξεκινήσαμε, η προσφυγή κατά της Samsung που μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους ευρεσιτεχνίες ε, καταχρηστικά και πρέπει να δούμε τους ε, άδικους όρους ε, ενώ πρέπει να μην χρησιμοποιείται στρέβλωση της αγοράς. Είναι σημαντικές οι προδιαγραφές διότι διαφορετικές συσκευές μπορούν να είναι συμβατές μεταξύ τους όταν υπάρχει μια κοινά συμπεφωνία αποκομιδογεννημένη τεχνολογία και η δημιουργία και το κόστος ενός ε, εφιούς τηλεφώνου χρειάζονται πάρα πολλά, πολλές ευαισθητεχνίες οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν ιδιαίτερη εξουσία και η εταιρεία που έχει τέτοιου είδους ευρεσιτεχνίες μπορεί πραγματικά να έχει στα χέρια της να πάρει στον έλεγχό της ολόκληρα τμήματα, παιδεία βιομηχανικά και επιχειρησιακά. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να βρίσκεται ως όμοιρος κανείς στα χέρια τέτοιων ε, υπηρεσιών. Έχουμε αντίστοιχε περιπτώσεις όσον αφορά την Μοτορόλα και θα τις εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς. Θα ήθελα τώρα για τη συζήτηση αυτή να αναφέρω τι προετοιμάζω για την μεταρρύθμιση των κρατικών επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων. Όμως αυτό ίσως θα παράτηνε υπερβολικά την παρέμβασή μου. Αν ενδιαφέρεστε μπορώ να σας διαθέσω αυτά τα στοιχεία ε, κατηδίαν υστερότερα. Όπως ανέφερα η μεταρρύθμιση της πολιτικής ανταγωνισμού θα συνεχίσει να είναι ένα στοιχείο κλειδί που έχει σημασία κλειδιού για τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Ε, όσον αφορά τις ε, εταιρείε. Ε, που δεν θα πρέπει να κλείνουν τις ε, πόρτες και τις οδούς για τις πιο ανταγωνιστικές είναι θεμελιώδης η σημασία του ανταγωνισμού για μια αποτελεσματική και τη δημιουργία αποτελεσματικής ε, ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς. Δεν θα μπορέσει όμως με διατάγματα να ολοκληρωθεί η ενιαία εσωτερική αγορά. Οι ρυθμίσεις και οι διατάξεις είναι κανόνας και πρέπει εμείς ως αρμόδιοι για την πολιτική ανταγωνισμού να μεριμνήσουμε αυτές οι διατάξεις και ρυθμίσεις να είναι σεβαστές. Είναι ένα αποτελεσματικό μέσο αυτό και πρέπει να δούμε ότι δεν κοστίζει τους Ευρωπαίους φορολογούμενος, ε, τίποτα. Μόνο θετικά αποτελέσματα παράγει και δεν είναι καμία επιβάρηση. Γι' αυτό η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα οποιασδήποτε πολιτικής ε, για την ανάκαμψη και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ολοκληρώνω. Το 2010 ο τότε Μάριο Μόντι, ο Επίτροπος, ε, προετοίμασε μια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ξεκίνημα της ενιαίας αγοράς. Σήμερα είναι Πρωθυπουργός τη Ιταλία. Σε αυτή την έκθεση ανέφερε ότι θα πρέπει να μην υπάρχει φθήνουσα υποστήριξη για την ενιαία εσωτερική αγορά είπε είναι λιγότερο δημοφιλής η εσωτερική αγορά σήμερα, την οποία όμως χρειάζεται περισσότερο από ποτεδήποτε η Ευρώπη. Δύο χρόνια αργότερα νομίζω πρέπει να θυμόμαστε και να κρατάμε αυτά τα όσα είπε ο Μόντι. Θα είναι επικίνδυνο να πορευθούμε προς την οδό του εθνικισμού και προστατευτισμού. Η πορεία μας πρέπει να είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς μια πορεία ανοιχτή, ανοιχτής αγοράς με καλές θετικές ρυθμίσεις για μια ανοιχτή αγορά προς όλους. Η πολιτική διαγωνισμού έχει τεράστια σημασία για όλα αυτά, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δύναμη και τις νομικές ε, αρμοδιότητες και ικανότητες για να αυτοπροστατευτούν έναντι καταχρηστικών ε, πρακτικών. Διότι αυτές είναι οι μικρές εταιρείες που θα ξεκινήσουν οι νέοι άνθρωποι και αυτές πρέπει να έχουν μια ευκαιρία να επιβιώσουν σε αυτή την αγορά. Ευχαριστώ. Well, thank you, Commissioner, very much indeed. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε ευρύτατο το φάσμα που καλύψατε στην ομιλία σας. Θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις, νομίζω. Όπως γνωρίζετε αυτή η Επιτροπή επίσης είναι στην πρώτη γραμμή μαζί με τον Μάριο Μόντι. Προωθούμε τη σημασία της ενιαίας αγοράς και προωθούμε και την, την πράξη για την ενιαία αγορά που ήταν μία από τις ιδέες μας μαζί με τον Μάριο Μόντι. Προσβλέπουμε σε συνεργασία μαζί σας πάνω σε αυτό και στην ε, αντιμετώπιση κάποιων άλλων θεμάτων όπου βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη ανταγωνισμού για τους καταναλωτές ή απογοήτευση για τους καταναλωτές που δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα ωφέλη της ενίας αγοράς. Κάνουμε σχετικά μια μελέτη για τις 20 ανησυχίε των πολιτών. Αρκετές από τις ανησυχίε είναι η μη δυνατότητα που έχουν οι πολίτες να αγοράσουν προϊόντα μέσω ιστοσελίδων κλπ. Και νομίζω ότι αυτό θα ανακύψει από τις ερωτήσεις που υποβληθούν. Έχουμε αρκετούς στον κατάλογο που θέλουν να πάρουν το λόγο. Αυτή τη φορά, όχι όπως το πρωί, θα κάνουμε ένα γύρο ερωτήσεων από τους συντονιστές πρώτα απ' όλα. Έχουμε τα ονόματα. Θα δώσω και τον κύριο Βερμάιερ, έναν εκπρόσωπο κάποια πολιτική ομάδα, Κονφεράτη, και τον καθηγητή Κορία Κάμπος. Θέλει κάποιος άλλος να εγγραφεί στον κατάλογο. Ο κύριο Σβάμπ ξεκινά και η κυρία Γκέπχαρτ. Πώς θα πάμε το χρόνο. Δύο ερωτήσεις μαζί σας ακούσουμε. Και μετά προχωρούμε πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, πρώτα απ' όλα χαιρόμαστε βέβαια που είσαστε εδώ απόψε. Διότι υπό την Πολωνική Προεδρία του Συμβουλίου και για την ημέρα καταναλωτών και ανταγωνισμού στην, στο Πόσναν στην Πολωνία. Συζητήσαμε για την προστασία των καταναλωτών αφενό και τι δράσει που πρέπει να αναλαμβάνονται αφετέρου. Η επιθυμία να προωθηθεί η ενιαία εσωτερική αγορά και στον τομέα της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς είναι η κατεύθυνση για την τυποποίηση και έχουμε καταβάλει προσπάθειες. Εμείς έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ομάδα εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce ο συνάδελφος που εργάζεται σε αυτή την ομάδα με παρακάλεσε θερμά να ζητήσω μια τοποθέτηση για το payment services, για τις υπηρεσίες πληρωμών. Το κάνατε ήδη εν μέρη και για το Google. Πώς μέσω του Google μια εταιρεία μπορεί να έχει πριτανεύοντα ρόλο, σε αυτό, δεσπόζοντα ρόλο σε αυτή την αγορά. Η ερώτησή μου όμως στρέφεται περισσότερο στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δημόσιων συμβάσεων αφενός και των αδειών καθώς επίσης και των νομικών διατάξεων και ρυθμίσεων αφετέρου. Γι' αυτό ερώτησή μου, στην εκπόνηση των νέων ρυθμίσεων για τις δημόσιες τέτοιες συμβάσεις, ε, κατά πόσον δεσμευθήκατε σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Πιστεύετε ότι οι επιδοτήσεις είναι νόμιμες και συνάδουν με τις νομικές διατάξεις. Κατά πόσον οι προτάσεις σας για τις άδειες, για την αδειοδότηση εξετάζονται υπό αυτό το σκηνικό ή σε σχέση με αυτές ε, έχετε και κάποιους, ε, ας το πω έτσι, κρυμμένους, ε, ε, κρυμμένα δεδομένα υποκρυπτόμενα δεδομένα για την, τις επιδοτήσεις που πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη αυστηρά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, ευχαριστώ πολύ. Θα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τις τοποθετήσεις σας που ήταν ενδιαφέρουσες και σίγουρα με ιδιαίτερη αξία θέσατε στο ότι τα εμπόδια, τα προσκόμματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είπατε ότι εντείνονται περισσότερο και αυτά είναι, είναι παλαιά αντανακλαστικά της ε, εθνικοποίησης. Σημερίζομαι αυτή την άποψή σας και πρέπει από κοινού να δράσουμε εναντίον μιας τέτοιας τάσης εθνικοποίησης και προστατευτισμού. Ένα πράγμα όμως δεν το θέσατε στο προσκήνιο όπως θα ήθελα εγώ να τεθεί στο επίκεντρο τα προσκόμματα, τα αντανακλαστικά που έχουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, τα σύνορα, οι διαχωριστικές γραμμές σε σχέση με τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούνται πάντα προς όφελός τους. Για το τέλος περιαγωγής, roaming, γιατί να υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν τόσες πολλές επιχειρήσεις που δρούν στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά δεν είναι πάντα προς όφελος όλα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά είναι ερωτήσεις που πρέπει να τα να, πρέπει να θέσουμε εναντί των επιχειρήσεων και όχι μόνο εναντί των κρατών. Και αυτό είναι κάτι που κάπως αγνοήθηκε στην παρέμβασή σας σήμερα, στις τοποθετήσεις σας. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι, στην αρχή των όσων μας εκθέσατε, κάνατε λόγο για την κατάσταση των πολιτών στην Ευρώπη, την ανεργία κυρίως την θέση των νέων όσον αφορά την ανεργία, την κατάσταση των νέων. Είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια υψηλά ποσοστά ανεργίας και τάσεις έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα εμπόδια ακόμα σήμερα. Εμπόδια, προσκόμματα, εναντίον μιας οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας, εγκάρσιας κοινωνικής ρήτρας ώστε οι νομοθετικές επιπτώσεις να μπορούν να, να δρουν άμεσα στο πεδίο της εργασίας ε, των ανθρώπων, της ποιότητας εργασίας τους, όπως ε, και οι οικονομικές ε, προϋποθέσεις και όροι αφορούν τις επιχειρήσεις. Με μια τέτοια εγκάρσια προσπάθεια θα είχαμε πολλά να κάνουμε και βλέπω να απουσιάζουν πολλά στοιχεία εδώ. Τρίτο και τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω, έχω όμως άλλα πολλά τα οποία δεν μπορώ όλα να τα καλύψω, αναφέρατε τις ευρεσιτεχνίες. Και είπατε σωστά ότι στον ψηφιακό τομέα το δικαίωμα, το δίκαιο ευρεσιτεχνιών μπορεί να οδηγήσει σε μονοπωλιακές καταστάσεις που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικέ τι γίνεται στον τομέα των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο αυτό. Έχω την εντύπωση ότι όλο και περισσότερο, όλο και πιο έντονα, μέσω του δικαίου για τις ευρεσιτεχνίες και μέσω της παρέμβασης στους πόρους της φύσης, περιορίζεται συνέχεια το πεδίο δράσης. Εσείς ως αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να κάνετε κάτι. Τι σκέπτεστε να κάνετε και για το δίκαιο για τις ευρεσιτεχνίες. Και αυτό είναι ένα θέμα για την καινοτομία ή μη καινοτόμο δράση που θα μπορούσε να επιτύχει κανείς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Επίτροπε, θέλετε να απαντήσετε στις δύο πρώτες αυτές ε, ομάδες ερωτήσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς προς τον κύριο Σβάμπα απευθυνόμενος για το σύστημα πληρωμών είπα κάποια πράγματα στην παρουσίασή μου το επεξεργαζόμαστε το ζήτημα αυτό. Ε, διενεργούνται έρευνες για τις φυτοτικές και τις χρηστικές κάρτες. Ε, είμαστε σε επαφή με εναλλακτικά συστήματα πληρωμών. Προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο υπάρχουν κάποιοι φραγμοί, κάποια εμπόδια για τους ερχόμενους σε αυτή την αγορά. Προσπαθούμε να βρούμε μέσω των μέσων μας για ανταγωνιστική πολιτική να αποφύγουμε τους φραγμούς για τις πληρωμές online. Συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους Μπαρνιέ και Ντάλι και προετοιμάζουμε την πράσινη βίβλο και, την, και ξεκίνησε και δημόσια διαβούλευση πρόσφατα. Και είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Τέλος, όπως είπα, ξεκίνησε μία έρευνα σχετικά με το έργο που έκανε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών που είναι ένας φορέας που είναι στο τραπεζικό πλαίσιο που προσπαθεί να δημιουργήσει ένα σύστημα που κατά την άποψή μας αυτό το σύστημα θα δημιουργήσει ίσως ε, νέους ε, φραγμούς για συστήματα πληρωμών εκτός τραπεζών και το ερευνούμε. Είναι σημαντικότατο το θέμα είναι ένα από τα στοιχεία που θα πρέπει να βελτιωθεί για να ολοκληρωθεί η αγορά. Και στην αναλογική μορφή της ενιαίας αγοράς και στην ψηφιακή μορφή της. Το δεύτερο ερώτημά σας, Google. με έρευνα, το γνωρίζετε πολύ καλά. Το συζητήσαμε και παλαιότερα στην άλλη επιτροπή. Το Νοέμβριο του 2010 ξεκίνησε η έρευνα. Λάβαμε καταγγελίες Λάβαμε υπόψη πληροφορίε εκείνων που έκαναν τις καταγγελίες, λάβαμε υπόψη τι απαντήσεις της Google, κάνουμε τη δική μας έρευνα, μαζεύουμε πληροφορίε. Η αρμόδια ομάδα και η, αρμόδια γενική διεύθυνση τέλος Μαρτίου θα με υποβάλουν έκθεση αρχές Απριλίου. Προς το τέλος του επόμενου μήνα θα μου δώσουν μια έκθεση. Και θα αποφασίσω ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Θα αποφασίσω αν προχωρούν αρκετά καλά οι έρευνες, αν έχουν προχωρήσει αρκετά, τόσο ώστε εμείς να προβάλλουμε σαφώς αντιρρήσεις. Εξακολουθούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες ή καταγγελίες και ανεπίσημες καταγγελίες. Δεν είναι εύκολη δουλειά να ερευνήσουμε το Google το Google ταυτόχρονα δεν έχει σταματήσει τις δραστηριότητές του και αλλάζει το Google. Νομίζω ότι μπορούμε να συναγάγουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα και αν χρειαστεί να στείλουμε μια δήλωση με τις αντιρρήσεις μας στους επόμενους μήνες. Ε, δεν προδικάζω κάποιο επόμενο βήμα αλλά πιθανότατα σε ένα, ενάμιση μήνα θα έχω πιο ξεκαθαρή εικόνα για την κατάσταση. Η δουλειά που έγινε ήταν πάρα πολύ σοβαρή, τεράστιο έργο. Όσον αφορά την κρατική βοήθεια, κρατικές ενισχύσεις, ε, δεν είχα το χρόνο να σας παρουσιάσω αυτό, παρουσίασα στο βήμα περί ανταγωνισμού στις Βρυξέλλες. Ετοιμάζω μία αναθεώρηση του καθεστώτος για τις κρατικές ενισχύσεις. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται για πολλούς λόγους. Ουσιαστικά στόχος της αναθεώρησης εν ολίγης είναι ο εξής. Οι κρατικέ ενισχύσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο βαθμό του δυνατού σαν ένα μέσο για την προώθηση της ανάπτυξης, την ενθάρρυνση δραστηριοτήτων που έχουν στόχο την ανάπτυξη, που είναι φιλικές προς την ανάπτυξη, για την προστασία της ενιαίας αγοράς, για τη χρήση των δημοσίων χρημάτων του το τρόπο ούτω ώστε δεν δημιουργούνται φραγμοί για την ενιαία αγορά, αντιθέτως ε, έρονται τα εμπόδια. Ταυτόχρονα πρέπει να χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι για την πρόθεση της ανάπτυξη ε, με ευφυή τρόπο. Και ευφυή τρόπο εννοεί τώρα με έναν τρόπο που να μην δημιουργεί και άλλα προβλήματα στα δημοσιονομικά. Από την άλλη πλευρά, να μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη της κυβερνήσης να κάνουν οικονομίες ή τουλάχιστον να μην σπαταλούν δημόσια χρήματα από τα κράτη-μέλη εξαρτάται το πώς θα δαπανίσουν τα χρήματα του εθνικού προϋπολογισμού. Θα πρέπει η χρήση των δημοσίων χρημάτων να τεθεί υπό έλεγχο και με τη χρήση αυτών των μέσων ελέγχου μπορούμε να τους βοηθήσουμε να εστιάζονται καλύτερα στις προτεραιότητές τους και στον προσανατολισμό τους τα κράτη και να αποφύγουν τη δημιουργία εσωτερικών φράγμων και να αποφευθεί σπατάλη χρήματος. Ε, αυτή είναι η γενική στόχη. Πώς θα το πετύχουμε. Ξεκινούμε την αναθεώρηση και την ενημέρωση πολλών προσανατολισμών, πολλών κατευθυντήριων γραμμών. Έχουμε 37 διαφορετικές ε, κατευθυντήριες γραμμές και χρειάζεται ενημέρωσή τους, εξυγχρονισμός τους. Και αυτό πρέπει να γίνει με ένα συνεκτικό τρόπο, βάσει των γενικών στόχων βάσει των γενικών προτεραιοτήτων. Ταυτόχρονα πρέπει να απλουστεύσουμε στο μέτρο του δυνατού τις διαδικασίες μας, χωρίς να χάσουμε την ποιότητα των ερευνών μας. Έχουμε μακροσκελείς διαδικασίες όμως και είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε την ίδια προσοχή σε μια και στις μικρότερες υποθέσεις όπως και στις μεγαλύτερες. Αυτό δεν ισχύει στις συγχωνεύσεις που έχουμε απλουστευμένη διαδικασία για μικρές συγχωνεύσεις. σε συγχωνεύσεις που δεν έχουν διαστάσεις που απαιτείται για να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην εσωτερική αγορά. Στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων πρέπει να διαρευνήσουμε πώς μπορούμε να κινηθούμε προς απλούστερο τρόπο αντιμετωπίσεως των απλών υποθέσεων. Ίσως και να αλλάξουμε και το κατώτατο όριο, το και τον κανονισμό και τα επίπεδα για τις ε, ομαδικές εξαιρέσεις και το σχετικό κανονισμό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι λόγω τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρέπει να εξετάσουμε τι καταγγελίε. Οι μισέ υποθέσει που ξεκινούν για τι κρατικές ενισχύσει δεν είναι από κοινοποιήσει ούτε από αυτεπάγγελτε έρευνε, αλλά από καταγγελίε. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις νομικές δυνατότητες που έχουμε και τα νομικά μέσα και την νομολογία και τα κριτήρια της νομολογίας για να οργανώσουμε καλύτερα τις εργασίες μας, να εστιαστούμε επί των μεγάλων υποθέσεων. Όπως κάναμε πρόσφατα με τις κοινοφελείς οικονομικές υπηρεσίες και να προσπαθήσουμε στο μέτρο του δυνατού να απλωστεύσουμε τις διαδικασίες για τις μικρές υποθέσεις. Πώς σχετίζεται αυτό με τις δημόσιες προμήθειες και τα διάφορα καθεστώτα εκχωρήσεων είναι προφανές. Έχουμε υθετήσει ένα πακέτο πέρσι σχετικό και προσπαθήσαμε να ευθυγραμμίσουμε στο βαθμό του δυνατού τη διαδικασία ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων με του κανόνε για τι δημόσιε προμήθειε. Οι κανόνες για τι δημόσιε προμήθειε άλλαξαν. Ο συνάδελφό μου Μισελ Μπαρνιέ υπέβαλε σχετικές προτάσεις για αλλαγέ στι δημόσιε προμήθειε, Θα συζητηθούν και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Και προσπαθούμε να ευθυγραμμιστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τι δικέ μα διαδικασίε με τι διαδικασίε για δημόσιε προμήθειες. Αυτό δεν είναι πάντα δυνατόν. Σε κάποιε περιπτώσει. δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία και δεν μπορούμε να υποθέσουμε το ότι ένα δημόσιο διαγωνισμό έλαβε χώρα δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση. Μπορούμε όμω να απλουστεύσουμε τι διαδικασίε και να τι συντονίσουμε καλύτερα. Προ την κυρία Γκέπχαρτ η απάντησή μου. Η φραγμή και τα εμπόδια στην ψηφιακή εσωτερική αγορά είναι πάρα πολύ υψηλή και υψηλά. Γιατί λόγω ρυθμιστικών φραγμών σε κάποιες περιπτώσεις από εσά εξαρτάται να αρθούν βάσει δικής μας πρωτοβουλίας αλλά η πολιτική ανταγωνισμού δεν αφορά τον κανονισμό. Αν υπάρχουν κανόνες, νόμοι που δημιουργούν φραγμούς ή συντηρούν τους φραγμούς, από εσά εξαρτάται όλα αυτά να τα βγάλετε. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να παρέμβουμε και παρεμβαίνουμε. Πιστεύω ένθερμα στον καλό συνδυασμό ρυθμίσεως και κανόνων και αποφάσεων με βάση τον ανταγωνισμό, ρυθμιστικών διαδικασιών και επιβολής του ανταγωνισμού. Χρειάζονται και οι δύο πτυχές. Χρειάζονται τα δύο φτερά για να πετάξει το αεροπλάνο του ΣΥΠΗΝ. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα προβλήματα μέσω των μέσων για την ανταγωνιστική πολιτική. Σε, στην κινητή τηλεφωνία, στην αγορά κινητή τηλεφωνία δεν μπορούμε να τα τα προβλήματα μόνο με μέσα ανταγωνισμού. Και η Νέλη Κρούς δεν πάνε όλα τα προβλήματα μέσω των κανονισμών που σας στέλνει σε εσά και στο Συμβούλιο. Χρειάζεται συνεργασία και συνεργαζόμαστε πράγματι στο μέτρο του δυνατού πάντα. Πνευματικά δικαιώματα, μεγάλος φραγμός και δύσκολο θέμα. Πνευματικά δικαιώματα, copyright, ε, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Χρειάζεται καινοτομία, χρειαζόμαστε νέες ιδέες δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων την ψηφιακή εποχή με τον ίδιο τρόπο που τα αντιμετωπίζαμε το θέμα αυτό στην αναλογική εποχή. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να διατηρήσουμε τα ίδια μέσα για την προστασία των δικαιωμάτων των εκείνων που παραγματοποιούν καινοτομίε και των δημιουργών και τα συναφή δικαιώματα των δημιουργών. Σε άλλες περιπτώσεις όμως πρέπει να βρούμε νέους τρόπους για να πετύχουμε τον ίδιο στόχο. Το διαδίκτυο άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού και πρέπει να αντιδράσουμε στις αλλαγές αυτές. Η κοινωνική ρήτρα είμαι υπέρ. Γνωρίζω ότι εδώ σε αυτή την αίθουσα στους συναδέλφους των διαφόρων πολιτικών ομάδων και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο υπάρχουν διαφορετικές ιδέες που επικρατούν. Εγώ είμαι υπέρ και περιμένω πώς και πώς να σχηματιστεί μια πλειοψηφία όσον αφορά αυτό το θέμα. Τώρα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείται με την προστασία για βιοτεχνολογικές εφευρέσεις, αν περί αυτού επρόκειτο. Αν κατάλαβα σωστά, αν έπιασα σωστά το ερώτημα. Στον τομέα της πληροφορικής Έχουμε κάποια τυποποιημένα είδη διπλωμάτων ευρεσιτεχνία και είναι προφανέ ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο καταχρήσεων θέσεων στην αγορά από εκείνους που κατέχουν τα δικαιώματα, που χρησιμοποιούν αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνία για να αποκλείσουν του ανταγωνιστέ. από τη στιγμή που σε κάποιε προδιαγραφέ συμπεριληφθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται επίσημα σε κάποιο πρότυπο, ε, ένα δίπλωμα ευαισθητεχνία χρειάζεται για διεπαφή, για τη λειτουργία συσκευών ή για το λογισμικό των ανταγωνιστών και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό και το κάνουμε. Αντιμετωπίζουμε τα θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίων στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας. Υιοθετήθηκαν μετά το 2009. Παρακολουθούμε διάφορες υποθέσεις κατά το trust που βλέπουν ότι χρησιμοποιούν από του αρχικού χρήστες ε, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, και έναντι των εταιριών γενοσύμων φαρμάκων υπήρχε και συγκεκριμένη υπόθεση συμπεριφοράς μεταξύ εταιριών παραγωγής γενοσύμων φαρμάκων που χρησιμοποιούσαν με λάθο τρόπο, αν θέλετε, ε, τα διπλώματα τεχνία. Αυτό το μέσο δίνει δύναμη στην αγορά και πρέπει να παρακολουθούμε από πολύ κοντά το ποιε δυνατότητε δίδονται και πώ χρησιμοποιούνται. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσέξουμε να μην σκοτώσουμε τα κίνητρα για την καινοτομία. Διότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνία είναι πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο για τον καινοτόμο, για τον δημιουργό. Ταυτόχρονα, όπως με κάθε δικαίωμα, υπάρχουν και όρια. Διότι μπορεί να υπάρξει και δυνατότητα κατάχρησης του δικαιώματος του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τα αποτελέσματα να είναι πολύ αρνητικά για πολλούς άλλους. Καλώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα σημεία που θίξατε. Έχουμε ακόμη ένα τέταρτο στη διάθεσή μας. Έξι ακόμη ομιλητέ έχω, εκτός αν θέλει κάποιος άλλος ε, να εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ένας από κάθε πολιτική ομάδα και ο κύριος Μπαλτεσάρε θέλει να πάρει το λόγο. Ρούλε, Κόζινσης και Μάιερ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ένα ερώτημα ο καθένας θα ήταν το καλύτερο. Και μετά θα λάβουν το λόγο οι υπόλοιποι ομιλητές. Κύριε Αρούλε. Πολλά τα προανέφεραν οι προαλαλήσαντες και έτσι θα είμαι σύντομη. Κυρίως ένα σημείο θέλω να τονίσω. Το σύστημα, <clears throat> διαδικτυακό σύστημα πληρωμών, Internet Payment System. Payment system. Εδώ πρέπει να μεριμνήσουμε να μην υπάρξει στρέβλωση στην αγορά. Σημαντικό είναι στις διαδικτυακές πληρωμές να υπάρχει εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη. Αυτό κάπως αγνοήθηκε από εσάς. Το σύστημα πληρωμών χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Win-win ε, κατάσταση προς αμοιβαίο όφελος. Αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους πολίτες. Έχουν την εντύπωση ότι δεν υπάρχει αρκετή ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η ουσιαστική μου ερώτηση όμως αφορούσε το θέμα των κρατικών δημόσιων επιδοτήσεων. Σωστό είναι αυτό που λέτε, ότι κυρίως οι μικρές επιδοτήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν διαφορετικά από ότι οι μεγάλε κρατικέ επιδοτήσει και ε, αναφέρατε την έκθεση του κυρίου Μάριο Μόντι στην αρχή. Ο Μάριο Μόντι, όπως και με πολλές άλλες μελέτες, αναφέρει ότι στον τομέα των επιδοτήσεων, κρατικών επιδοτήσεων και στον τομέα των συμβάσεων υπάρχει υπερβολικό γραφειοκρατικό βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δυσχεραίνει ιδιαίτερα τα πράγματα και κατεπηγόντως πρέπει να πλουστευθεί, να ανακουφιστεί. Ερώτησή μου, μπορείτε να περιγράψετε επακριβέστερα με περισσότερες λεπτομέρειες πώς τοποθετήσετε στο θέμα της απλούστευσης των μικρών επιδοτήσεων, μικρών κρατικών επιδοτήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοζίτνικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα χρησιμοποιήσω την ισπανική γλώσσα για να μην χαθούμε με τις μεταφράσεις. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα έλεγα υπό ένα πρίσμα, υπό την άποψη της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών, το τρίγωνο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει τέλεια τα πράγματα και εμείς μπορούμε να χειροκροτήσουμε, να επικροτήσουμε τις προσπάθειες αυτές από διαφορετικές κοινοβουλευτικέ ομάδες. Εκείνο το οποίο με ανησυχεί κάπως στα όσα είπατε είναι μια σύντομη περιγραφή, κάπως υποκριμένη θα έλεγα, την αναζήτηση πόρων που είπατε, αναζήτηση δυνατοτήτων και πόρων. Θα ήθελα υπό αυτό το πρίσμα, υπό τη δική μου κοινοβουλευτική ομάδα να πω, θα ήθελα να γνωρίζω αν υπάρχει κάποια εγγύηση, κάποια εχέγγυα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ υπό το δικό σας αξίωμα της, ε, του Αντιπροέδρου ότι δεν θα υπάρξει νέα νομοθεσία με νέα επιβολή νέων φόρων για την δημιουργία αυτού του πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για τα εξαιρετικά σας ισπανικά. Κύριε Σοβερμάιερ. Ο κύριος Σοβερμάιερ. Ευχαριστώ πρόεδρε στρέφομαι προς τον Αντιπρόεδρο αμέσως για το θέμα του δικαίου καταπολέμησης των μονοπωλίων. Ανακοίνωσε το έτος αυτό ότι θα υπάρξει προσφυγή για την παραβίαση του δικαίου για τον ανταγωνισμό και θα δημιουργηθεί αυτή η δυνατότητα. Αυτό θα είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τι γίνεται σε σχέση με τέτοιες προσφυγές από ιδιώτες πότε θα μπορούν να, να έχουν πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία μέσα στο πλαίσιο του προγραμματός σας. Και αυτό θα είναι σημαντικό ώστε να ε, μην υπάρξει νομική αβεβαιότητα και νομική ανασφάλεια στην Ευρώπη. Και είναι εδώ θέμα το οποίο πρέπει να συνεισφέρει σε αποσαφήνιση των πραγμάτων. Θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η βάση όσον αφορά την ποιότητα των προγραμμάτων αυτών. Κανένας εθελοντικά δεν θα είναι πρόθυμος να τοποθετηθεί από αυτόν και να δώσει στοιχεία για τις προσφυγές για αποζημίωση. Χωρίς μια ρύθμιση ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα υπάρξει κατάτμιση, κατακαιρματισμό στο νομικό πλαίσιο της Ευρώπης και αυτό είναι το αρνητικό το οποίο δεν πρέπει να υπάρξει. Να γυρίσουμε στα εθνικά δικαστήρια τα οποία θα αποφασίζουν αν θα διασφαλίζεται πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα σε κάποιους που έχουν ασκήσει προσφυγές ή όχι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην κατάσταση που διαμορφώνεται όταν έχει κάποιο απέτηση για αποζημίωση να μην κάνει ε, το shopping, να μην επιλέγει την χώρα εκείνη στην οποία θα υπάρχει η πιο ευνοϊκή για εκείνον κατάσταση όσον αφορά τι αποζημιώσει. Ελπίζω θα βρεθεί καλύτερη λύση από εσά. Αλλά ερώτηση. Μπορούμε να γνωρίζουμε κάτι από τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χρονοδιάγραμμα. Τι γίνεται σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και προς ποια κατεύθυνση θα κινηθείτε. Αφενός ε, όσον αφορά το ε, δίκαιο, το δημόσιο δίκαιο ή και το ιδιωτικό δίκαιο για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές και η Επίτροπη το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε παρότι ρώτησε στα ε, Ισπανικά και εγώ θα ήθελα εδώ λοιπόν να επιλέξω να απαντήσω και στην ε, δική μου γλώσσα στα Ισπανικά. Το σύστημα πληρωμών, η εμπιστοσύνη που αναφέρθηκε για τους χρήστες, αυτό το σύστημα χωρίς αμφιβολία είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. <clears throat> Δεν βρίσκεται άμεσα συνδεδεμένο με τον ανταγωνισμό, με την πολιτική ανταγωνισμού, όμως έχει τεράστια σημασία. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό με κανένα τρόπο. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Κάθε φορά που κάνουμε μια πληρωμή στο διαδίκτυο με την πιστοτική κάρτα ηλεκτρονικά έχουμε πάντα αμφιβολία αν μήπως κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει καταχρηστικά τα στοιχεία μας αυτής της κάρτας μας. Εγώ μέχρι σήμερα δεν είχα καμιά αρνητική εμπειρία, κανένα αρνητικό βίωμα. Μου αφαιρούσαν από το, ε, την κάρτα μου ε, αυτά τα οποία έπρεπε να παρακρατήσουν και δεν χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία μου για κανέναν άλλο ε, αρνητικό σκοπό. Λοιπόν, έχω αποκτήσει και, έχω εμπιστοσύνη σε αυτά τα συστήματα. Αν κάτι μπορώ να κάνω περισσότερο και δεν είμαι πραγματο... ειδικό, θα έπρεπε να γίνει. Διότι είναι χωρί αμφιβολία η πληρωμή του μέλλοντο, η ηλεκτρονική πληρωμή. Όλο και λιγότερο χατονομίσματα θα χρησιμοποιούμε και κέρματα όλο και λιγότερο θα χρησιμοποιούνται τα χρήματα και όλο περισσότερο το κλικ ηλεκτρονικά. Θα αυξάνεται και η κατανάλωση έτσι ε, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Για τις κρατικές επιδοτήσεις, μικρές κρατικές επιδοτήσεις, τι μπορεί να γίνει. Όπως προανέφερα, δεν μπορούμε να απορρίψουμε τα, τις προσφυγές και τα παράπονα. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκρινόμαστε και να απαντούμε σε όλα τα παράπονα και προσφυγές για κρατικές επιδοτήσεις όταν μας υποβάλλονται. Όμως ε, αρχίζουμε την εργασία σε αυτό και έχουμε την πρόθεση να πλουστεύσουμε στο μέγιστο τις ε, διεργασίες ανάλυσης, την ανάλυση αυτών των μικρών κρατικών επιδοτήσεων. Υπάρχουν μέτρα που έχουν υιοθετηθεί στο παρελθόν κιόλα. Υπάρχει ένας κανόνας κατελάχιστον, de minimis, που θεσπίζει ένα επίπεδο κάτω από το οποίο ένα ποσό κάτω από το οποίο θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πλέον επιδότηση. Και στην μεταρρύθμιση των κρατικών επιδοτήσεων θα θέλαμε να αυξήσουμε αυτό το επίπεδο de minimis, το κατελάχιστο. Θα δούμε μέχρι ποιο επίπεδο θα φτάσουμε και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Υπάρχει μια εξαίρεση ανακατηγορία γενικά που οδηγεί στην δυνατότητα του να μην προειδοποιείται, να μην υποβάλλονται γνωστοποιήσεις για τέτοιες επιδοτήσεις, παρότι μπορεί να πρόκειται για επιδοτήσεις υπό την έννοια της συνθήκης επιχορηγήσεις. Σήμερα το 80% των κρατικών επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων που γνωρίζουμε και καταχωρούμε, καταγράφουμε, <clears throat> γίνονται μέσω εθνικών προγραμμάτων έτσι δεν, τις, ε, δεν τα αναλύουμε αυτά ατομικά επιμέρους, αλλά αναλύουμε τι γίνεται σε σχέση με ένα εθνικό πρόγραμμα. Έχουμε προχωρήσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να υπάρχει και ανταπόκριση, να προχωράμε και να υπάρχει και περαιτέρω πρόοδος, να ελέγχεται ο έλεγχος εκ των υστέρων, εξ για το πόσο καταβάλλονται τέτοιες εθνικές επιδοτήσεις μέσα στα εθνικά προγράμματα. Με αυτά όλα τα στοιχεία, με αυτές όλες τις μορφές, με βάση αυτές τις αρχές, μπορούμε να πλουστεύσουμε να απλοποιήσουμε περισσότερο το σύστημα των επιδοτήσεων και πρέπει, χρειαζόμαστε να γίνει αυτή η απλούστευση. Αληθεύει ότι καμιά φορά η διάρκεια όσον αφορά αυτή την ε, ενέργεια εξέτασης κάποιων συγκεκριμένων επιδοτήσεων είναι χρονοβόρα διαδικασία. Το κράτος μέλος ε, αντίστοιχα σε σχέση με τις ε, υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης για τον Ανταγωνισμό στρέφεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει καθυστερείτε πολύ και Πρέπει να σας πω ότι σήμερα το πρωί είχα δύο τέτοιες υποθέσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσω εναντί εκπροσώπων δύο κρατών μελών. Είπα δεν είμαστε εμείς εκείνοι που καθυστερούμε. Είσαστε εσείς εκείνοι που καθυστερείτε να μας υποβάλλετε τα στοιχεία εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε για να λάβουμε αποφάσεις, πληροφοριακά στοιχεία για ενημέρωση για τις αποφάσεις μας. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις ίδιες προθεσμίες νόμιμα όπως για παράδειγμα υφίστανται στο σύστημα ε, συγχωνεύσεων και ενώσεων. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην κατάσταση σεβασμού, ε, να σέβονται όλοι αυτές τις προθεσμίες όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Νέοι ναι, ευρωπαϊκοί φόροι τώρα. Στο θέμα του ανταγωνισμού δεν έχουμε καμιά αρμοδιότητα να επιβληθούν κάποιοι φόροι. Έχουμε πολλέ ευθύνε όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευρά μα, αλλά δεν μπορώ να εγκρίνω εγώ φόρου ή να του απορρίψω. Να είσαστε ήσυχοι λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να επιστρέφονται τα αχρεωστήτω καταβληθέντα ή σε σχέση με ε, το δημόσιο από το 2010, πέρα από την ε, ανάκτηση τέτοιων ε, ποσών στι επιδοτήσει, τα πρόστιμα για την παραβίαση όσον αφορά αφορά την κατάσταση ολιγοπολίων και καρτέλ ήταν πάνω από 3 δις. Το επόμενο έτος είχαμε μικρότερες, μικρότερο τέτοιο όγκο. Είχαμε και λιγότερες τέτοιες ε, περιπτώσεις. Οι αποφάσεις που ελάβαμε δεν ε, ανήρχονται σε τέτοιο υψηλό ποσό. Δεν μπορώ να θυμηθώ τα ποσά του 2012, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις στο τέλος, τέλος ε, το συμπέρασμα όσον αφορά τις αποφάσεις για την επιβολή προστίμου ή όχι είχαμε κάποιες, κάποιους, κάποια τέτοια πρόστιμα που δεν είναι ε, τόσο υψηλά αλλά που θα βοηθήσουν να, να ανακουφιστούν τα δημοσιονομικά κάποιων κρατών μελών. Και όσον αφορά τις, τα, τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως εισπράττονται από τα κράτη-μέλη στο τέλος τέλος. Και σε σχέση με το να ε, δηλώνονται ε, ασύμβατα όσον αφορά τα κράτη τέτοιου είδους ε, δράσεις, επιστρέφονται αυτά τα ποσά. Έτσι λοιπόν δεν εργαζόμαστε, ας το πω έτσι, προς όφελος ατομικό εμείς οι ίδιοι, αλλά έχουμε ο όφελος υπέρ των δημοσιονομικών των κρατών μελών στα οποία επιστρέφουν αυτά τα ποσά. Όσον αφορά αυτό, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει κανόνες για την πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα που θεωρούμε ότι είναι αρκετά πιο ανοιχτοί αυτοί οι κανόνες και αρκετά πιο γενναιόδοροι αυτοί οι κανόνες από ό,τι σε σχέση με άλλα θεσμικά όργανα ή σε σχέση με κράτη-μέλη. Ε, και για την δυνατότητα αναφοράς ε, για να υπάρξει τέτοια τεκμηρίωση σε σχέση με τη συμμόρφωση προς αυτά τα στοιχεία είμαστε υποχρεωμένοι εμείς οι ίδιοι να δίνουμε πολλές περισσότερες πληροφορίες σε ένα Εθνικό Κοινοβούλιο από ότι για παράδειγμα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή άλλα θεσμικά όργανα που έχουν και εκείνα στην κατοχή τους τέτοια στοιχεία που αναφέρονται σε αναφορές που καταλήγουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνειδητοποίηση των ορίων, των ορίων που υπάρχουν και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για οποιοδήποτε και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο <clears throat> και για τα εθνικά κοινοβούλια για τέτοιου είδους στοιχεία που έχουμε εμείς ε, στην κατοχή μας. Αν ξεπεράσουμε κάποια συγκεκριμένα όρια μπορεί να παραβιάσουμε το θέμα της προστασίας απορρίτων, business secrets, δηλαδή να αποκαλύψουμε απόρριτα επαγγελματικά ή επιχειρηματικά και να προσέξουμε την αναγκαία εκείνη συνεργασία ώστε οι έρευνές μας να μπορέσουν να προχωρήσουν για την καταπολέμηση των ολιγοπολίων χωρίς να αποκαλύπτονται στοιχεία όπως δεν θα έπρεπε. Έχουμε κάποια όρια λοιπόν και μέσα σε αυτά τα όρια πάντα είμαστε υπέρ πάντα της διαφάνειας ώστε να, έχουν, να μπορούν να έχουν πρόσβαση ε, πολίτες σε τέτοιου είδους ε, έγγραφα. Δεν είναι έγγραφα ή στοιχεία δικά μας, τα έχουμε εμείς στην κατοχή μας, αλλά σε αυτό αναφέρεται, σε αυτό το πλαίσιο αναφέρονται. Για το τελευταίο σας σχόλιο, σε κάποιους τομείς υπάρχουν πρόοδοι που σημειώνονται προς μια μεγαλύτερη σύγκληση όσον αφορά τα δικαστικά συστήματα, τα δικονομικά συστήματα των κρατών μελών, αποφεύγοντας το μέτρο του εφικτού το proper shopping, την επιλογή δηλαδή προς ε, ατομικό ευνοϊκότερη αντιμετώπιση κάποιου. Σε σχέση τώρα παραβίασης κάποιων διατάξεων για τον ανταγωνισμό και σε σχέση και με την εμπλοκή εθνικών αρχών για την καταπολέμηση του, ε, των περιπτώσεων αυτών παραβίασης του ανταγωνισμού λειτουργούν τα πράγματα καλά και έχουμε και σε σχέση με την ειδοποίηση για μια συγχώνευση δυνατότητες και σε σχέση με, μια εθνική, με τις εθνικές αρχές και έτσι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζεται η παράκαμψη των κανονισμών. Έτσι λοιπόν, μπορούμε και λειτουργούμε σωστά. Αν εσείς όμως αναφέρεστε στο συσχετισμό μεταξύ του δημόσιου ε, ε, χαρακτήρα ε, σε σχέση με μια τέτοια αρμοδιότητα, αρμοδιότητα δική μας έναντι των εθνικών αρχών για το δημόσιο ιδιωτικό χαρακτήρα αντιστάθμιση και αποζημίωση ζημιών εκείνων που υπήρξαν θύματα ε, περιπτώσεων παραβίασης του δικαίου για τον ανταγωνισμό. Για τέτοια πράγματα πρέπει εμείς να παρεμβαίνουμε νομοθετικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό τον ίδιο μήνα υιοθέτησε ένα ψήφισμα πολύ σημαντικό για συλλογικές προσφυγές. Υπό αυτό το πρίσμα ο η αρμοδιότητα για, τον ανταγων... για την αποζημίωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ατομικές προσφυγές αλλά και τις συλλογικές προσφυγές. Και αυτό αναγνωρίζεται και στο ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έτσι εκρεμεί και πρέπει να ρυθμιστεί πώς θα διαμορφωθεί στην, πρακτική, ε, στην χειροπιαστή πρακτική η δέσμευση που είχαμε και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, φέτος. Ότι θα υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα υποβληθεί στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ιδιωτικό αυτό χαρακτήρα, την ιδιωτική ή αυτή η αυτή η συνιστόσα του δικαίου για τον ανταγωνισμό. Αντιστάθμιση για προσφυγέ που θα υποβάλλονται όσον αφορά τέτοιε παραβιάσει του δικαίου του ανταγωνισμού. Uh, um, Αγαπητοί συνάδελφοι, τέσσερα ακόμη ονόματα έχω στον κατάλογο μιλητών. Δέχθηκε ο Επίτροπος να μείνει λίγο ακόμη μαζί μας. Κοφεράτη, Κορίδα Κάγκος, Μπίλα και Βαλτεσάρε. Ένα ερώτημα μπορώ να σας ζητήσω να ε, απευθύνετε. Ένα σύντομο ερώτημα. Γιατί και η κυρία Κόμη είναι εδώ να μας παρουσιάζει το δικό της θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ανέφερε και ο Επίτροπος. Κύριε Κοφεράτη, ένα ερώτημα. Το ίδιο ισχύει για τους υπολείπους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση Ευθεία, κατά μέτωπο, δεν ξέρω αν επιτρέπετε. Ανευχάριστη μάλλον. Ξεκινήσατε επενθυμίζοντάς μας την οικονομική κατάσταση, την χείριστη των ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων ε, ε πολλές από αυτέ είναι σε ύφεση. Και υπενθυμίσατε και κάτι άλλο. Ε, του, του Πρωθυπουργού μου, του κυρίου Μόντι, όσον αφορά την ανάγκη να υπάρχει μια νέα αγορά ισχυρότερη από αυτή που υπάρχει σήμερα. και ότι δεν προσέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες το θέμα αυτό. Υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών. Έχω την εντύπωση ότι όταν οι οικονομίες πάνε άσχημα, ο όλα στη δουλειά μας γίνονται δύσκολα, λόγω διότι οι ενώσεις, τα μονοπόλια ε, προβάλλουν μεγαλύτερες αντιστάσεις. Σε μία περίοδο έλλειψης ανάπτυξης προσπαθούν να προφυλάξουν τα υπάρχοντα. Διερωτώ με μήπως για αυτό το λόγο δεν θα χρειαζόταν μία παραπάνω προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα πριν και μετά σε αυτές τις δραστηριότητε. Και δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να σταματήσει καμία εργασία, αλλά ίσω θα χρειαζόταν έκτακτη προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εντοπίσει πόρου και να δώσει πραγματικό μήνυμα για την ανάπτυξη μέσω παραδοσιακή και νησιανή παραδοσιακή πολιτική. Διαφορετικά και η δική σα και η δική μα ζωή θα είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι θα ήταν λογικό να είναι. There was a Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι αναφερθήκατε στο Collective Redress και το ότι αναφέρατε ότι στην ατζέντα σας έχετε υπόψη να προπαρασκευάσετε νομοθετική πρόταση για την ιδιωτική συνιστόσα του ιδιωτικού δικαίου για τις αποζημιώσεις σε περίπτωση παραβιάσεως του δικαίου για τον ανταγωνισμό. Το θέμα εδώ είναι, θα ήθελα να αναφέρω το θέμα σε σχέση με τα εθνικά συστήματα όπου υπάρχουν επιθεωρήσεις και παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανοχή ακόμα που έχουν τα κράτη και που υπάρχει μεταξύ κρατών είναι τεράστια διότι θεωρούνται στρατηγικό αγαθό, στρατηγικού χαρακτήρα αυτά τα ε, θέματα. Είναι δύσκολο να πείσουμε έναν Ευρωπαίο πολίτη ότι όταν υπάρχει μια ε, τέτοια κατηγορία εις βάρος ε, ε του στις τηλεπικοινωνίες ε, εθνικού παρόχου να πείσουμε ότι πρόκειται για κάτι σωστό και ιδιαίτερα όταν υπάρχει μονοπωλιακός χαρακτήρας ότι πρέπει να υπάρξει άμεση δράση. Αναφέρον στο ευάλωτο, ε, στον ευάλωτο χαρακτήρα των αρχών για τον ανταγωνισμό. Τι σκέπτεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσει τις, ευρωπαϊκές, τις ε, αρχές των κρατών μελών για τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. E, kredytowych według e, Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των πληρωμών και στο θέμα των τελών στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Η Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας ε, ε, γνωστοποίησε μια έκθεση για τέτοιου είδους τέλη. Στη χώρα μας είναι διπλάσια αυτά τα τέλη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές από ό,τι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και οκταπλάσιο κιόλας ε, σε σχέση με τέτοιες συναλλαγές ένα ολόκληρο σημαντικό ε, ποσοστό χρησιμοποιείται ε, όσον αφορά την βίζα και ε, 0,72 σε άλλες χώρες ενώ 1,60 στη δική μου χώρα. Δηλαδή δεν κατανοώ γιατί πρέπει να είναι το διπλάσιο ή πολλαπλάσιο. Και για ιδιοκτήτες ε, επιχειρήσεων αναφέρουν, αναφέρουν ότι αυτά τα υψηλά τέλη αποθαρρύνουν τους πολίτες να χρησιμοποιούν στις πληρωμές τους ε, τις πιστοτικές τους κάρτες ε, ηλεκτρονικά. Αυτό το οποίο αφορά σε σχέση με τα όσα αναφέρατε θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Έχετε υπόψη σας ρυθμιστική δράση μέσα στη δική σας θητεία για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο σε σχέση με τους όσους εκδίδουν αυτές τις πιστοτικές κάρτες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα ήθελα να μας πείτε τι θα κάνετε. Ευχαριστώ. Κύριος Μπαλτασάρη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα Προτάσει σα. Το θέμα τη διαφάνεια, κύριε Επίτροπε, και τη τακτικότητα των δημοσίων διαγωνισμών, κυρίω εκείνων που πραγματοποιούνται με κες, είναι θεμελιώδου σημασία για την εσωτερική αγορά και για τον ανταγωνισμό. Όμω, ακόμα σήμερα, πολλέ επιχειρήσει αντιμετωπίζουν δυσκολίε όσον αφορά τη συμμετοχή του σε δημόσιες ε, στους δημόσιους διαγωνισμούς, κυρίως στις νέες χώρες που προσεχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στη, ας πούμε, ζητούν στους διαγωνισμούς να συμμετέχουν κάποιοι επαγγελματίε οι οποίοι έχουν διαμείνει σε κάποιες χώρες ή να συστήσουν εταιρείες που είναι καταχωρημένες σε κάποια μητρώα ή απαιτήσει ε, που ε, διαγωνισμοί που ακυρώνονται και δεν μπορούν να κάνουν πολλά προβάσει Ευρωπαϊκή Ενώσεω, διότι η αρμοδιότητα είναι του κράτου μέλου. Τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίω τι προτίθεται να κάνει εκεί όπου πολλοί από αυτού του διαγωνισμού στην πραγματικότητα χρηματοδοτούνται από τα χρήματα του στόχου 1, των στόχων τη σύγκληση με χρήματα τη Ευρωπαϊκή ε, Κοινότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια και υπήρξαν δύο παρεμβάσεις ε, στα Ιταλικά και στα Πορτογαλικά, θα μιλήσω Ισπανικά απαντώντας. Η ανάπτυξη. Πού βρίσκεται η ανάπτυξη. Αυτή είναι η ερώτηση. Με κεφαλαία γράμματα. Ελπίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 1 ε, και Δευτέρας Μαρτίου ε, μεθαύριο και την ε, Παρασκευή θα γίνει αυτό από το Συμβούλιο, διότι οι προσαρμογές από πλευράς προϋπολογισμών δημοσιονομικά είναι απόλυτα αναγκαίες συνθήκες και υποχρεωτικά αναγκαίες στις χώρες μας. Αληθεύει ότι ήδη υπό το πρίσμα το δυναμικό για ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομιών ήταν χαμηλό πριν και τώρα κατά τη διάρκεια ή και μετά την κρίση μειώθηκε ακόμα περαιτέρω. Πρέπει να αυξηθούν λοιπόν οι δυνατότητες ανάπτυξης με μεταρρυθμίσεις διαθωτικού χαρακτήρα. Αληθεύει ότι το οικονομικό σύστημα αντιμετωπίζει δυσκολίες, πολύ μεγάλες δυσκολίες. Εν μέρη ως αίτιο με προέλευση την ίδια την κρίση. Εν μέρη όμως σαν συνέπεια μιας δεύτερης ενός δεύτερου πλήγματος της κρίσης που είναι η κρίση του χρέους, των κρατικών χρεών. Και γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη σε ένα οικονομικό σύστημα ή σε εκείνο το οικονομικό σύστημα <clears throat> σε σχέση με την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας ε, τους επόμενους μήνες και ακόμα περισσότερο για την δημιουργία βάσεων και ε, δυνατότητας ε, κεφαλαίου για την συνέχιση της δράσης της μόχλευσης και υπό το πρίσμα της χρηματοδότησης βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολύ περίπλοκη και σύνθετη. Όμως, από την άλλη πλευρά του των λεχθέντων, Χρειαζόμαστε απόλυτα την ανάπτυξη. Χωρίς ανάπτυξη δεν θα μπορέσει να εξηγιανθεί το οικονομικό, δημοσιονομικό οικονομικό σύστημα. Δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κρίση του χρέους. Και οι διαθροτικές ε, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις δεν θα δώσουν τους επιθυμητούς καρπούς. Η απάντηση πιο ορθόδοξη σε όλα αυτά είναι ότι αυτή η ανάπτυξη θα προέλθει από την δημιουργία εμπιστοσύνη. Και αυτό αληθεύει. Όσο μεγαλύτερο κλίμα εμπιστοσύνη υπάρχει μεταξύ των εμπλεκόμενων στον οικονομικό τομέα, επενδυτών, εμπλεκόμενων, τόσο και πιο εύκολο θα είναι να βρεθεί μια λύση για την ανάπτυξη. Αλλά επίση αληθεύει και είναι μια ορθόδοξη, ορθόδοξου χαρακτήρα απάντηση ότι χρειάζεται επίση η εξωτερική, εξωτερική ζήτηση να συνεισφέρει για αυτή την ανάπτυξη. Γύρω από την Ευρώπη υπάρχουν οικονομίες που αναπτύσσονται αρκετά περισσότερο από τη δική μας και θα συνεχίσουν. Γι' αυτό η εξωτερική ζήτηση ναι μεν θα βοηθήσει, αλλά δεν επαρκεί, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Εγώ προσπάθησα να τα πω αυτά και τα πιστεύω στεναρά ότι η χρήση μέσων πολιτικής για τον ανταγωνισμό είναι αναγκαία, που θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για την καινοτομία. Θα δημιουργήσουν λιγότερα εμπόδια και προσκόμματα για όσους θα εισέρχονται σε αυτή την αγορά για την, και θα βοηθήσουν για την ανάπτυξη. Αληθεύει αυτό, ιστορικά έχει αποδειχθεί, καταδειχθεί πιστεύω. Ούτε όμως αυτό πάλι μόνο του επαρκεί. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ενιαία εσωτερική αγορά με πλήρη απόδοση και αποδοτικότητα. Η ενιαία εσωτερική αγορά θα λειτουργήσει με πλήρη αποδοτικότητα πρώτον. Αν μειώσουμε στο μέγιστο τα προσκόμματα και τα εμπόδια που ακόμα σήμερα υπάρχουν στην αναλογική, στην κανονική αγορά όχι στην ψηφιακή, αλλά στην κανονική σημερινή κατάσταση αγοράς και στην εσωτερική ψηφιακή αγορά που μόλις ξεκινήσαμε με το έργο, με τον στόχο να μειωθούν, να συρρυκνωθούν αυτά τα εμπόδια. Όμως πιστεύω ότι επίσης χρειάζεται και η ζήτηση από την άλλη πλευρά. Και αν η εξωτερική ζήτηση δεν είναι επαρκής, τότε αρχίζει μια συζήτηση και κρεμεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί, να απαντηθεί. Δεν είναι πολύ ορθόδοξα, το έχω πει και το έχω πει κατηδίαν και δημόσια πολλέ φορέ. Πιστεύω ότι μεταξύ των οικονομιών που βρίσκονται στη δική μα περίμετρο τη αγορά, δηλαδή τη ενιαίας εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς, πρέπει να συζητήσουμε με σοβαρό τρόπο Πώ θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την εσωτερική ζήτηση στη ζώνη ευρώ επενδύσεων και κατανάλωση. Γιατί αν δεν γίνει αυτό δεν θα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα με τους λογαριασμού για την ανάπτυξη. Αυτή είναι η συνθετική μου απάντηση στην δική σα απλή ερώτηση. Στον κύριο Κορέντε Κάμπο. συμφωνώ απόλυτα μαζί σα, να ενισχυθούν οι εθνικές αρχές για τον ανταγωνισμό. Σίγουρα, στην συγκεκριμένη περίπτωση τη Πορτογαλίας νομίζω είναι και μία από τι συστάσει του προγράμματο της αποκαλούμενης Τρόικα, της ε, Τριμερούς Επιτροπής δηλαδή για την οικονομική βοήθεια προς την Πορτογαλία. Δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή. Υπάρχουν και άλλες χώρες ε, στις οποίες ε, τέτοιου είδους συστάσεις στο ευρωπαϊκό, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο ή σε συγκεκριμένα άλλα πλαίσια έχουν προταθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και όσον αφορά τη δική μας αρμοδιότητα ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2004 εργαζόμαστε μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού European Competition Network όπου πιστεύω ότι ο συντονισμός που έχει θεσπιστεί και θεσπίζεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής για τον Ανταγωνισμό, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή και των 27 ε, εθνικών αρχών για τον ανταγωνισμό θα πρέπει να προωθηθεί και να τονωθεί, να ενταθεί. Είναι ένα πρότυπο που πρέπει να αναλυθεί και να το δούμε παράλληλα με, μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο δημόσιων ε, φορέων και στο εθνικό επίπεδο και, στα κράτη, και στο ευρωπαϊκό επίπεδο όπου δεν συνεργάζονται και δεν συντονίζονται επαρκώς ώστε να υπάρξουν τα αναγκαία ωφέλη αμοιβαία κάθε φορά που συνερχόμαστε οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητάμε για τους κοινού μας στόχους, για τις δικές μας εμπειρίες και βιώματα, για τις βέλτιστες πρακτικές, για τα εμπόδια. Μαθαίνουμε ένας από τον άλλο και βγαίνουμε ενισχυμένοι από αυτό το εγχείρημα. Κάθε φορά που συνεργαζόμαστε για την αντιμετώπιση και επίλυση μια συγκεκριμένη περίπτωσης και όχι μόνο στα ευρωπαϊκά σύνορα εσωτερικά αλλά και με τις αρχές των ΙΠΑ, των, ε, Ιαπωνές, των, της Ιαπωνίας ή των, της Κορέας για να αντιμετωπιστεί το ένα ή άλλο πρόβλημα ενισχυόμαστε ο ένας από τις προσπάθειες του άλλου και βγαίνουμε όλοι ενισχυμένοι. Όταν έχουμε περίοδο δημοσιονομικών δυσχεριών και δυσκολιών δεν είναι ευχάριστο να λέμε στις χώρες ότι πρέπει να διαθέσουν περισσότερους πόρους για την καλύτερη λειτουργία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού τους, ανταγωνισμού που έχουν. Αλλά κάθε φορά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν βλέπουμε ότι ακολουθείται μια πολιτική ε, ενίσχυσης, εξυγίασης όταν μειώνονται τα κονδύλια για τις αρχές του ανταγωνισμού εμείς θα σηκώνουμε την κόκκινη κάρτα και θα λέμε αυτό είναι απαράδεκτο διότι αυτό θα σημαίνει ότι θα παίζουμε στο στρατόπεδο του εχθρού, του αντιπάλου και δεν θα κάνουμε αυτό το οποίο χρειάζονται οι οικονομίες που πρέπει να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Τώρα σε σχέση με την περίπτωση για τα τέλη ε, που επιβάλλονται στις επιστοτικές χάρτες, ε, κάρτες. Χρησιμοποίησα το επίπεδο των τελών που ισχύει στην Πολωνία σε αρκετές δημόσιες παρεμβάσεις μου που έκανα δημόσια για το πώς λειτουργεί το σύστημα πληρωμών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πολωνικό αυτό παράδειγμα το, το ε, χαρακτήρισα το πιο δαπανηρό, το πιο ακραίο στην Ευρώπη έχουμε μπροστά μας μέρος του προβλήματος. Αντιμετωπίζουμε αυτό το μέρος του προβλήματος και στην περίπτωση Mastercard με την προσφυγή στο δικαστήριο και με την περίπτωση της ε, των πιστοτικών κατών Visa που εκρεμεί εν μέρη και εν μέρη έχει ρυθμιστεί. Και έχουμε και το μίξ, το μείγμα των ε, διαφόρων πολυμερών ε, τελών που επιβάλλονται και επιβαρύνουν αυτές τις κάρτες είτε με τις εταιρείες αυτές που τις εκδίδουν και που εισπράττουν από τους ε, ε, χρήστες αυτών των καρτών μέσω συναλλαγών τους. Μέρος αυτών των τελών από τους ίδιους τους εκδότες αυτών των πιστοτικών κρατών καθορίζονται και εισπράττονται. Και δεν είναι πρόβλημα ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γνωρίζουμε όμως περιπτώσεις ε, που άνοιξαν από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού κατά τέτοιου είδους εκδοτών και θεσμικών οργάνων που σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος ε, έχουν θεσπίσει υπερβολικά τέλη, υπερβολικά υψηλά τέλη. Εδώ υπάρχει, ας το πω έτσι, στρέβλωση που, στην οποία καταλήγουμε μέσω αυτής της σύμπραξης. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε το θέμα της προστασίας καταναλωτών. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως προανέφερα, είναι θέματα προστασίας καταναλωτών που ξεπερνά το όριο της δικής μου αρμοδιότητας. Όμως για τα θέματα ανταγωνισμού, και δεν είναι η πρώτη φορά που τοποθετούμε δημόσια για αυτά τα πράγματα, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες να δημιουργηθούν εναλλακτικέ δυνατότητες όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληρωμών. Μια από τις πρωτοβουλίες αυτές ε, έχει ένα πολύ γνωστό ευρωπαϊκό όνομα. Είναι έτσι ελκυστικό με μια πρώτη ματιά, αν το δει έτσι. Αν δει κανείς όμως τους όρους και προϋποθέσεις ε, αυτών που προτείνουν ως εναλλακτικό ε, ε, πρότυπο πληρωμών, τότε βλέπει κανείς ότι τα τέλη τα οποία θέλουν να εισπράττουν ήταν ακόμα περισσότερα από τα σημερινά που καθορίζονται από παραδοσιακά εμπλεκόμενους παίκτες. Έχω κάθε σεβασμό για αυτό το φιλευρωπαϊκό όνομα ή την ονομασία αυτή, που χρησιμοποιείται για να ε, χαρακτηριστεί με ιδιαίτερο τρόπο ένα τέτοιο εγχείρημα, ένα τέτοιο πρόγραμμα. Όμως θα πρέπει με χαμηλότερα τέλη να γίνεται κάτι τέτοιο και όχι με υψηλότερα. Γιατί να προαγάγουμε ένα σύστημα με υψηλότερα τέλη αν οι ίδιες υπηρεσίες παρέχονται από άλλους. Δεν είναι αυτό δική μας δουλειά να το κάνουμε. Δική μας δουλειά είναι να χαμηλώσουμε, να μειώσουμε τα τέλη προς όφελος όλων. Προσπαθούμε να σκεφτούμε και να δούμε ποια θα ήταν επαρκή επίπεδα. Δεν είναι καθόλου εύκολο για τα τέλη αυτά αυτό. Ε, ξεκινούμε με μια μελέτη. Δεν είναι εύκολο να απαντηθούν τα ερωτήματα. Προσπαθούμε να θεσπίσουμε ένα επαρκές επίπεδο εισπραξης τελών. Και κατά το τέλος ε, όταν ολοκληρωθεί αυτή η δυσχερής ανάλυση και οι συζητήσει αυτέ, ίσω κάποια μέρα θα πρέπει να, να... να συμπεράνουμε ότι χρειάζεται ρυθμιστική δράση και παρέμβαση από πλευρά μα. Ίσως, ίσως βέβαια. Δεν έχει καθοριστικά απαντηθεί αυτό το θέμα. Και όχι μόνο εδώ τίθεται στην Ευρώπη, αλλά και στη ΣΥΠΑ επίση αυτό το ερώτημα και σε νόμο των ΙΠΑ υπάρχουν τέτοιες διατάξεις και προβλέψεις για παρέμβαση και διατάξεις, ρυθμίσεις θέμα το οποίο ε, είχε, έχει αποτέλεσμα αντίδραση τραπεζών λοιπά. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να συζητηθεί και να ρυθμιστεί. Και η διακριτική κατάσταση που δημιουργείται όσον αφορά τις ε, κρατικές συμβάσεις ε, είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσα στο πλαίσιο της συμμόρφωσης ή όχι με διατάξεις της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Ο συνάδελφός μου Μισελ Μπανιέ και η Γενική Διεύθυνση για τις Αγορές πρέπει να αρχίσουν τέτοιες προσφυγές αν δεν έχουν γίνει σεβαστές οι διατάξεις ε, για τις δημόσιες συμβάσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, ευχαριστούμε πάρα πολύ που για πρώτη φορά, όπως είπατε, είστε εδώ μαζί μας. Όπως βλέπετε, ήταν πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον πολλές ερωτήσεις. Ναι, ευχαρίστω να ξανάρθετε. Θα χαρούμε πάρα πολύ γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που έχουμε να συζητήσουμε και ένα θέμα που θα θέσω εγώ μαζί σας ε, όσον αφορά τις εξαιρέσεις για, ε, για, για το εμπόριο μέσω διαδικτύου. Την επόμενη φορά ε, θα το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι σας αξίζει ένα χειροκρότημα. Uh, um, Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την εισηγήτριά μας που τόσο σκληρά δουλεύει, την κυρία Κόμη, που την καθυστερήσαμε και την αφήσαμε να περιμένει για την παρουσίαση της έκθεσής της. Θα θέλαμε όμως να την καλέσουμε να, μας αρχίσει, να, μας, να ανοίξει τη συζήτηση όσον αφορά τις ε, τροπολογίες ε, για μια πολύ σημαντική πρόταση, ευρωπαϊκή τυποποίηση, Μα είχε παρουσιάσει την έκθεσή τη, οπότε θα ήθελα να σας καλέσω να μας παρουσιάσετε τις τροπολογίες και την πρώτη σας αντίδραση σε αυτές. Δεν ξέρω αν ο κύριο Κρόιτσμαν είναι εδώ ή ο κύριος Μάντες. Ήρθατε πάλι στην Επιτροπή μας, σας είχαμε εξορίσει στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Μήπως είχατε έρθει για να μιλήσετε, έχετε έρθει για να μιλήσετε εκ μέρους του κυρίου Μάντες. Πολλοί συνάδελφοι δεν είναι εδώ. Ο κύριος Σαμπίνη επίσης απουσιάζει. Λιλιάνα Μπρίγκμαν και κύριε Φάισερχομ, ε, καλώς ήρθατε. Είστε οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ε, το θέμα αυτό. Και ο κύριος Τόμσον είναι εδώ από το Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Ε, κυρία Τόμσον, συγγνώμη. Α, κύριος, διορθώνει ο πρόεδρο. Κύριος Τόμσον τελικά. Κύριος. Είστε από το Συμβούλιο, αλλά δεν είστε κυρία, είστε κύριος Τόμσον. Αν θέλετε κι εσείς ε, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Κύριε Ακόμη, σας δίνουμε το λόγο για να μας παρουσιάσετε μια πρώτη άποψη των τροπολογιών. Λοιπόν, είχα περιορισμένο χρονικό διάστημα διότι πήρε το χρόνο επί το ο Σαλμούνιο, αλλά πρέπει να επεκταθώ κάπως τελικά, διότι οι τροπολογίες είναι πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες, ζητώ συγγνώμη, αλλά θα κλέψω κάποια λεπτάκια, λεπτάκια παραπάνω. 21 ε, ε, Μαρτίου θα ψηφιστούν οι τροπολογίες. Σήμερα ε, ψηφίστηκαν στην Επιτροπή Βιομηχανίας και πάνω απ' όλα σας ευχαριστώ για τις τροπολογίες που προτείνατε, διότι σίγουρα επικεντρώνονται επί των εργασιών που προωθούμε. Διάβασα, ανάλυσα προσεκτικότατα τις τροπολογίες και έχουν πλήρες όραμα τελικά των διαφόρων... Έχω γενική εικόνα των απόψεων. Ολοκληρώνεται η εργασία, αλλά ξεκίνησε πολύ παλιά. Θέλουμε να ετοιμάσουμε συμβιβασμούς επί των βασικών σημείων, διότι θέλω να προχωρήσω όπως έκανα τώρα Όπω ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, προσπαθώντα να συνεργαστούμε, οι σκιώδεις συγητές και εγώ, για να βρούμε λύσεις ε, που υποστηρίζονται του περισσότερου δυνατού για να έχουμε αποτελεσματικό αποδοτικό μέσο και για του καταναλωτέ και τι ευρωπαϊκέ ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είναι βασικό μου στόχος. Παρακολούθησα και τι εργασίε του Συμβουλίου προσεκτικά, διότι στόχο μου και όλων μα, πιστεύω, είναι να υιοθετήσουμε αυτόν τον κανονισμό στην πρώτη ανάγνωση. Θα περάσω τώρα αναφερόμενοι σημείο προς σημείο, δεν θα αναφερθώ και στις 220 τροπολογίες χωριστά, αλλά θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω σε μακροομάδες. Πρώτα απ' όλα, τομέα εφαρμογή του κανονισμού. Επεξεργαζόμενοι το σχέδιο εκθέσεως το σκέφτηκα πολύ και επέλεξα να δεχτώ την επιλογή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, να μην τίθεται όρια όσον αφορά ε, τη μέθοδο εφαρμογή. Προτείνω μια τροπολογία για να προστεθεί μια ιδεολογική σκέψη που αφορά τα ελεύθερα επαγγέλματα εντό των επαγγελματικών προσόντων. Ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαφυλάξει το πνευματικό και δημιουργικό χαρακτήρα των υπηρεσιών που παρέχονται. Είναι δύσκολο να ισχυριστούμε ότι ένα τομέα μπορεί να αποκλειστεί εκ των προτέρων το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού διότι τα πρότυπα μπορεί ενδεχομένω να είναι κάτι που ισχύει για όλους τους τομείς. Αυτό είναι βασικό σημείο κλειδί πρέπει να αναλυθεί. Γι' αυτό το λόγο δεν ήθελα να θέσω κάποια όρια όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής. Αφήνοντας την απόφαση αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αξιολογήσει σε, αυτή, σε κάθε περίπτωση τι θα κάνει αφού έρθει σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Όσον αφορά αυτό το θέμα, ε, παρουσιάστηκαν πάρα πολλές τροπολογίες από συναδέλφους διαφόρων πολιτικών ομάδων ε, που ήθελα να εξαιρέσω κάποιου τομεί, στον ιατρικό τομέα, τη υγεία, των ελευθέρων επαγγελμάτων. Εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε εμεί σε θέση να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια, έναν αποκλεισμό ενό ή άλλου τομέα. Εγώ προσανατολίζομαι στο μη προβλέπω καμία εξαίρεση ρητή τομέων, αλλά αξιολογήσω τη δυνατότητα να περιορίσω τους υπηρεσίες που σχετι... σε... σε αυτές που σχετίζονται με αγαθά. Θα δούμε ποια είναι τα κριτήρια. Δεύτερον, ορισμοί. Όσον αφορά του ορισμού, υπάρχουν διάφορε προτάσει που τι εκτιμώ και ευχαριστώ για τι προτάσει Διαβελτιώνουν όλοι το προτινόμενο κείμενο, όλε οι προτάσει στο βελτιωμένο κείμενο. Όλα αφορούν τι οργανώσει τυποποίηση. και λέει αναγνωρισμένοι οργανισμοί τυποποίηση με τη λέξη αναγνώριση. Δεν συμφωνώ με την τροπολογία 122, διότι ένα πρότυπο είναι πάντα εθελοντικό εξορισμού. Και καμιά φορά α, ε, μπορεί να μπει σε πράξη δεσμευτική ένα πρότυπο, αλλά δεν προέρχεται από εκεί ο δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά από την οθετική πράξη που συνδεύει το κείμενο. Ε, δεν θέλουμε. Ε, είναι θελοντικό λοιπόν το σύστημα. Πέστε μου αν πηγαίνω πολύ γρήγορα, θα προσπαθήσω να μην προχωρώ πολύ γρήγορα. Τρίτο σημείο. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών Θα προχωρήσω πιο αργά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το τρίτο σημείο συνδέεται με την συμμετοχή ε, των ε, stakeholders, των εμπλεκομένων μερών. Ε, είμαι υπέρ της συμμετοχής αυτών των εμπλεκομένων μερών και να αναφέρονται και άλλες κατηγορίες. Παραδείγματο χάρη είδαμε τους εργαζομένους, τους αναπήρους, τις οργανώσεις, τις ενώσεις των καταναλωτών. Όλοι αυτοί θα πρέπει να συμβάλλουν με σημαντικό και αποφασιστικό τρόπο στην εφαρμογή των προτύπων. Αυτός ο κανονισμός δεν έχει σαν στόχο μόνο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά θέλει να δώσει μία συνεισφορά και στην κοινωνική ένταξη. Ε, και αυτό το πέρασμα κάνουμε. Όσον αφορά το δικαίωμα ψήφου στο παράρτημα 3 στις οργανώσεις, δεν είμαι υπέρ, διότι θέλω να εξασφαλίζω την αποτελεσματική ε, συμμετοχή σε εργασίες. Αυτό θέλω να κάνω, να έχουμε επαρκή εκπροσώπηση των διαφόρων συμφερόντων στη διαδικασία της τυποποίησης. Παρά να υπάρχει μια συμβολική αναγνώριση που μετά στην πραγματικότητα πολλές φορές δεν έχει πρακτική εφαρμογή και εκχωρείται σε άλλους. Η τέταρτη πτυχή είναι τα νέα άρθρα όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σημείο κρίσιμο για όλους μας, ένα σημείο επί του οποίου το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφραστεί με έναν τρόπο πάρα πολύ στεναρό και είμαι ικανοποιημένη που πολλοί συνάδελφοι εξέφρα, ε, υπέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση τροπολογίες. Μπορώ να πω ότι είναι μια επιτυχία αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο, το φιλόδοξο και το σημαντικό όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αν και πρέπει να παραδεχτώ ότι όσον αφορά αυτό το θέμα υπήρξαν αποκλήσεις ή αντίθετες απόψεις όσον αφορά την ελεύθερη πρόσβαση στην ε, δραστηριότητα της τυποποίησης. Υπήρξαν προβλήματα ερμηνευτικά και επ' αυτής της συγκεκριμένης πτυχής ε, προσπάθησα να διευκρινίσω ε, τι εννοούμε με την ελεύθερη πρόσβαση. Τι, τι σημαίνει αυτό. Ελεύθερη πρόσβαση δεν σημαίνει ελεύθερη πρόσβαση στα πρότυπα, δηλαδή ε, ελεύθερα, ελεύθερη τυποποίηση δωρεάν, αλλά οι εργασίες επεξεργασίες των προτύπων, που είναι κάτι διαφορετικό, ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό. Γι' αυτό μετά αναπτύξαμε και εξηγήσαμε τον ορισμό και τις συστάσεις και την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής 361 του 2003 όσον αφορά την μέση επιχείρηση, μικρή επιχείρηση και πολύ μικρή επιχείρηση. Κάποιο είπε ότι η ελεύθερη πρόσβαση στι επιχειρήσει θα κόστιζε πάρα πολύ και θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα σε εθνικό επίπεδο. Όπου οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι το βασικό υπόστρωμα τη βιομηχανία. Και εδώ προτάθηκαν δύο εναλλακτικέ. Η πρώτη είναι αυτή του, του, περιορισμού της ελεύθερης πρόσβασης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και η άλλη να προβλέπεται η εφαρμογή ειδικών τελών χωρίς να γίνεται διαφοροποίηση με βάση το μέγεθος της επιχειρήσης. Αυτές είναι οι δύο προτάσεις. Επ' αυτού θα ήθελα να ακούσω βεβαίως και την άποψη των άλλων σκιωδών ε, και να συμφωνήσουμε επ' αυτού. Να μου πούνε με τι συμφωνούν. Λοιπόν, θα πρέπει να πολεμήσουμε υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κυρίως όσον αφορά τη συμμετοχή που θα πρέπει να έχουν εντός της διαδικασίας τυποποίησης, διότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο συγκεκριμένο και αποτελεσματικό, ούτω ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και να μην ε, υποκύπτουν στις ε, αποφάσεις των μεγάλων απλώς. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποστηρίξει αυτή την ε, προσέγγιση, τα μέτρα που προτείνω για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν τα εφεύρα εγώ, δεν ξύπνησα πρωί-πρωί ε, και φίβρα αυτό. Ακούσαμε ε, κατά τη διάρκεια της ακρόασης ε, τι γίνεται στη Γαλλία, πώς εφαρμόζεται στη Γαλλία αυτό. Άρα είναι δυνατό να γίνει. Μπορεί να γίνει, ήδη γίνεται με πολύ καλά αποτελέσματα. Έκανα την επιλογή να, θες, να κάνω δεσμευτικά τα μέτρα βάζοντας το στον κανονισμό πραγματικά, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε σαφή κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να κινηθούμε. πώ τα που πρέπει να κινηθεί η ευρωπαϊκή τυποποίηση και αυτό είναι ο στόχο του κανονισμού. Συγκεκριμένε τεχνικέ. Αυτό είναι ένα άλλο σημείο το οποίο δημιούργησε δυσκολίες όσον αφορά τον όρο χρήση και αναγνώριση. Πρέπει να τα διευκρινίσω αυτό, διότι επέλεξα τη λέξη χρήση και όχι αναγνώριση. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πήγαινε προς την κατεύθυνση αύξησης των προτύπων, των ειδικών ε, τεχνικών σε επίπεδο ε, προτύπων. Ε, με κριτήρια που είναι στο παράδειγμα 2. Εγώ ήθελα να συνεχίσουμε να αποκαλέψουμε αυτά ειδικέ τεχνικέ και όχι πρότυπα, διότι υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ των πτυχών. Το στάνταρ, το πρότυπο είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο, πολύ πιο περίπλοκη έννοια. Μια πτυχή που απαιτεί ε, και μια διαδρομή, ε, αν θέλετε, και διαδικασία πιο δύσκολη και πιο μακρά. Εάν οι τεχνική. Ε, δεν γίνει, ε, γίνει πρότυπο, τότε δεν χρειάζεται η έννοια αναγνώριση. Γι' αυτό έβαλα χρήση. Σε αυτό το σημείο υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις και προτάσεις. Θα ήθελα να ακούσω φυσικά ποιε είναι οι απόψη σας για να μπορέσω να καταλάβω καλύτερα την επιχειρηματολογία που μπορεί να προβληθεί όσον αφορά τη χρήση του όρου χρήση. Η αρχή τη συνοχή θα ήθελα να πω ότι εδώ δεν είμαι υπέρ αυτή, διότι από την πλευρά είναι κάτι σημαντικό να υπάρχει διαφορά μεταξύ προτύπου και ειδικών τεχνικών στο συγκεκριμένο τομείο, αλλά δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε όμω φραγμό στην ανάπτυξη των ειδικών τεχνικών. Εάν υπάρχουν και τις δέχεται η αγορά, δεν μπορούμε να το ε, αρνηθούμε. Μιλάμε για ένα θελοντικό σύστημα, άρα προς αυτή την κατεύθυνση που προτείνω πρέπει να κινηθούμε. Έβδομο σημείο, και για να μην σας κουράζω ε, κράτησα σχεδόν το χρόνο είναι το θέμα του φόρουμ και της πλατφόρμας ε, των πολλών εμπλεκομένων, multi-stakeholders. Ε, εγώ δεν είμαι αντίθετη όσον αφορά τη δημιουργία ενός φόρουμ ή μιας πλατφόρμας των stakeholders, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ενταχθεί εντός του κανονισμού στο διατακτικό διότι δεν πρέπει να δημιουργούμε ε, υπερκατασκευές που τελικά επιβραδύνουν τη διαδικασία. Πρόκειται περί κανονισμού, είναι κάτι δικό. Οι επιχειρήσεις το χρηματοδοτούν, επιθελοντικής βάσης εφαρμόζεται και γι' αυτό δεν θέλω να δημιουργήσουμε και, άλλ, και άλλους φορείς. Ε, στο μέλλον βεβαίως θα μπορέσουν να δημιουργηθούν αν απαιτείται και αν θεωρήσουμε κάτι σκόπιμο. Δεν πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να εντάσσεται Σκέφτεται ένα ναι ή ένα όχι εντός ενός κανονισμού κάτι που συνεπάγεται κάποια δέσμευση. Η πτυχή της χρηματοδότησης, α, συγγνώμη, επ' αυτού του σημείου ε, πιστεύω ότι είναι καλύτερο να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα προχωρήσει προς την διαβούλευση, διότι είναι τεχνικό ειδικό πλαίσιο αυτό και πιστεύω ότι αρμόζει περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει και φτάνω στο τελευταίο σημείο που είναι αυτό της χρηματοδοτήσεως. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια μόνο όσον αφορά τη χρηματοδότηση εν γέννη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσον αφορά τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Τυποποίηση. Ε, δεν θελήσαμε να τροποποιήσουμε τις προδιαγραφές οι οποίες προτείνονται και που είχαμε αποδεχτεί ως ιδέα. Σε αυτή την πρώτη φάση ζωής του κανονισμού οι κανόνες θα πρέπει να είναι λίγο πιο άκαμπτοι για να διαθρώσουν καλύτερα την όλη διαδικασία της τυποποίησης. Θα ήθελα όμως να επαναλάβω στεναρά ότι πιστεύω προσωπικά ότι τα πρότυπα θα πρέπει να πλουστευτούν στο μέλλον και η χρηματοδότηση θα πρέπει να εδράζεται επί προσέγγισης οικονομικής και αποκλειστικά και να μειωθεί η γραφειοκρατία που προβλέπεται τώρα. Και γι' αυτό πρότεινα μια ρήτρα επανεξέτασης μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2015. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτή την ανάγκη απλούστευσης και απογραφειοκρατικοποίησης. Ζητώ συγγνώμη επειδή έκλεψα χρόνο. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους. Θα να σας πω ότι στόχος μου σε αυτή τη φάση είναι να δημιουργήσουμε ένα κείμενο σύντομο, περιεκτικό, ακριβές νομικά. Πρόκειται περί κανονισμού, άρα χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβείς όρους για να αποφύγουμε εσφαλμένες ερμηνείες ή ερμηνευτικές αμφιβολίες. Πιστεύω ότι είναι ένας κανονισμός που απαιτεί, όπως και ο κύριο Ταλιάνη ότι χρειάζεται γρήγορα να εφαρμοστεί και για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και για το παραγωγικό σύστημα που χρειάζεται ε, απόλυτα την έγκριση αυτού του κανονισμού και αυτά και αφήνω το λόγο σε εσά. Ευχαριστώ. No, I think the whole idea is... Νομίζω ότι η ιδέα είναι πραγματικά να γίνει μια συζήτηση για τις τροπολογίες. Γι' αυτό άλλωστε το εγγράψαμε σε μερίσια διάταση του. Άλλωστε θα έχουμε εξυμβαστικέ τροπολογίε ε, που πάλι θα τι συζητήσουμε όσο χρειάζεται. Ο κύριος Κρόιτσμαν πρέπει να επιστρέψει στην ε, κύρια επιτροπή του. Μήπως ε, η κυρία Σάλτεμορ μπορεί να μου, δώσει, να μου επιτρέψει να του δώσω το λόγο. πήγα στην άλλη επιτροπή, είμαι λίγο ε, ξένος στην άλλη επιτροπή, είμαι εξοικειωμένος περισσότερο με την επιτροπή εδώ. Θα ήθελα πρώτα να θέσω ένα ερώτημα για τη χρηματοδότηση. Πρέπει να είναι σαφές ότι θα καταλαβαίνουμε πολύ καλά ε, ότι έχει νόημα να μειώσουμε το κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλοι θα θέλαμε να το υποστηρίξουμε αυτό, αλλά όταν ε, ένας φορέας ε, τυποποίησης χρειάζεται πόρους για να λειτουργήσει, το ερώτημα είναι κατά πόσο θα μπορέσει να λειτουργήσει όντως. Εγώ σε γενικέ γραμμέ είμαι πολύ υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα το γνωρίζετε, αλλά όταν ένα φορέα δεν μπορεί να λειτουργήσει επειδή δεν έχει πόρου, δεν έχει χρήματα, τότε δεν έχει κανένα νόημα. Και αυτή είναι η άποψή μου για το θέμα αυτό. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να αναφερθώ στα ζητήματα που μου ζήτησε να αναφέρω ο κύριος Μάντερς σε γενικές γραμμές ε, είναι ικανοποιημένος με την έκθεση της κυρίας Κόμη και τις τροπολογίες ε, και το πρωί όταν ψηφίσαμε στην Επιτροπή ε, Βιομηχανίας ήταν πολύ καλό το αποτέλεσμα και πιστεύουμε ότι θα μπορέσετε να συγκεράσετε τις απόψεις και των δύο επιτροπών. Του αρέσει πολύ η διάταξη η διάταξη για το standstill. ο συνάδελφος είναι επίσης ε, υπέρ ε, της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών σε εθνικό επίπεδο. Επίσης είναι υπέρ ε, της, του ενισχυμένου ρόλου των κυβερνήσεων στη διαδικασία τυποποίηση, όπως επίσης και υπέρ του φόρουμ συμμετοχής των ε, ενδιαφερομένων ε, μερών. Ο κύριος Μάντερ θα, ήθελε, Μάντερ θα θέλει να τονίσει ιδιαίτερο στο γεγονό ότι πρέπει να υπάρξει ασφάλεια δικαίου σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε και τι διαδικασίες προσφυγής. Ελπίζουμε λοιπόν ε, η ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες να, να είναι καρποφόρα και θα ήθελα να προσθέσω ότι για την ενιαία αγορά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Ελπίζω λοιπόν ότι η Λάρα Κόμη θα μπορέσει να ε, υποστηρίξει τις σχετικές αλλαγές στην νομοθεσία. Η νομοθεσία μπορεί να αλλάζει μόνο προς το καλύτερο. Έτσι μου έχουν πει θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσω τη ψηφοφορία για να βελτιώσουμε την νομοθεσία. Ναι, ευχαρίστω μπορείτε πάντοτε να ζητάτε καταφύγιο στην Επιτροπή μας. Ε, η κυρία... Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κόμη για την παρουσίασή της και ε, είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε συμβιβαστικές τροπολογίες, άλλωστε δεν διαφωνούμε τόσο πολύ επί πολλών θεμάτων. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα όμως για το πεδίο εφαρμογής, για τις υπηρεσίες συγκεκριμένα, κατά πόσο θα πρέπει να είναι τμήμα της δουλειάς για την τυποποίηση ή όχι. Εγώ από την αρχή το λέω αυτό. Είμαστε κάπως ε, επιφυλακτικοί στους σοσιαλδημοκράτες για το θέμα αυτό, στους σοσιαλιστές για το θέμα αυτό, γιατί θεωρούμε ότι κάποιοι τομείς δεν έχουν συμπεριληφθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να το συζητήσουμε και η κυρία Ρούλε έχει ε, υποβάλει τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή και ο κύριος Φαμπ. Οπότε πρέπει να δούμε οπωσδήποτε τι θα κάνουμε εν προκειμένου. Πολλοί τρόποι υπάρχουν να επιλύσουμε το πρόβλημα, αλλά κατά την άποψή μου θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τη συζήτηση αυτή στη συζήτηση με την ε, πλατφόρμα συμμετοχής πολλών ενδιαφερομένων μερών. Γιατί αν θα συμπεριλάβουμε τις υπηρεσίες ε, στην ε, εργασία για την τυποποίηση, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συμμετέχουν. Πρέπει να διαβουλευτούμε με όλους του ενδιαφερομένους. Αν λοιπόν μπορούμε να συνδέσουμε τη, συζήτηση για την πλατφόρμα για τους ενδιαφερομένους ε, ε, και για το, με, το, με το πεδίο εφαρμογής, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τη λύση. Για διάφορους άλλους τομείς, νομίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να βρούμε λύση. Θα ήθελα να πω κάτι ε, σε σχέση με αυτό που είπε ο συνάδελφο προηγουμένω για το κόστο και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Όλοι συμφωνούμε ότι η εργασία για την τυποποίηση είναι ένα εθελοντικό, ιδιωτικό σύστημα. Απ' την άλλη όμως πιστεύουν όλοι ότι πρέπει να αποφασίσουμε ποιο θα είναι το κόστος, ποια θα είναι η τιμή για να μπορεί κανείς να συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα βρίσκω ότι αυτά τα δύο πράγματα δεν συνδυάζονται σωστά. Όλοι θέλουμε λοιπόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία, αλλά από την άλλη οι μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις ε, είναι περίπου το 80% των ευρωπαϊκών εταιριών. Δηλαδή το 20% πρέπει να πληρώσει για όλη τη δουλειά της τυποποίησης. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βγούμε από αυτό το αδίέξοδο. Ένας τρόπος θα μπορούσε να είναι, να πούμε για παράδειγμα, ας κάνουμε κάτι για τις, ε, για τους, ε, για τις, για τις εταιρείες που απασχολούν 10 ή λιγότερους ε, υπαλλήλους. Γιατί διαφορετικά μιλάμε ε, για όλες τις εταιρείες με προσωπικό κάτω των 250. Είναι πάρα πολλές αυτές οι επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν για τις πολύ μικρές, πολύ πολύ μικρές επιχειρήσεις μια λύση. Είναι πάντως ένα εθελοντικό σύστημα, ιδιωτικό και πρέπει να είμαστε λίγο, λίγο προσεκτικοί όσον αφορά τις τιμές ε, συμμετοχή ε, στι σχετικέ εργασίε. Είπα σε γενικέ γραμμέ τι θεωρώ σημαντικό, αλλά είμαι βέβαιη Ούτω ή άλλω, εξ όσων γνωρίζω, έχουμε ήδη μια συζήτηση προγραμματίσει με του σκιώδει εισηγητές και πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Βέβαια, δεν πρέπει να θέσουμε ένα αμφιβόλο το αποτέλεσμα. Πρέπει να ε, έχουμε και το χρόνο να βρούμε τι σωστέ λύσει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κόμη. Είναι εξαιρετική η δουλειά της. Ήταν πολύ καλή από την αρχή, πολύ καλή και η συνεργασία μαζί της και γι' αυτό πιστεύω ότι θα καταλήξουμε επί πολλών σημείων σε συμβιβασμό. Μιλήσατε για αυτή την πλατφόρμα ε, πολλών ενδιαφερομένων μερών. Νομίζω ότι την απορρίψατε. Όμως εγώ πιστεύω ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πεδίο εφαρμογής. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι οι υπηρεσίες ή θα ενσωματωθούν σε συγκεκριμένη έκθεση χωρίς καμία ρύθμιση και ότι δεν έχουμε κανένα όργανο, κανένα φορέα πριν από την τυποποίηση στον τομέα των υπηρεσιών. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Δεν έχουμε πουθενά ορίσει το market driven. Είπαμε ότι πρέπει να είναι ένα εθελοντικό σύστημα να βασίζεται στην αγορά, αλλά ποτέ δεν το έχουμε ορίσει. Ακούω από πολλούς ε, ενδιαφερομένους ε, ε, φορείς ότι δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται απαιτήσει τυποποίησης που θα έπρεπε να την κάνουν διαχείρισης από άλλους φορείς. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μία ακόμα διαφούλευση ε, επί του θέματος αυτού. Λέτε ότι πρέπει να αφήσουμε το θέμα στην Επιτροπή. Ναι, αλλά εγώ μίλησα με την Επιτροπή και από ό,τι κατάλαβα η Επιτροπή δεν το θέλει καθόλου αυτό. Αν λοιπόν αφήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό στην Επιτροπή δεν πρόκειται να υπάρχει τέτοιου είδους πλατφόρμα ε, πολλαπλή συμμετοχή που όπως την αναφέρατε. Όμως πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο, πώς μπορούμε να δράσουμε ώστε να παίρνουμε αυτές τις ε, αποφάσεις ε, τις οποίες ε, βασίζουμε πάση περιπτώσει στην αγορά. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Εκ μέρους του συναδέλφου, Νομίζω ότι σε γενικέ γραμμέ ε, έχουν δίκιο στα σχολιά του συνάδελφοι και συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που είπε ε, η κυρία Σουάλντε Μόζε για τη χρηματοδότηση. Είναι πάρα πολύ σαφέ ότι είναι σημαντική η πρόσβαση για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει ε, Η όλη διαδικασία τυποποίηση πρέπει να χρηματοδοτείται ανεξαρτήτως, ενδεχομένω με κάποια δημόσια υποστήριξη. Αλλά δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε τη βάση του όλου εγχειρήματο και νομίζω ότι κάποιε από τι ιδέε ότι κάποιοι φορεί ε, ούτως ή άλλως ε, ε, δίνουν δωρεάν κάποια πρότυπα τυποποίησης για να δουν πια τις εξυπηρετούν ώστε να τα αγοράσουν στη συνέχεια. Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν λογικό συμβιβασμό όσον αφορά τώρα τις υπηρεσίες. Θέλουμε την αναγνώριση, όμως δεν θέλουμε να, να ξεφύγει από τον έλεγχο η όλη διαδικασία. Η Επιτροπή μας λέει ότι υπάρχει ε, εξέλιξη σε μερικούς τομείς ε, για... Ε, διότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι πιο εύκολο να αντικαταστήσουν το ένα το άλλο Καλή ιδέα είναι βέβαια τα εθελοντικά ε, πρότυπα, υπάρχουν ήδη στην ε, ε, σχετική νομοθεσία, όμως μου φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφής. Θα μπορεί να, μπορεί να βασίζεται είτε στην αγορά είτε στο δημόσιο συμφέρον. Ακούσαμε λοιπόν πολλές παρεμβάσεις ε, οι οποίες προσπαθούν να οριοθετήσουν κάπως τα πράγματα και δεν χρειάζεται αυτό γιατί ούτως ή άλλως ε, θα περάσουμε σε τυποποίηση όταν υπάρχει δημόσιο συμφέρον, ε, κυρίως για τα προϊόντα και ενδεχομένως να υπάρξει και επέκταση και σε άλλους τομείς. Δεν είμαι λοιπόν ιδιαιτέρως υπέρ αυτών των πολύ λεπτομερών περιγραφών ή ορισμών και το λέω αυτό ε, απευθυνόμενος προς τον κύριο Σφάμπ γιατί εκείνος είναι ο ειδήμων τέτοιου είδους ε, ορισμών. Είμαι σίγουρος όμως ότι η κυρία Κόμη θα καταφέρει να συμβιβάσει τα πράγματα. Και ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θέσω ε, η συμμετοχή των δημοσίων αρχών. Νομίζω ότι έχουμε τροπολογίες που λένε ότι πρέπει να ενθαρρύνουν, πρέπει να ενθαρρύνουμε τις δημόσιες αρχές, αλλά δεν χρειάζεται εμείς ε, να ζητήσουμε από καμία δημόσια αρχή να συμμετέχει οπωσδήποτε στην όλη διαδικασία. Τώρα, βέβαια, ε, επί τη βάση του γεγονότος ότι ε, ο μοχλός της όλης διαδικασίας είναι το δημόσιο συμφέρον Αυτά ε, είναι τα σχόλια που θα ήθελα να κάνω εγώ. Ο συνάδελφος φαντάζομαι θα υποβάλει περαιτέρω σχόλια και στην κυρία Κόμη. Η κυρία Καλινιέτε θέλει να πάρει το λόγο. Υπάρχει κανένας άλλος που θέλει να πάρει το λόγο πριν δώσω μετά ε, το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, κυρία Καλινιέτε. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κόμη για την ε, πάρα πολύ καλή προσέγγιση της σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τις ανησυχίες ε, της ίδιας της εισηγήτριας. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στη, στο πρόγραμμα μετάφρασης των εθνικών προτύπων που είναι ε, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για χώρες όπως η Λιτωνία. Δεν συμφωνώ με τις τροπολογίες 143 και 147 γιατί τέτοιου είδους απέτηση ε, θα είναι πολύ πιο δαπανηρό για τη διαδικασία τυποποίησης και θα δημιουργήσει επιπλέον διοικητικό ε, άχθος ε, στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης. Αυτό που προτείνω ως εναλλακτική λύση είναι να εξασφαλίσουμε να μεταφέρονται οι τίτλοι στις γλώσσες των εθνικών οργανισμών τυποποίησης. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντικό η απέτηση αυτή να μην συμπεριλαμβάνει την προϋπόθεση της μετάφρασης. Και να επανεπισημάνω ότι οι τροπολογίες 154, 156 και 171 με βρίσκουν σύμφωνοι. Ο, ο όρος «insures» εξασφαλίζει θα πρέπει να αλλάξει με διευκολύνει ή ενθαρρύνει facilitates or encourages. Γιατί ένας από τους στόχους της τυποποίηση δεν είναι μόνο η διαφάνεια και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στην τυποποίηση, αλλά και η εθελοντική συμμετοχή ε, στην τυποποίηση. Υποστηρίζω επίση όλε τι τροπολογίε ε, στι οποίε ο στόχο τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαδικασία τυποποίηση ε, έχει συμπεριληφθεί. Αλλά είμαι κάπως επιφυλακτική γιατί δεν υπάρχει αξιολόγηση του οικονομικού αντικτύπου. Για παράδειγμα, ποιο θα είναι το κόστος ε, ελεύθερης πρόσβασης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, στη διαδικασία τυποποίησης και όπως είπε η κυρία Σιολδεμόζε, Καταλαβαίνω τη σημασία αυτής της πρόσβασης. Η καλή, η σωστή λύση είναι ενδεχομένως από όλε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να διαλέξουμε τι πολύ πολύ μικρέ επιχειρήσει. Αυτό ενδεχομένω να αποτελεί τη σωστή λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Καλνιέτε. Να ε, δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα μιλήσει και πάλι η συγγήτρια για να μας πει το χρονοδιάγραμμα. Πέντε η ώρα η κυρία Κορόλα θα ε, αναλάβει την Προεδρία γιατί πρέπει να συναντηθώ με την Επίτροπο Βασιλείου και να συζητήσω μαζί της. Αλλά θα παρακολουθώ βέβαια τις συζητήσεις μας. Κυρία Μπρίγκμαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εξ ονόματος της Επιτροπής να ευχαριστήσω θερμά για την έκθεση αυτή και εμείς ε, εξετάσαμε τις τροπολογίες και θεωρούμε ότι οι κύριοι στόχοι, οι κυριότεροι στόχοι του κανονισμού όσον αφορά την συνέχιση πάνω στα σωστά θεμέλια τυποποίησης θα πρέπει να έχουμε ένα ευρύ φάσμα αναγκών στο οποίο θα ανταποκριθούμε βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, καλύτερη συμμετοχή, τυποποίηση, θέματα που είναι ευρέως αποδεκτά τούτων λεχθέντων και άλλα σημαντικά θέματα τα οποία τίθενται στις τροπολογίες που συντάχθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής αυτής καλωσορίζουμε εμεί ιδιαίτερα αυτές τις τροπολογίες. Την ανάγκη για παράδειγμα να συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα, Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης να συμπεριλαμβάνεται και να τονίζεται η ανάγκη για τον γυρασμένο υπερήλικα πληθυσμό και τις ανάγκες του και των ενώσεων καταναλωτών υπό το παράτημα 3 της πρότασης της Επιτροπής. Ιδιαίτερα εκτιμούμε τις προσπάθειες να τονιστεί η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να βελτιωθεί περαιτέρω ο ρόλος τους στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης. Και αυτό είναι ένα μέλημα το οποίο συμμερίζεται απόλυτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης εκτιμούμε την έμφαση που τίθεται στην πρόσβαση διεθνώς στην τυποποίηση. Ανταποκρινόμαστε στη δική μας ανακοίνωση σε λεπτομέρειες, όμως ε, θα πρέπει να δούμε και εξειδικευμένα τις πτυχές αυτές του κανονισμού ξεχωριστά. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποιες ξεχωριστές τροπολογίες, όπως προτάθηκαν από τους ευρωβουλευτές μέλη αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, που αφορούν πρώτα απ' όλα το θέμα των υπηρεσιών που προαναφέρθηκε από προλαλήσαντες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις τροπολογίες αυτές που θέλουν να στενέψουν το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού επικεντρωνόμενες σε κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες ή αποκλείοντας ε, την, ε, τις περιπτώσεις ε, περίθαλψης και υγείας. Νομίζουμε ότι όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι περιττοί και θα μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Μια και δεν μπορούμε να προδικάσουμε πλήρως όλες τις ανάγκες, μελλοντικές ε, ανάγκες των ε, πολιτικών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτό στοχός ε, η τυποποίηση, αλλά ένα μέσο, ένα εργαλείο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναπτυχθούν προδιαγραφές από τις Ευρωπα... τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την νομοθεσία και την ποιότητα που θα πρέπει αφ' αυτό να σέβονται τις προτεραιότητες που θεσπίζονται από τις ίδιες τις συνθήκες της Ένωσης. Πρότυπα, πρότυπα υπηρεσιών πρέπει να είναι εθελούσιου, εθελοντικού χαρακτήρα και όχι υποχρεωτικά, ενώ σε σχέση με τα προϊόντα και άλλες υπηρεσίες δεν πρέπει να αποκλείονται απριόρι ε, εξορισμού. Όσον αφορά τροπολογίες που αφορούν την εμπλοκή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εμπλεκόμενων από πλευρά του στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης. Καλωσορίζουμε την ε, ανάγκη να υπάρχει ολοκλήρωση και να εντάσσονται και αυτοί. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε να μην διακυβευθεί το πρότυπο το οποίο έχει υιοθετηθεί από τους εθνικούς θεσμούς τυποποίησης και για κάποιες άλλες τροπολογίες που συνδέονται με τις απαιτήσει ε, όσον αφορά εξειδίκευση ε, διατάξεων για τον τομέα ICT περίπτωση παρατήματος 2 έχουμε σημειώσει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που θέλουν να εισαγάγουν στον κατάλογο, στον πίνακα των κριτηρίων που θα εντάσσονται σε αυτό το σχέδιο κανονισμού αναφορές σε δύο άλλα νέα στοιχεία συνεκτικότητα το ένα και νομιμοποίηση το άλλο. Για την συνεκτικότητα η συνοχή. Πιστεύουμε πράγματι ότι η συνεκτικότητα, η συνοχή είναι ένας γενικότερος στόχος. Θέλουμε να υπάρχει συνεκτικότητα και συνοχή σε σχέση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και προτύπους. Δεν είναι ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, αλλά είναι ένα είδους προϋπόθεση, αναγκαία προϋπόθεση. Και αυτό το οποίο έχουμε υπόψη είναι η αναγνώριση ή η αναφορά τεχνικών προδιαγραφών και τεχνικών χαρακτηριστικών στον τομέα αυτό θα πρέπει να γίνονται και να απαριθμούνται μόνο όταν καλύπτουν το μίσο όπου ε, ε, τα όργανα τυποποίησης δεν δραστηριοποιούνται ή όπου οι προδιαγραφές και τα πρότυπα έχουν καταστεί ανεδαφικά ή ανεδαφικές και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ε, μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ώστε να μπορεί να καλυφθεί το κενό. Έτσι καθορίζουμε την περίπτωση αναφοράς αυτών των στοιχείων, των τεχνικών αυτών προδιαγραφών ή χαρακτηριστικών στο ICT. Αφ' αυτού δεν είναι λοιπόν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο αυτό. Αν θα θέλαμε να απαριθμιστεί Ίσως θα υπήρχαν κάποιες περιπλοκές. Η ιδέα δεν είναι να αλλάξει εκ βάθρων μια υφιστάμενη διάταξη και οι, δια... κανονισμοί για το ICT όπως ισχύουν στο... στην αγορά δεν θα μπορούσε να είναι στόχος της Επιτροπής ή κανένας άλλου να τροποποιήσει, να αλλοιώσει αυτές τις ε, διατάξεις και ρυθμίσεις ICT. Οι άλλες τροπολογίες αφορούν την ανάγκη να καθοριστούν οι διαδικασίες νομιμοποίησης και πάλι εδώ πιστεύουμε ότι κάποιο λάθος μπορεί να έχει παρισφρήσει. Διότι εδώ γίνεται λόγος και για έγκριση και αυτοί, αυτές οι έννοιες είναι ε, σκόπιμες και θετικές όταν αφορούν τις βέλτιστες προδιαγραφές ε, για τέτοια θέματα. Εδώ δεν κάνουμε όμως λόγο για τη δημιουργία νέων προτύπων και προδιαγραφών, αλλά κάνουμε μόνο λόγο για το να επιτραπεί η χρήση ήδη υφιστάμενων διατάξεων για τις δημόσιες προμήθειες και αγορές. Όλες αυτές λοιπόν οι διεργασίες θα ήταν ο έλεγχος της συμβατότητας και της πληρότητας πληροφοριών σε σχέση με αυτές τις απαιτήσει. Και αυτό για τους ε, πολυμερείς εμπλεκόμενους σε ένα πολυμερές πλαίσιο για τις πλατφόρμες ICT. Αυτό θα ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο αν θα το επιτρέπαμε θα δημιουργούσε κάποιες ε, κάποια σύγχυση για την αναγνώριση ή την αναφορά σε τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά όσον αφορά το ICT. Ας επαρκεστώ σε αυτά τα σχόλια. Υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Όμως ευελπιστώ ότι όλες οι προσπάθειες μπορούν να συνεισφέρουν ώστε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό και έτσι να μπορέσουμε να εγκρίνουμε το δυνατόν ταχύτερα αυτή τη στρατηγική σημασία και προσέγγιση πρόταση. Και στο τέλος τέλος ελπίζω ότι θα καταλήξουμε με ένα καλό κανονισμό, θετικό κανονισμό, που δεν θα χαμηλώσει, δεν θα μειώσει το επίπεδο φιλοδοξιών μας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι από χρονική απόψεω καλά τα πηγαίνουμε. Θέλετε, κυρία, Κόμη, να συνοψίσετε τη συζήτηση. Ναι, σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το φόρουμ και την πλατφόρμα, επαναλαμβάνω ότι δεν βλέπω τη χρησιμότητα να βάλουμε εντός του κανονισμού το φόρουμ που μπορεί να δημιουργηθεί σε ιδιωτικό πλαίσιο. Δεν βλέπω να υπάρχει αντίθεση όσον αφορά τα φόρουμ και τις πλατφόρμες, αλλά δεν βλέπω κατά πόσο είναι χρήσιμο να ενταχθούν στο κείμενο του κανονισμού. Αυτή είναι η διαφορά. Και θα ήθελα να αφήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ελευθερία να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα γίνει η διαβούλευση. Διότι εμεί αντικειμενικά υποχρεώμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε διαβούλευση όσον αφορά τον τρόπο που προτιμάει όμω να την αφήσουμε να κάνει, ε, να το διαμορφώσει, να τον διαθρώσει αυτό το διάλογο. Ε, θέλουμε να βαθύνουμε σε αυτό και είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε τελική συμφωνία, συμβιβασμό όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Πράγματι θα ήταν καλύτερο να απλουστευθεί από τώρα. Δεδομένου όμω ότι περνάμε από οδηγία σε κανονισμό, ίσω είναι καλύτερο να αφήσουμε μεγαλύτερη ακαμψία σε αυτή την πρώτη φάση και να απλουστεύσουμε σε μερικά χρόνια. Διότι πρέπει να βρούμε μια διάρθρωση και καλύτερη ενίσχυση τη εθνική πτυχή και αυτό είναι ο στόχο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και για τη χρηματοδότηση και για την απλούστευση όσον αφορά την είσοδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μετά να πετύχουμε έτσι ενίσχυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίθετα στι υπηρεσίε, στο πεδίο τη εφαρμογή, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ρητά ότι τα το πρότυπα δεν πρέπει να δημιουργείται σε κάποιου τομεί που δίνει αρμοδιότητα τη Ένωση. Γι' αυτό το λόγο εγώ ίδια πιστεύω ότι κάποιοι σε κάποιους τομείς τα πρότυπα μπορούν να είναι πιο προβληματικά από ό,τι για άλλους τομείς, αλλά ήθελα να δημιουργήσω μια γενική γραμμή. Δηλαδή, μια πτυχή κατευθυντηρίων γραμμών για να καθορίσουμε αργότερα ποιοι τομείς θα μπουν ή ποιοι όχι. Δεν ήθελα να πω επακριβώς υπέρ ποιων τομέων είμαι υπέρ και υπέρ είμαι κατά, για ποιους τομείς είμαι κατά, διότι θα ανοίγαμε ε, προβλήματα και θα δημιουργούσαμε ε, σφάλματα, εξαιρώντας και συμπεριλαμβάνοντας κάποιες τομείς. Ήθελα κατευθείαν γραμμή. Τώρα για τη ε, γλώσσα, αυτό θα το δούμε στην πράξη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κλείνοντας τη σημασία που έχουν οι... τα άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με τους εργαζομένους, τους καταναλωτές, με τα συνδικάτα, με τους περιβαλλοντολόγους αλλά εγώ θα έλεγα ότι τα πρότυπα που αναφέρονται στους ανθρώπους με αναπηρία είναι μία από τις προτεραιότητες που θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Είμαι ικανοποιημένη που παρέμεινε εντό του χρονικού περιθωρίου. Ευχαριστώ όλου τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους και θα τα ξαναπούμε στη συζήτηση για τις συμβαστικές ε, λύσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. I think we have to move on. Μάλιστα, ωραία. Να συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Την οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία. Η συγγήτριά, η συγγήτριά μας, η Μπερναντέτ Φερνιό, που είναι και αντιπρόεδρος, θα μας κάνει μια εισαγωγή. Madame la Présidente. Euh, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous, nous commençons Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για ένα ζήτημα το οποίο βέβαια είναι θεμελιώδου σημασίας και για την ε, εσωτερική αγορά, αλλά και για την ευημερία και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών μας με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια είτε για τους επαγγελματίες, είτε για τους χρήστες, τους ασθενείς, τους καταναλωτές. Θα ήθελα καταρχάς μία ακόμη φορά να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βλέπω ότι είναι παρούσα εδώ με πολλούς εκπροσώπους. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω γιατί εδώ και πολλούς μήνες έχουν εργαστεί πολύ σκληρά και κυρίως σε πάρα πολύ καλό πνεύμα διαλόγου μεταξύ των δύο οργάνων μας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και οι πολίτες μας ε, χρειάζεται να γνωρίζουν ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι πάντοτε υποχρεωτικά κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποχρεωτικά κατά των πολιτών. Νομίζω ότι όταν εφιώς εργαζόμαστε μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα εφιές κείμενο. Έχουμε τέλος πάντων ήδη μια καλή δομή. Και νομίζω ότι σε αυτό το πνεύμα ε, θέλουμε όλοι να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα είναι και ποιοτικό αλλά και πιο εύληπτο για τους ε, ε, πολίτες. Και αυτό που θέλουμε όλοι και που είναι στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και παρά τις ανησυχίες που είχαμε, Υπήρξαν κάποιες ανησυχίες για την αναλογικότητα, την επικουρικότητα. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία δεν αντίκειται σε αυτές τις δύο αρχές, αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Είναι προφανές ότι όσο προχωρούσαν οι διαπραγματεύσεις, ε, ότι σε γενικές γραμμές έχει τύχει καλής αποδοχής, ε, υπήρχαν όμως, ε, υπάρχουν όμως ακόμη κάποια ερωτήματα και γι' αυτό ζήτησα να ε, έχουμε τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων με όλους τους ενδιαφερομένους. Το χρονοδιάγραμμα ήταν ε, λίγο εκτεταμένο, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, πολλές ιδιαιτερότητες για να εξασφαλίσουμε καλύτερα την ασφάλεια των επαγγελματιών, των ασθενών και των καταναλωτών και είναι ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και δικός μας ρόλος ως συνομοθέτη να λάβουμε υπόψη ε, του τι είναι, το τι είναι σημαντικότερο για την ανάπτυξη ε, της εσωτερικής αγοράς και, επίσης, και από την άλλη να μην πλήξουμε τους πολίτες, να μην τους δημιουργήσουμε φόβους. Θα ήθελα, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, δεν θα ήθελα να συζητήσουμε και πάλι το ανοιχτό πνεύμα της συγκεκριμένης ε, πρότασης ε, και την ε, προσπάθεια εναρμόνισης των επαγγελματικών προσόντων και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπερβούμε τις αδυναμίες που υπάρχουν ε, στην υφιστάμενη οδηγία, γιατί ακριβώς δεν είχαμε το χρόνο, ε, ούτε τοποθετήσαμε σωστά τα πράγματα ε, στο πλαίσιο ενός οράματος για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το μέλλον των πολιτών σε 20-30 χρόνια. Είναι ένα κείμενο πολύ σημαντικό και νομίζω ότι η οδηγία του 2005 δεν τα κατάφερε πολύ καλά. Δεν θα ήθελα λοιπόν ε, να παραδοθούμε σε διάφορες τάσεις ε, συγκεκριμένων κατηγοριών ε, και προστατευτισμού μπορώ να σας πω. Είμαστε άλλωστε και σε περίοδο κρίσης και έχουμε τέτοιου είδους αντανακλαστικά μερικές φορές. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω μια πρώτη εικόνα αρχίζοντας το διάλογο. Πρώτον, η αντικατάσταση των κοινών ε, ε, πλατφορμών από το άρθρο 49α, όπως επίσης και του ε, πλαισίου ευρωπαϊκής κατάρτισης. Αυτά έχουν τύχει καλής αποδοχής και αυτό είναι πολύ καλό νέο, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα. Πρέπει λοιπόν να επιβεβαιώσουμε και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι θα υπάρχει πλήρη εκπροσώπηση των ε, αρμοδίων ε, και ακαδημαϊκών αρχών, όπως επίσης και παρακολούθηση πάρα πολύ τακτική της ε, του, σωστού επίπεδου. Μερικές φορές έχουμε μια σοβαρή ανησυχία ε, όσον αφορά την προσφυγή στις κατεξουδότες πράξεις. από ό,τι κατάλαβα από τις πρώτες διαβουλεύσεις που είχα, θα πρέπει πραγματικά να ε, έχουμε μέσα διαφανή, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στο κείμενο. Επίσης, η μερική πρόσβαση, αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους, ε, γιατί παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται σε αποφάσεις του δικαστηρίου, είναι πηγή πολλών φόβων και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε εδώ ένα, ε, μια όσο δυνατόν μεγαλύτερη πλαισίωση αυτής της πρόσβασης. Όσον αφορά τώρα τα ε, ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και αναφέρομαι κυρίως ε, στα σημεία που ανησυχούν τους επαγγελματίε, για τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη, ένας μεγάλος φόβος ανοίγματο, άρθρο 59 και απορρίθμισης. Ε, νομίζω το συζήτησα και με τις υπηρεσίε Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμφωνούν αν κατάλαβα καλά με τις δικές μας ανησυχίες. Δεν θέλουμε να υπερνομοθετήσουμε ε, τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και αναφέρομαι κυρίως ε, στους... Ε, ε μηχανικούς, γιατί μερικές φορές ζητούν μία εξαίρεση όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των ε, ε, συμβολεογράφων, που είναι επίσης ένα κλειστό επάγγελμα. Είχαμε επίσης ε, πολλά ζητήματα τα οποία είχαν προκύψει και στην υπηρεσία για, την οδηγία για τις υπηρεσίες και μπορεί να επανέλθουν και εδώ. Υπάρχει μια σύγχυση εντός ορισμένων επαγγελματικών κλάδων. Μόλις διάβασα ένα κείμενο το οποίο Ήρθα από τη Γαλλία, δεν θα σας κάνει εντύπωση, τεράστια σύγχυση σε σχέση με το κείμενο που έχουμε μπροστά μας μεταξύ της αρχής ε, της ε, ε, χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής και τις τεράστιες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν και παρεμβολές. Τέλος πάντων υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να εξηγήσουμε και θα είναι και καθήκον μας. Δεν Τώρα όσον αφορά αυτή την επαγγελματική ε, κάρτα που βασίζεται σε ένα σύστημα πολύ πιο εξελιγμένο, πιο ε, εκλεπτισμένο. Τέσσερα-πέντε χρόνια, ήταν, πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια το συζητήσαμε πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο. Προχωράμε σιγά-σιγά και όσο προχωράμε οι επαγγελματίες θεωρούν ότι αυτή η ιδέα είναι καλή. Χαιρόμαστε βέβαια, αλλά από την άλλη παραμένουν ερωτήματα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς επί των πέντε σημείων που πρέπει να συμπεριλάβουμε ε, στο συγκεκριμένο αυτό θέμα την αξιοπιστία, την διεξοδικότητα, ε, τα προσωπικά δεδομένα ε, που προστατεύονται ε, και βεβαίως την προαιρετική πτυχία. Εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ κατηγορηματικοί γιατί υπάρχουν φόβοι και ερωτηματικά που δεν είναι και πολύ ευπρόσδεκτα. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα αντιστάθμισης και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτά τα μέτρα πρέπει να παραμένουν δυνατά στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας και αυτό κυρίως για τα ιατρικά επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων βέβαια ε, των ζητημάτων γλωσσικής κατάρτισης. Ε, το συζητήσαμε και με την Επιτροπή. Εγώ δεν συμφωνώ πάρα πολύ με την ιδέα ε, οι γλωσσικές ε, δεξιότητες να αξιολογούνται από ε, βέβαια, οι περισσότεροι επαγγελματίες ε, συμφωνούσαν ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο από αρμόδιες ε, αρχές επαγγελματιών και, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι πολύ σοβαρά ζητήματα ετέθησαν ως προς αυτό το θέμα. Καλό θα ήταν να σταματήσω κάπου εδώ Γιατί αυτά είναι τα ζητήματα που δημιουργούν τα περισσότερα ερωτήματα και θα ήθελα να τα συζητήσουμε γιατί έχω πολλά ακόμη να πω, αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο και στους σκιώδεις εισηγητές γιατί για το θέμα αυτό που μπορεί, για το οποίο μπορούμε να καταλήξουμε σε πολύ ισχυρό συμβιβασμό παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διστάμενες απόψεις εγώ βασίζομαι στην ε, αλληλοκατανόηση, στο διάλογο με τους επαγγελματίες και με όλες τις ομάδες του Κοινοβουλίου και με τις υπηρεσίες της Επιτροπής βεβαίως και με το Συμβούλιο. Γιατί και το Συμβούλιο είναι εδώ, από ό,τι βλέπω. Το λέω αυτό γιατί την τελευταία φορά είχα θέσει ερωτήματα στην Δανική Προεδρία και δεν μου είχε απαντήσει κανείς. Από ό,τι ξέρω θα έχετε συναντήσει στο Μάρτιο για το θέμα αυτό. Υπάρχει ένα επίπεδο εναρμόνισης για την κατάρτιση. Αυτό είναι πραγματικά ζήτημα κλειδί. Και είναι και το ζήτημα το οποίο Γνωρίζω ότι θα δημιουργήσει πολλές δυσκολίες ε, μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο, γιατί ο καθένας θα θέλει να ε, υπερασπιστεί τα προνόμια του και τη δική του κατάρτιση. Και το, δίσκο, το επίπεδο εναρμόνισης θα είναι δύσκολο. Είναι όμως ένα ζήτημα κλειδί και βασίζομαι στο Συμβούλιο ότι θα προχωρήσουμε επιτέλους ε, και μάλιστα εις βάθος ως προς το θέμα αυτό. Να πάρουν τώρα το λόγο και οι συνάδελφοί μου. Είμαστε σε μια φάση διαβούλευσης. Ε, θα έχουμε συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητής, θα κάνουμε και ακρόαση. Για την ώρα βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς το πλαίσιο και τα θέματα. Μια ακρόαση 24-25 Απριλίου. Θα προσκαλέσουμε και τους επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες για ε, θέματα τα οποία είναι προβληματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρχεται η συζήτηση, μάλλον μίλησα και πολύ. Οπότε έχουν το λόγο οι συνάδελφοί μου. Κυρία Πρόεδρε. Yes, thank you. Ευχαριστώ. Κυρία Φερνιού. Πράγματι ήρθε η ώρα να δώσουμε το λόγο στους Κιώδης. Χαίρομαι που βλέπω ότι οι περισσότεροι σκιώδεις εισηγητές είναι παρόντες. Και ίσως καταφθάνουν και άλλοι, δύο από αυτούς. Πρώτα απ' όλα, Κώστας Λεκρή από το ΕΛΚ. Και εγώ, Πρόεδρε, χαίρομαι που ανταλλάσσουμε απόψεις επί σημαντικότητα του κειμένου. Μερικές εβδομάδες μετά την παρουσίαση τον περασμένο Δεκέμβριο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της προτάσεως της οδηγίας, αναθρημένης προτάσης οδηγίας. Και θα ήθελα στην αυγή αυτού του δρόμου του κοινοβουλευτικού να πω κάποια βασικά λόγια. Η βελτίωση τη διαδικασία αναγνώριση των προσόντων, επαγγελματικών προσόντων, είναι ο στόχο τη οδηγία αναθεωρημένης και εντοπίζεται από τον Επίτροπο Μπαρνιέ σαν ένα από του 12 μοχλού ανάπτυξη. Ότι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναβρει το δρόμο τη ανάπτυξη και τη ευμάρεια. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε λοιπόν αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία, ούτε το ότι η ουσία του αναθεωρημένου κειμένου είναι μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη απλούστευση, μεγαλύτερη κινητικότητα, με μια κουβέντα να ξεκινήσει η δημιουργία πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Euh, euh, euh, Όπως έλεγε και η Μπερναντέτ Βερνιό, Έχουμε συναντήσει πολλούς επαγγελματίες, έχουμε έρθει σε επαφή με πολλές οργανώσεις, οργανισμούς ενώσεις και έχουμε ακούσει τις απόψεις όλων εκείνων ε, που ενδιαφέρονται για το θέμα. Όλων των φορέων. Των Ευρωπαίων συμπολιτών μας τις απόψεις. Που πρέπει να ζήσουν στα πλαίσια ενό νέου συστήματος αναγνωρίσεως επαγγελματικών δεξιοτήτων και προσόντων. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι τελικές θέσεις που θα υιοθετηθούν από την ε, ομάδα του ΕΛ και ονόματι του οποίου δεν θέλω να σήμερα. Εκφράζω κάποιε ανησυχίε όμω κάποιε παρατηρήσει. Να μοιραστώ κάποια σχόλια. Ξέροντα ότι οι συζητήσει και εντό του ΕΛΚ ξεκίνησαν ήδη και είναι αρκετά ζωηρέ όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αυτή Κάρτα των ε, Γερματικών Προσόντων. Ε, θα έχουμε και στην προηγούμενη θητή έχει τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το σημαντικότερο εργαλείο, συγκεκριμένο εργαλείο τη Ευρώπη των Πολιτών όμως οι επαγγελματίες με τους οποίους συναντηθήκαμε ε, έχουν κάποιες παρατηρήσεις, κάποια σχόλια να κάνουν, κυρίως όσον αφορά το θέμα των χρονικών ορίων που έχουν ε, προβλεφτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση του αναθεωρήσεως της οδηγίας, φαίνεται να δημιουργούν κάποιο προβληματισμό. Και ίσως θα μπορούσαν να προσαρμόσουμε κάπως τα χρονικά περιθώρια. Από ό,τι ακούμε στου επαγγελματίε, θεωρούν ότι 15 μέρε σε κάποιε περιπτώσει, ένα-δύο μήνε σε κάποιε άλλε περιπτώσει, θεωρούνται αρκετά σύντομα χρονικά διαστήματα. Υπάρχει και ένα θέμα που δημιουργεί ανησυχίε. Δηλαδή η χώρα υποδοχής δεν έχει τόσο πολύ δυνατότητα απόφασης και ελέγχου όσον αφορά τη χορήγηση επαγγελματική κάρτας. Δεν θέλουμε να ξαναδημιουργήσουμε περίπλοκα συστήματα και επαχθή και περιοριστικά που μας οδηγούν σε απώλεια χρόνου, όμως θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι κάποιοι ενδιαφερόμενοι ε, θέλουν να μπορέσουν να διατηρήσουν ένα είδους επίσημης εξακρίβωσης που θα διεξάγεται από τη χώρα υποδοχής. Και εκεί, όπω μα είπε η κυρία Βερνιό, πιστεύω ότι μπορούμε στο κείμενο το παρόν, όπω μα υπευλήθη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να διευκρινίσουμε ακριβώ τον εκούσιο χαρακτήρα τη επαγγελματική χάρτας, κάρτας, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Όσον αφορά την μερική πρόσβαση, γιατί να κρυβόμαστε, υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες, ε, να μην πω ότι κάποιοι επαγγελματίε εξέφρασαν και εχθρότητα ε, για αυτή τη μερική πρόσβαση. Και στην έκθεση Μακλάρκιν εμεί είχαμε εκφράσει κάποιες επιφυλάξεις και θέλαμε αυτή η αρχή να εφαρμόζεται κατά περίπτωση στα πλαίσια των επαγγελμάτων όπου μπορεί να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα όρια και θέλαμε να υπάρχει ε, όσον αφορά τα εθιζόμενα επαγγέλματα κάποια προσοχή να δοθεί όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας, υγείας κλπ. για τη μερική πρόσβαση. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω σήμερα αυτή, την ευχή που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την πλαισίωση και τον ακριβή ορισμό του τι εννοούμε όσον αφορά τη μερική πρόσβαση, όσον αφορά την αναγνώριση των, γλωσσικών γνώσεων, χρειάζεται απλούστευση Θέλουμε να εξασφαλίζουμε μεγαλύτερη ασφάλεια κλπ. Αλλά μέσω αυτού δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ξανά ένα περίπλοκο σύστημα και να δημιουργήσουμε εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία με το πρόσχημα της επαλήθευσης και εκ νέου επαλήθευσης ξανά επαλήθευσης των γλωσσικών δεξιοτήτων. Υπάρχει αντικειμενόμενο. θέλουμε ευελιξία που θα χορηγεί τις αρμόδιες αρχές για να δούμε κατά πόσο είναι σκόπιμο να γίνει κάτι τέτοιο και πώς εξασφαλίζουν τα γλωσσικά τεστ. Και έχει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα Εθνικό Σύστημα ε, Περίθαλψης Υγείας. Αυτός ο όρος, αυτή η ονομασία δεν ξέρω τι καλύπτει. Όσον αφορά την επαλήθευση των γλωσσικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, και εδώ χρειάζεται διευκρίνηση. Όσον αφορά το ρόλο των διαφόρων αρμοδίων αρχών των εθνικών συστημάτων υγείας ενώσεων ασθενών. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να παρεμβαίνουν εν πρώτη θα θεωρούν σκόπιμο όσον αφορά την επαλήθευση των ε, ε, γλωσσικών ε, δεξιοτήτων. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε και σε άλλες ανταλλαγές απόψεων επί των διαφόρων θεμάτων στα ιατρικά επαγγέλματα θέλουν η αρχική διάρκεια της κατάρτισης να εκφράζεται όχι μόνο σε χρόνια αλλά και σωρευτικά σε ώρες είναι μια διεκδίκηση που θα μπορούσε να εισακουστεί. Η δημιουργία κοινών πλαισίων κατάρτισης, άρθρο 49α, αυτό είναι κάτι που το χαιρετίζουμε, ένα βήμα προόδου σημαντικό. Ίσως ε, θα ήταν καλό να δούμε τι όρους θα βάλουμε για την πιστοποίηση μιας δημιουργίας με την ε, αξιολόγηση συστήματος κατάρτισης από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους που χορηγεί την, ε, το πιστοποιητικό για να έχουμε τα αναγκαία αχέγγυα. Δεν διατείνομαι ότι υπήρξε εξαντλητική. Θα ήθελα να αναφέρω ακροθυγός δύο επαγγέλματα που δεν ακούγονται πολύ. Ε, ε, η κυρία Βερνιό αναφέρθηκε σε βολογράφους που είχαν εξαιρεθεί από την οδηγία που εξακολουθεί να ισχύει και θα ήθελαν να εξακολουθούν να εξαιρούνται το πεδίο εφαρμογή τη αναθωρημένη οδηγία. Πρέπει να εξετάσουμε μεγάλη προσοχή μια ιδιαίτερη κατάσταση. Άκουσα τα διάφορα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν συμβολογράφοι διαφόρων κρατών μελών και έχω υπόψη μου την κατάσταση ενός άλλου επαγγελματό, πολύ αξιοπρεπούς των νοσοκόμων, ανδρών και γυναικών. και σήμερα και στο μέλλον πρέπει να καλύψουμε κάποια μεγάλα κένα αυτόν, αυτού του τομέα των νοσοκόμων. Χρειάζεται να βελτιωθεί η κινητικότητα αυτών των επαγγελματιών. Όμως η αύξηση του, ε, των πληροφοριών πρέπει να χορηγούνται δημιουργεί προβλήματα σε κάποιες χώρες και τις προθεσμίες κατάρτισης επίσης δημιουργεί κάποια προβλήματα. Πρέπει να ακούσουμε τι λένε και οι επαγγελματίες και οι διάφορες χώρες που έχουν διαδικασίες κατάρτισης ε, ιδιαίτερες. Αυτά κλείνοντας για να δημιουργήσουμε την πραγματική αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή έχουμε πολύ δρόμο να τραβήξουμε ακόμα. Ξεκινά λοιπόν όμως ε, μια νομοθετική δουλειά που θα, τελικά θα οδηγήσει στο να κάνουμε κάποια σημαντικά βήματα πρόοδο. Αυτά και ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στη γενική προσέγγιση που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εξυγχρονισμό του νομικού πλαισίου σε σχέση με τα επαγγελματικά προσόντα, βλέπω πολύ ισορροπημένη προσέγγιση. Αυτά που έχουμε στο τραπέζι είναι σαφή και καλά ως αφετηρία, ως γραμμή αφετηρίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη αρκετά σημεία που εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο εμείς αναφέραμε και εξετάσαμε στις πρώτες συζητήσεις που είχαμε στην περίοδο εκείνη που εμείς συζητούσαμε το ίδιο θέμα αναμέταξύ μας. Επίσης πιστεύω και κάτι άλλο, ότι το εύρος, ε, η, παράταση, η επέκταση του ε, εύρους του φάσματος δεν είναι κάτι το θετικό. Υπάρχουν κάποιες ε, εξειδικευμένες ανάγκες και χαρακτηριστικά αυτών των επαγγελμάτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο φυσικά είπε ότι εδώ δεν πρόκειται πάντα για θέμα δημόσιας αρχής. Όμως, σε σχέση με κάποιες δραστηριότητες ε, που ε, εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο και κάποιες άλλες ε, που απαιτούν διαδικασίες από τα κράτη-μέλη, είναι μέρος πολλές φορές του ιδίου επαγγέλματος και έτσι δυσχεραίνεται η διαφοροποίηση στις ιδιαιτερότητες. Δεν ξέρω σε σχέση με τους συμβολεογράφους αν αυτό βοηθά τα πράγματα πράγματι. Έχω αμφιβολίες σε σχέση με τους συμβολεογράφους το να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε ένα άλλο κράτος μέλος όταν μόνο περιορισμένες δραστηριότητες μπορούν να ακολουθήσουν. Όπως η κυρία Βερνιό και όπως η κυρία Λεγκρίπ, έτσι και εγώ, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο περισσότερο σε βάθος αυτό το θέμα. Υποστηρίζω την ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα επαγγελματικό τέτοιο ε, διοντολογικό ας το πω έτσι, πλαίσιο και θα πρέπει έτσι να ξεκινήσουμε την δική μας παρέμβαση προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Κάπως ε, ανησυχώ όσον αφορά την ιδέα της πιστοποίησης αυτής της κάρτας ιδερτίου ε, όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα από κάποιο κράτος. Έχω ήδη, έχουμε κάποια μηνύματα από κράτη-μέλη ότι είναι πολύ πιεστικές οι προθεσμίες και για να υπάρξει εμπιστοσύνη που θέλουμε να εμπνέει το σύστημα πρέπει να λάβουμε νομίζω υπόψη όλες τις εναλλακτικέ λύσεις για να καταλήξουμε στο τέλος τέλος ε, με κάποια λύση την οποία θα συμφωνήσουν όλοι με μια ιδέα που θα εμπνέει το σύστημα αυτό και θα είναι πιο αποτελεσματικό για την προστασία των καταναλωτών και των ασθενών θα έλεγα σε σχέση με την σιωπηρή ε, πιστοποίηση ή έγκριση αυτής της κάρτας ακόμα και αν υπάρχουν ε, οι δυνατότητες του να γίνουν σεβαστές οι προθεσμίες πρέπει να βρούμε δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων. Για την διάρκεια αυτής της ε, κάρτας ιδερτίου προτείνονται δύο έτη ενώ είχαν προταθεί αρχικά, είχε προταθεί ένα έτος. Πρέπει να δούμε εκ του σύνεγγυς περισσότερο τα πράγματα. Μετά από τα πρώτα δύο χρόνια θα πρέπει να ανανεώνεται αυτή η άδεια ή δελτίο σε μια ετήσια βάση έτσι όπως λέγουν. Δεν κατανοώ τον λόγο αυτό. Γι' αυτό σε σχέση με την επιλογή του Συμβουλίου για μία μονοετή περίοδο για τους άλλους μηχανισμούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προτείνονται υποστηρίζονται όπως ε, θα πρέπει να εντάσσονται στην τρέχουσα ενισχύ νομοθεσία και να προβλέπεται η καλύτερη προστασία των καταναλωτών ή των ασθενών. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις εξειδικευμένες λεπτομέρειες, να εξετάσουμε για παράδειγμα την ε, ενεργοποίηση του μηχανισμού προειδοποίησης ή συναγερμού με μια δυνατότητα να δούμε ένα ολόκληρο εύρος γεγονότων ή συμβάντων που θα μπορούσαν να, αναφέρονται στις πρακτικές εφαρμογές. Για τις γλωσσικές δεξιότητες ή ικανότητες πρέπει να διασφαλίσουμε για το προσωπικό περίθαρψης... και παροχής υπηρεσιών στον υγειονομικό τομέα να υπάρχει η πρόβλεψη για μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας υποδοχής. Όμως Πιστεύω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αποσαφήνιση αυτού του άρθρου, επιμερισμός αρμοδιοτήτων με σαφήνεια διότι δεν θέλουμε αυτές οι γλωσσικές δοκιμασίες στο τέλος τέλος να χρησιμοποιηθούν ως πρόσκομα στην κινητικότητα. Ας καταστήσουμε σαφέστερο αυτό το πλαίσιο, να μην υπάρχει δυνατότητα να αυτό να χρησιμοποιείται ως άλοθη, ως φραγμός για την κινητικότητα των εργαζομένων. Για τις γλωσσικές ικανότητες και δοκιμασίες ένα ευρύτερο πλαίσιο πρέπει να εντάσσονται αυτές. Γλωσσικές ικανότητες για να μπορεί κάποιος να περνά μια συνέντευξη, όχι κλασικού τύπου εξετάσεις γλωσσικές. Ολοκληρώνω με μια παρατήρηση για την εισαγωγή, την προσέγγιση των ε, αναγκαίων προσόντων και δεξιότητας ε, μαζί με τις ε, προδιαγραφές ε, κατάρτισης ε, και εκπαίδευσης. Δεν μπορούν όλα να γίνουν και να ρυθμίζονται μέσα σε μια τέτοια οδηγία. Είναι όμως θεμελιώδους χαρακτήρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμπλακεί σε διαβουλεύσεις με τους επαγγελματικά εμπλεκόμενους και τις αρμόδιες αρχές προτού συνταχθούν οι κατεντολήν πράξεις, οι εντεταλμένες πράξεις. Και σε διάλογο με θυμόν έλαβαν υπόψη πολλές από τις παρατηρήσεις μας τότε. Είμαι βέβαιος και ευελπιστώ ότι η ίδια προσέγγιση θα υιοθετηθεί όταν θα έρθει η ώρα της έγκρισης τέτοιων κατεντολήν πράξεων. Ευχαριστώ. Thank you very ευχαριστώ πολύ. Η Εμίλη Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω δανέζικα λοιπόν. ja, jeg er enig ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έγιναν από ε, πλευρά συγγήτριας ότι είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό σε σχέση με την πρόταση αυτής της οδηγίας και την αναδιατύπωση για την διοικητική συνεργασία που θα πρέπει να εμβαθυνθεί ιδιαίτερα σε ηλεκτρονικό επίπεδο, ηλεκτρονικά και να υπάρχει και μια δυνατότητα διαιτησίας ο πολιτικός στόχος βρίσκεται, πιστεύουμε, στην ισόρροπη σχέση, ισορροπημένη σχέση μεταξύ ασφάλειας καταναλωτών και ασφάλειας ασθενών και των επαγγελματικών προσόντων και κατάρτισης των επαγγελμάτων σε αυτές τις υπηρεσίες. Θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει περιοριστικό αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και τα θέματα κινητικότητας και ελεύθερης κυκλοφορίας Όλα αυτά πρέπει με ισορροπημένο τρόπο να λαμβάνονται υπόψη και πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη πρόταση. Σε πολλές επαγγελματικές ομάδες και οι ίδιοι οι επαγγελματίες θεωρούν ότι όταν ξεπερνάμε κάποια ε, όρια ε, κάποια σύνορα από μια χώρα σε άλλη μπορεί κανείς να μάθει πολλά πράγματα. Οι εξελίξεις οι επαγγελματικές πρέπει να είναι κάτι με το οποίο θα εξοικειώνονται και θα ενημερώνονται πάντα οι επαγγελματίες. Σε σχέση πάντα και με την αγορά εργασίας, επάγγελμα, επαγγελματική κατάρτιση που πολλές φορές θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα όταν υπάρχουν επικαλύψεις να έχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο εναρμονισμού των προσόντων αυτών τα πράγματα δυσχεραίνονται όταν περιπλέκονται τα πράγματα. Πρέπει οι επαγγελματικές αυτές ομάδες να εντάσσονται στο μεγαλύτερο βαθμό στις ανάγκες που υπάρχουν. Κάποιες, ε, κάποιες χώρες ή κάποια επαγγέλματα ε, βρίσκονται σε μεγάλη, ας το πω έτσι, σε ιδιαίτερη, ε, ιδιαίτερα προνομιούχα θέση ως πρωτοπόροι στην επαγγελματική τους κατάρτιση. Είναι σημαντικό να έχουν και περιόδους που θα εργάζονται στο εξωτερικό. Εφόσον ακολουθείται μια τέτοια πολιτική μπορούν να φτάσουν μακριά αυτοί οι επαγγελματίες. Δεν μπορούμε όμως να επιβάλλουμε έναν εναρμονισμό σε κάποιους ή κάποιες ε, χώρες που έχουν πολιετής παραδόσεις. Νομίζω μπορούν να έχουν, μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα με τέτοιες πρωτοβουλίες. Σημαντικό είναι με τις επαγγελματικές ομάδες και ενώσεις να συνεργαζόμαστε ώστε εκείνη να είναι η κινητήρια μηχανή, ο κινητήριος, ε, η κινητήρια δύναμη και όχι εμείς. Και σε σχέση με την δυνατότητα πρόσβασης ε, δεν βρήκα κανέναν ακόμα που να ε, είναι ικανοποιημένος με τις προτάσεις ε, και τα πρότυπα αυτά. Έχουμε αρχίσει αυτό το έργο ε, εδώ και κάποιο καιρό και ακούω πάντα, ενημερώνομαι ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Ναι, μεν πρέπει να αναγνωρίζονται κάποια πράγματα, αλλά να λαμβάνουμε υπόψη και την χειροπιαστή πραγματικότητα σε κάποιες χώρες και τομείς. Ας πάρουμε υπόψη τώρα μία νοσοκόμο ή ένα νοσοκόμο που εργάζεται σε αυτό το επάγγελμα και διασυνοριακά πώς μπορεί κανείς να λάβει ως σημείο αναφοράς το θέμα της αιμοληψίας ή όχι. Νομίζω στην πρακτική εφαρμογή στα ίδια τα νοσοκομεία και τις κλινικές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχουν και άλλες διαφοροποιήσεις που πρέπει να τις δούμε πάντα διαφοροποιημένα και προσπαθώντας να επιλύσουμε τις διαφορές. Μια τελευταία παρατήρηση για τους ε, ε, νέους. Η ανεργία των νέων είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα και λόγω κρίσης στην Ευρώπη. Αλλά επίσης και επειδή σε κάποιους τομείς υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης προσφοράς από τους εργοδότες. Δεν υπάρχουν λέει τα αναγκαία προσόντα και δεξιότητες από πλευράς των νέων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες εργασίας και εδώ υπάρχει η δυνατότητα στο εξωτερικό να βρει κανείς μια πρώτη εργασία, μια πρώτη θέση απασχόλησης. Θα πρέπει εδώ να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους μπορεί κάτι τέτοιο να επιτευχθεί ώστε να υπάρχουν ξεχωριστά θέσεις εργασίας για νέους, ξεχωριστά για τους νέους, για εκείνους που μπορούν να ταξιδέψουν, να μεταβούν στο εξωτερικό, ώστε να μπορέσουν έτσι να δραστηριοποιηθούν καλύτερα. Απαιτείται λοιπόν μια ισορροπημένη προσέγγιση και οι ομάδες οι επαγγελματικές πρέπει να εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο ισχυρής ενισχυμένης συνεργασίας. Ευχαριστώ. Από την Ενωτική Αριστερά η επόμενη παρέμβαση αλλά δεν βλέπω από πλευρά σκιώδους εισηγητή να παρίσταται κάποιος Γκούσταυσον για παράδειγμα. Υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει δικαίωμα παρέμβασης από την Ενωτική Αριστερά. we... Εντάξει, συνεχίζουμε λοιπόν. Η κυρία Μακλάκιν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως πάντα, Χαίρομαι ιδιαίτερω ε, όταν βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη πολλές από τις προτάσεις ε, και τις απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε, την ενίσχυση της κινητικότητας, ε, όπως επίσης και να μπορούν οι επαγγελματίε με προσόντα να εργάζονται ευκολότερα εντός της ενιαίας αγοράς και να γίνονται επίση και οι έλεγχοι για ανθρώπους που δεν έχουν προσόντα είναι ένα από τα βασικά ωφέλη της ενιαίας αγοράς ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε πρέπει να εργαστούμε ώστε να απομακρυνθούν ε, τα εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται και να αυξήσουμε την κινητικότητα. Εξετάζοντας όμως ε, τα πράγματα, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη ρύθμιση στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και να απομακρύνουμε όλα τα, όλες τις διαδικασίες που μπορούν να δημιουργούν επιπλέον εμπόδια. Όμως ε, πρέπει να το κάνουμε τώρα, σε συνεργασία δηλαδή Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη, γιατί νομίζω ότι έχουμε καθιστορήσει, γιατί μπορεί να χάσουμε το παράθυρο ευκαιρίας που έχουμε αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή λόγω της κρίσεως. Έχω επίσης πολύ σοβαρούς ενδιασμούς ε, για τον κώδικα τον επαγγελματικό, ε, πώς είναι δυνατόν να δουλέψει αυτό για κάθε μεμονωμένο επάγγελμα και όσοι θέλουν να επιλέξουν να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να παραμένει προαιρετικό, ε, να έχουν καλύτερες προτάσεις από αυτές που έχει υποβάλει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε σχέση με τις πρώτες προτάσεις που είδαμε πέρσι στην Πράσινη Βίβλο. Αλλά ε, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μία αξιολόγηση αντικτύπου, ε, μία πλήρης ανάλυση κόστους και ωφέλους και τα επαγγέλματα άλλωστε θα το κάνουν και από μόνα τους αυτό το εθελοντικό πρόγραμμα για να εξασφαλιστεί ότι το να συμμετέχουν θα έχει προστιθέμενη αξία για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα και θα λειτουργεί καλά για αυτά. Και χαίρομαι που έχουν εγκρίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ηλεκτρονικές μας λύσεις για την κάρτα αυτή. Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και τα τέλη ε, για την υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, όσον αφορά την εισαγωγή τελών και όσον αφορά τώρα τα επαγγέλματα για, ε, υγείας, στον τομέα της υγείας, εν πάση περιπτώσει, η βασική μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η ασφάλεια των ασθενών και γι' αυτό πιστεύω ότι ε, γλωσσικός ε, έλεγχος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρέπει να είναι σαφές στο κείμενο ότι οι έλεγχοι αυτοί περιορίζονται μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τον ασθενή και ε, όταν ε, οι επαγγελματίες και οι ρυθμιστές θα πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος και θα κάνουν εκείνη τον έλεγχο. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε στην ικανότητα των ε, εργοδοτών να κάνουν ένα τέτοιο είδους γλωσσικό έλεγχο. Πάντοτε είχαν τη δυνατότητα αυτή σε σχέση με την πρόσληψη ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, όμως είναι λίγο ασαφές στο κείμενο και ίσως θα έπρεπε να είμαστε απολύτως σαφείς στο τι θέλουμε να πούμε για τους ελέγχους αυτούς της γλώσσας. Ε, ο μηχανισμός προειδοποίησης είναι πάρα πολύ σημαντικός για την αύξηση της ασφάλειας των ε, ασθενών, αλλά πρέπει να ξέρουμε πότε θα σταλεί, θα αυτή η προειδοποίηση και τι ανταλλαγή πληροφοριών θα γίνουν και είμαι σίγουρη ότι θα γίνουν και άλλες συζητήσεις ε, επ' αυτού στην Επιτροπή μας. Όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσει, πρέπει να τις ενημερώνουμε αλλά πρέπει επίσης να δίνουμε και κάποιο δυνατότητα ευελιξία σε σχέση με τους γιατρούς και τους οδοντιάτρους θα έπρεπε ε, ειδικότερα σε επίπεδο ας πούμε μεταπτυχιακό να μπορούν να έχουν κάποιο περιθώριο ε, ελιγμών. Δεν χρειάζεται να πρέπει να μένουν στην εκπαίδευση ε, τέτοιου είδου επαγγελματίε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να μπορούν να κινηθούν στο πλαίσιο τη ε, αγορά εργασία και δεν πρέπει να του κρατάμε μακριά από αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια ευελιξία στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση. Και όπω και η συγχύτρια έχω κάποιες ε, επιφυλάξει για τι κατεξοδότηση πράξεις. Θα ήθελα να ενθαρρύνω πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβουλευτεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ειδικότερα όσον αφορά τι ελάχιστε απαιτήσει. Και θα ήθελα επίσης να υποστηρίξω κάθε συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Η μερική πρόσβαση επίσης ετέθηκε από την εισηγήτρια και από την κυρία Τουρούνεν. Δεν είναι κάτι που θέλουν οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί οι επαγγελματίε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην είναι ένα παραθυράκι ε, μπορεί να οδηγήσει κόσμο στην αγορά εργασία συντομότερα, αλλά μπορεί επίση και να αποδυναμώσει την ποιότητα τη ε, υπηρεσία που θα λάβουν ε, οι καταναλωτές, οι ασθενεί, ας πούμε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντα ότι με πολύ χαρά θα συνεργαστώ και πάλι με την κυρία Βερνιό και του υπόλοιπου συζητητέ ε, που συμμετείχαν Ούτως ή άλλω ε, θα διαβουλευτούμε με όλους του επαγγελματίε, το κάναμε ήδη και έχουμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη διάθεσή μας για τις διαβουλεύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να τα καταφέρουμε ε, και να επιτύχουμε τους στόχους μας για να επιφέρουμε και τα απαραίτητα αποτελέσματα για τους επαγγελματίες μας. Ευχαριστώ κύριο Σαλβίνη Λύπη. Οπότε πάμε με κάποιον, να ακούσουμε κάποιον άλλον. Okay, yes. And, uh, and uh, I have on my list Schaldemose, Schaldemose, αυτή τη σειρά θα πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα δανέζικα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλά από αυτά που υπόθηκαν με κάλυψαν. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι υποστηρίζω βασικά την μεγαλύτερη κινητικότητα στην εσωτερική αγορά για το εργατικό δυναμικό. Είναι σημαντική η διευκόλυνση της κινητικότητας, να μπορούν να μετακινούνται οι πολίτες μαζί με τα προσόντα τους. Καταλαβαίνω όμως και πολλές από τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι διάφοροι επαγγελματικοί κύκλοι και οι εργαζόμενοι. Διότι είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί ανησυχούν αυτή την περίοδο της κρίσης και ανησυχούν διότι πιστεύουν ότι ίσως μεγαλύτερη κινητικότητα πιέσει προς τα κάτω τις αμοιβέ, τα εμερομίστια και είναι ίσως πιο δύσκολο να μπει κανείς να, δουλε, να βρει δουλειά αν έρχεται κάποιο από μια άλλη χώρα με χαμηλότερη ε, εκπαίδευση, χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευση και χαμηλότερη αμοιβή και παίρνει τη θέση του άλλου. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό δεν θα συμβεί. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να μην χρειάζεται να φοβηθούν έναν ανταγωνισμό προ τα κάτω των αμοιβών Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι ευκολότερο να χρησιμοποιεί κανείς τις ικανότητες του αλλού. Το σημαντικότερο κατά την άποψή μου είναι να αντιμετωπίσουμε το θέμα της μερικής ε, αναγνώρισης. Υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πράγματι και απαιτείται να κάνουμε κάποια πράγματα. Θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικότερα κατά πόσο θα είναι δυνατόν στην πράξη να χρησιμοποιήσουμε μερική αναγνώριση, σύστημα μερικής αναγνώρισης αν πετύχουμε σωστή λύση εκεί θα ανησυχεί λιγότερο το κοινό για το θέμα της αμοιβέ αναγνώρισης των προσόντων. Βέβαια, αν πάρουμε ένα παράδειγμα, τους νοσοκόμους και τις νοσοκόμες, Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν είναι κανείς νοσοκόμος δεν σημαίνει ότι ε, σε κάθε χώρα όλες οι χώρες έχουν τέτοια προσόντα. Είναι νοσοκόμοι. Ας... Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις στη Γερμανία και στη Δανία. Υπάρχει διαφορά, πρέπει να αναγνωριστεί και να ληφθεί υπόψη. Δεν είναι πρόβλημα. Και να μπορούμε έτσι να αξιολογούμε τις διάφορες δεξιότητες. Υποστηρίζω μεγαλύτερη κινητικότητα μένα, αλλά υπάρχουν και πολλές ανησυχίες ε, που εκφράστηκαν και ίσως δεν θα πρέπει να μπούμε πολύ στην πτυχή της μερικής αναγνώρισης ε, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα καθησυχάσουν πολλές ανησυχίες. Ευχαριστώ. Κέμπερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω είμαι υπέρ της αναδιατύπωσης ε, της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες διότι πιστεύω ότι συνεισφέρει και δημιουργεί μια πραγματικότητα για την κινητικότητα και λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή συγκυριακά πρέπει να δούμε ότι υπάρχει και έλλειψη σε τέτοια προσόντα και πρέπει να προαγάγουμε αυτήν την κινητικότητα. Σήμερα ως εισηγήτρια θα ήθελα να λάβω τον λόγο και θέλω να το υπενθυμίσω αυτό για άλλη μια φορά στους συναδέρφους. Στην Επιτροπή Υγείας είμαι εισηγήτρια πλέον για μια σύνταξη γνωμοδότησης για αυτά τα θέματα και γι' αυτό σήμερα στρέφομαι σε εκείνα τα θέματα και θα περιοριστώ περιοριστώ σε αυτά που αφορούν τα επαγγέλματα του τομέα υγείας και τον τομέα υγείας γενικότερα. Χωρίς αμφιβολία η ασφάλεια των ασθενών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ως αγαθό και γι' αυτό ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης που προβλέπει και προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και οι γλωσσικές ε, αυτές ε, εξετάσεις είναι κάτι το οποίο καλοχαιρετίζουμε. Στρέφομαι στον συνάδελφο Μπούσο και συμφωνώ μαζί του όσον αφορά τις γλωσσικές αυτές δοκιμασίες ή εξετάσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτές οι εξετάσεις να μην γίνονται μετά την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, αλλά ταυτόχρονα, ώστε να εγγυόμαστε ότι επαρκούν αυτές οι γλωσσικές γνώσεις να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά αυτό το άτομο σε μια άλλη ξένη χώρα είναι σημαντικό με αυτόν τον τρόπο που θα έχει κάποιο επαφή με ένα τέτοιο άτομο να τον κατανοεί και να γίνεται κατανοητός. Έτσι είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το θέμα των γλωσσικών γνώσεων. Ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και για τη συνάδελφο Λεγκρή που το προανέφερε είναι σημαντικό και για μένα το θέμα των ελάχιστων επαγγελματικών απαιτήσεων ιδιαίτερα όσον αφορά νοσοκόμες και μαμές εργαζόμαστε σε αυτό το σώμα υπό το σύνθημα και την έννοια υπό την πολυμορφία ενωμένη, διαφορετική ο ένας από τον άλλον, αλλά ενωμένη σε μια κοινή Ευρώπη. Οι παραδόσεις, οι εκπαιδευτικές και σχολικές πρέπει τουλάχιστον να λαμβάνονται υπόψη. Να έχουμε μια ελάχιστη εναρμόνιση, ναι, αλλά πρέπει να προσέξουμε από την άλλη πλευρά να μην ισοπεδώσουμε οι ιδιομορφίες κάποιων κρατών μελών και αυτό δεν αφορά μόνο τη Γερμανία γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε δυσκολίες. Για μας είναι ένα πρόβλημα για παράδειγμα ότι προβλέπει αυτή η πρόταση η γενική σχολική εκπαίδευση για τις νοσοκόμες και μαμές να αυξάνεται από 10 σε 12 χρόνια. Και θα ήθελα να σας πω ότι μετά από τη συζήτηση που είχαμε την τελευταία φορά καταδείχθηκε σαφώς ότι αυτή η τριετής επαγγελματική απέτηση επαγγελματικής δηλαδή άσκησης του επαγγέλματος ως προϋπόθεση υπάρχουν χώρες που βρίσκονται στο διπλό σύστημα. Δηλαδή η προσυπολογίζεται σε αυτή την ε, δωδεκαετή ετη περίοδος και η επαγγελματική ε, αυτή άσκηση. Παράδειγμα 10 συν 2 χρόνια, 12 Τώρα όταν λέμε 10 χρόνια σχολική εκπαίδευση ή και κάποιο ισοδύναμο 2 επιπλέον χρόνια συν 3 χρόνια επαγγελματική εξάσκηση όμως το ισοδύναμο δεν είναι απόλυτα σαφές τι εννοεί και τι καλύπτει και ακριβώς ε, μας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα εμάς διότι σε εμάς στη Γερμανία ήθιστε και με 10 χρόνια σχολικής εκπαίδευσης και τριετή επαγγελματική κατάρτιση να μπορεί να γίνεται κάποια νοσοκόμα. Τώρα όμως στο ε, ευρωπαϊκό επίπεδο χρειαζόμαστε αυτούς τους ε, επαγγελματίες. Χρειαζόμαστε κατεπηγόντως κάθε νέα και νέο που είναι πρόθυμοι να αφοσιωθούν σε αυτόν τον τομέα. Και θέλω να το πω αυτό ελεύθερα. Δεν πιστεύω ότι οι προϋποθέσεις ε, είναι δεδομένες πρέπει κάποιος να έχει οπωσδήποτε το απολυτήριο, το σχολικό απολυτήριο. Όχι, πρέπει να έχει κυρίως το πάθος ε, και την ε, ας το πω έτσι έφεση και τάση να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορεί να είναι μόνο το σχολικό δίπλωμα ε, το κριτήριο. Πρέπει να είναι πρόθυμος και πρόθυμη να ασκήσει αυτό το επάγγελμα και να αφοσιωθεί σε αυτό. Δεν κάνω λόγο για την διοίκηση και τις ανώτερες βαθμίδες και κλίμακες αυτών των επαγγελμάτων. Κάνω λόγο για το επάγγελμα των νοσοκόμων που όχι μόνο στη Γερμανία έχει ανάγκες και δημιουργεί προβλήματα. Σε αυτό το σημείο θα να το πω. Θα ήταν σημαντικό να μπορούσαμε να βρούμε μια λύση που δεν θα είναι ισοπεδωτική και θα αφορά μόνο αριθμητικά κάποια έτη, θα αφορά περισσότερο την ουσία και σε σχέση με την προηγούμενη παρέμβαση θα πρέπει να δώσουμε σημασία στην ουσία όλων αυτών. Υπάρχει ένα παράρτημα το οποίο ρυθμίζει ίσως ε, τέτοια πράγματα να δουλέψουμε με ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά τη σχολική εκπαίδευση και να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα και στην ουσία. Εναρμονισμός όσον αφορά έναν ελάχιστο, ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμονισμού. Αυτό είναι σημαντικό για την αρχή της επικουρικότητας που πρέπει να είναι πάντα σεβαστή. Ολοκληρώνω και αναφέρω ως παράθεμα στην πρόταση ψηφίσματό μας. Ψηφίσματός μας. Λέει, επισημαίνει ότι τα επαγγέλματα αυτά και η ε, ε, κατάρτιση, η επαγγελματική κατάρτιση έχει μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα και η ε, χρονική διάρκεια θα πρέπει να προσυπολογίζεται που στα διπλά διτά τέτοια συστήματα προβλέπει σχολική εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτή ήταν η κοινή θέση της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής στο παρελθόν. Θα χαιρόμουν αν μπορούσαμε να βρούμε λοιπόν μια διέξοδο μέσω τέτοιου είδους προσεγγίσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να είστε σύντομοι στα σχόλιά σας, γιατί περνάει η ώρα. Και έχουμε ακόμη ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη μετά από αυτό. The next speaker will be and then... Η κυρία Γκέπχαρτ. Η κυρία Γκέπχαρτ, ευχαριστώ. Θα έλεγα, σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα μπροστά μας. Και γι' αυτό δεν μπορώ να υποσχεθώ θα είμαι τόσο σύντομη όσο επιθυμείτε εσείς κυρία Πρόεδρε διότι θα ήθελα να πω ότι εδώ εμπλέκονται θέματα αρχών και ως προηγούμενη συγγήτρια για αυτά τα θέματα θέλω να συνεισφέρω με την πραγματογνωμοσύνη μου. Να ξεκινήσω με ένα σημείο λοιπόν, το οποίο η κυρία Βερνιό στην αρχή προανέφερε. Αυτούς τους φόβους και δισταγμούς σε σχέση με τη συζήτηση για την οδηγία περί παροχής υπηρεσιών και την οδηγία περί αναγνώρισης επαγγελμάτων. Αυτά πρέπει να τα αποφύγουμε ως τρίβες. Για την παροχή υπηρεσιών είχαμε ως αρχή ότι η δισταγμοί και επιφυλάξεις ε, υπήρχαν και ήταν δικαιωμένοι λόγω των, ε, της, ε, των συστημάτων στα κράτη-μέλη. Με την τωρινή τώρα αναγνώριση των επαγγελματικών αυτών διπλωμάτων δεν συμβαίνει. Και έτσι θέλω να τραβήξω μια σαφή διαχωριστική γραμμή ότι εδώ πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό και δεν πρέπει να παραμείνουμε στην προηγούμενη συζήτηση. Και χρειάζεται εδώ πραγματικά αυτή την οδηγία να την επικαιροποιήσουμε, να την ενημερώσουμε διότι υπάρχουν πάρα πολλά, υπερβολικά πολλά εμπόδια για τους ανθρώπους, τους πολίτες να ασκούν τα επαγγέλματά τους ελεύθερα και απρόσκοπτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <coughs> όσον αφορά για παράδειγμα θέματα τα οποία δεν αφορούν την ποιότητα ή τα προσόντα αλλά αφορούν οι εθνικές, εθνικά αντανακλαστικά. Κάθε χώρα πιστεύει μέσα σε ένα περιορισμένο φάσμα ότι η δική της εκπαίδευση και κατάρτιση είναι η καλύτερη παγκόσμια και η άλλη κατάρτιση και εκπαίδευση των άλλων κρατών είναι υποδεέστερη. Λοιπόν, αυτό να το λάβουμε υπόψη Θέλω να αναφερθώ σε ένα σημείο που από την κυρία Μακλάκιν προηγούμενα, όταν ήταν εκείνη η συγγήτρια για μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, πάντα εδώ αναφερόταν και πρέπει εδώ να διαφωνήσω. Το πρόβλημα δεν είναι η ρύθμιση. Το πρόβλημα είναι η αμοιβαία αναγνώριση των ε, προσόντων. Η ρύθμιση είναι σίγουρα αναγκαία, ώστε τα προσόντα και η ποιότητα να διασφαλίζονται. Αν όλα τα απελευθερώσουμε μέσα σε ένα απόλυτα ελεύθερο πλαίσιο για τα επαγγέλματα θα έχουμε μια ολέθρια κατάσταση. Ένα απόλυτο χάος. Δεν μπορούμε να το θέλουμε αυτό. Απόλυτο όχι κάθετα λοιπόν στην απελευθέρωση. Δεν είναι η απελευθέρωση εκείνο που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε όμως κοινού κανόνες και διατάξεις πανενοσιακά, ευρωπαϊκά που να δημιουργούν ένα εναρμονισμένο πλαίσιο. Τώρα, για τη χρονική διάρκεια, να πω δύο λόγια για αυτό το θέμα. Στι πρώτε συζητήσει εδώ στην κοινοβουλευτική μα επιτροπή, όταν εθίγει και συζητήθηκε αυτό το θέμα, είχα πολλέ επιφυλάξει. Ήμουνα ιδιαίτερα σκεπτική και ειλικρινά πρέπει να πω ότι μείωσα αυτές τις, ε, τους δισταγμούς μου και την, ε, τις σκέψεις, ε, την επιφυλακτικότητά μου, διότι είπα πού βρίσκονται τα προβλήματα, αυτό να δούμε, πώς μπορούμε αυτά τα προβλήματα να τα αντιμετωπίσουμε και να τα μειώσουμε, να τα άρουμε. Σε αυτή την επικαιροποίηση δεν πρόκειται μόνο για επαγγέλματα στον τομέα της υγείας, αλλά και για πολλούς άλλους τομείς επαγγελματικά. Και πρόσφατα Ακούσαμε και για την περίπτωση του δασκάλου snowboard που δεν μπορούσε να ασκήσει το επάγγελμά του κάπου, μια και είναι καθηγητής δάσκαλος snowboard, μια και αποτελεί τμήμα του επαγγέλματος των δασκάλων του σκι και δεν του δίνουν το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα αυτό. Γιατί λοιπόν να μην μπορεί, μια και είναι ε, δάσκαλος του snowboard ε, αυτού του αθλήματος, γιατί να μην μπορεί να ασκήσει αυτό το επάγγελμα στο επιμέρους αυτό, ε, στην ειδίκευσή του εξειδικευμένα και όχι διαφορετικά. Αυτές είναι οι σκέψεις που με απασχόλησαν. Νέες ιδέες που πρέπει να μας εμπνέουν στην προσέγγιση αυτή. Να σκεφτούμε πώ μπορούμε θετικά στοιχεία να δούμε για μια νέα διαμόρφωση με θετικό πνεύμα και προσέγγιση για τέτοιου σε επαγγέλματα και επαγγελματική δραστηριότητα. Γι' αυτό με θετικό τρόπο πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, θετικότερο από ό,τι συνήθως. Τρίτο σημείο, το θέμα των νοσοκόμων και μαμών ακούσαμε πολλά και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Θα πρέπει να απευθύνω έκκληση στη Γερμανία και στους Γερμανούς βουλευτές ε, και ευρωβουλευτές. Εμείς θέλουμε μια Γερμανίδα νοσοκόμος να έχει τη δυνατότητα επαγγελματικά να δραστηριοποιείται και σε μια άλλη χώρα μέλος όταν πηγαίνει σε αυτήν και θέλει εκεί να εργαστεί. Και πρέπει να επανεξετάσουμε και να δούμε αν τα επαγγελματικά προσόντα μιας Γερμανίδας νοσοκόμας ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμα σήμερα, όσο έχει σήμερα η κατάσταση. Επ' αυτού πρέπει να συζητήσουμε. Η Γερμανία έχει την επιλογή. Θα έχει την επιλογή η Γερμανία. Θα μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε μία συμφωνία για τα επαγγελματικά προσόντα για 12 ετή σχολική εκπαίδευση. Δεν σημαίνει αυτό το απολυτήριο, έτσι. Σημαίνει τη σχολική εκπαίδευση, δηλαδή σχολική ε, εκπαίδευση. Έχουμε το διπλό, διτό σύστημα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση στη Γερμανία, ότι ένα τέτοιο διτό σύστημα ε, θα μπορούσε να ισχύει και να μην, να μην υπάρχει πρόβλημα. Ή η Γερμανία θα παραμείνει στο, ε, ε, στην κατάσταση ως ισχύει σήμερα και τότε θα βρίσκεται εκτός νυμφώνος. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ως Γερμανία ότι 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το περαιτέρω σύστημα που έχουν για, τις επαγγελματικές, την επαγγελματική αναγνώριση θα πρέπει να το περιορίσουν για να ε, ταιριάζει στα όσα συμβαίνουν και ισχύουν στη Γερμανία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αν στη Γερμανία έχουμε τόσες πολλές δυσκολίες τους νέους να τους προσελκύσουμε στο επάγγελμα της νοσοκόμου ή της μαμής, ε, τότε αυτό θα συναρτάται μάλλον με τους όρους και προϋποθέσεις για την αναγνώριση αυτών των επαγγελματών στη Γερμανία, για το τι ισχύει και πώς πληρώνονται αυτά τα επαγγέλματα. Ε, και γι' αυτό πρέπει να ξαναπροβληματιστούμε και να τα ξαναδούμε όλα αυτά. Δεν είμαι λοιπόν εδώ υπέρ του απολυτηρίου, σχολικού απολυτηρίου ως προϋπόθεση, αλλά να έχουμε ένα υψηλά ποιοτικό αναβαθμισμένο επίπεδο που να διασφαλίσει επαγγελματικά τα προσόντα αυτών των ατόμων. Να μην τα απορρίψουμε όλα λόγω κάποιων αβεβαιοτήτων ή κάποιων ανασφαλιών, να καθορίσουμε επακριβώς το τι θα ισχύει ώστε το διτό σύστημα σχολικό και επαγγελματικής κατάρτισης να, βρίσκει, να μπορεί να γίνεται αποδεκτό από πλευρά αυτής της οδηγίας. Να μην απορρίπτουμε όμως όλα τα άλλα επειδή δεν ταιριάζουν σε αυτό το σύστημα συλλήβδιν. Αυτά. Και επαρκούμε σε αυτά. Νομίζω αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα που ήθελα να καλύψω με την παρέμβασή μου. Θα έλεγα ότι τα άλλα σημεία σε άλλη συγκυρία θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε. Δεν ήθελα να μακρηγορήσω. Ευχαριστώ. Um, uh, um, Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, εσείς αν μπορείτε. Ναι, είχαμε τον Ανδρέα Σβάμπ, αλλά και δεν μπορούμε μετά να επεκτείνουμε περισσότερο. Εντάξει, ήθελα ουσιαστικά να ζητήσω τον λόγο για τις νοσοκόμες. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Γκέπαρτα να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Εγώ, εμένα με αφορούν τα άτομα, όχι το σύστημα. Μπορεί σίγουρα κανεί να συζητήσει για το γερμανικό σχολικό σύστημα και να ζητήσει θεμητά να βελτιωθεί. Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει είναι οι νέε γυναίκε να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν επαγγέλματα με τη σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι νέοι, οι άντρε νέοι μπορούν στο διτό αυτό σύστημα να το κάνουν. Οι νέε γυναίκε δεν θα είχαν τέτοια δυνατότητα σε σχέση με το διτό σύστημα δεσμεύονται με την επίσημη αναγνωρισμένη σχολική εκπαίδευση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η προσχολική εκπαίδευση μπορεί να ενταχθεί, προσυπολογίζεται στο διτό σύστημα. Όμως το τυπικό αυτό απολυτήριο ως κριτήριο δεν είναι εκείνο το οποίο πρέπει να μας κάνει να αναγνωρίζουμε ένα επάγγελμα ή όχι. Ε, τότε δεν σας κατανόησα καλά, λέει η ομιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά αναφέρθηκαν και γι' αυτό θα είμαι σύντομο. Πιστεύω για τη συζήτηση μεταξύ κυρία ε, Γκέπαρτ και κυρία Ρούιλε δείχνουν οι συζητήσει τίνο πρόκειται και σε αυτή την οδηγία. Όπω σε όλε τι οδηγίε που αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, βρισκόμαστε μπροστά στο πρόβλημα ότι αναμένουμε, προσδοκούμε κάποιε ικανότητε και δεξιότητε που όμως ε, δυστυχώς μόνο με κάποια διπλώματα ή πτυχία μπορούν να καλύπτονται. Δεν είναι εύκολο έργο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διατύπωση αυτών των προτάσεων και στη συζήτηση που έχουμε δεν είναι απλό θέμα να αποσαφινιστεί μεταξύ μας. Όμως πιστεύω ότι οπωσδήποτε πρέπει να θεωρήσουμε σημαντικό και παρακαλώ να γίνει αυτό το διτό σύστημα εκπαίδευσης κατάθεσης που δεν υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην το θεωρήσουμε κάτι χειρότερο αλλά απλώς κάτι διαφορετικό με κάποια ετερότητα, διαφορετικότητα. Και σε πολλά επιμέρους σημεία, και προαναφέρθηκε αυτό, για τους ε, νοσοκόμους δεν θέλω να μακρηγορήσω, πιστεύω ότι πρέπει να μεριμνήσουμε να υπάρχει ένα συμβατό σύστημα το οποίο θα ισχύει και για τις νοσοκόμες στη Γερμανία Πιστεύω ότι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω μπορούμε να τα καταφέρουμε, να επιλύσουμε τα πρόβλημα. Το δεύτερο σημείο θέλω να αναφέρω είναι το θέμα της εκπαίδευσης ε, ε, στα ιατρικά επαγγέλματα. Θα το ε, συντμίσουμε, θα το περικόψουμε κατά ένα έτος. Έχω αμφιβολίες. Θέλω να το ξανασκεφτούμε αυτό από πλευρά εισηγητών και να το ξανασυζητήσουμε την επόμενη φορά. Τρίτο σημείο αφορά την επιθυμία της κοιόδου εισηγήτριας Κωνσταν για την εξαίρεση για τους συμβολεογράφους για τους συμβολεογράφους ε, υπάρχει φυσικά και το ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών κρατικό λειτουργήμα μέσα σε μια κρατική δομή. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να εναρμονιστούν. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν νομολογίες ε, ευρωπαϊκών ε, δικαστηρίων κρατών μελών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Από το τέταρτο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω και είναι το τελευταίο στο οποίο αναφέρομαι πρόεδρε αφορά το Ευρωπαϊκό Επαγγελματικό Δίπλωμα ή πτυχίο. Θα πρέπει να είμαστε το λιγότερο γραφειοκρατικοί όσο περισσότερο γίνεται λειτουργικά να προσαρμοστούμε, να προσανατολιστούμε, να μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο πτυχίο ή δίπλωμα, όμως την πραγματική του ε, επίπτωση θα μπορούσε να την έχει μόνο όταν θα υπάρχει αυτόματη αναγνώριση ή για τις νοσοκόμες που αναφέραμε, το πρόβλημα δεν θα ε, υφίστατο με αυτόν τον τρόπο. Δεν ταιριάζει αυτόματα σε όλα τα επαγγέλματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχουν πολλά ε, προηγούμενα, προαπαιτούμενα που μπορούν να οδηγήσουν στην ε, ε, αναγνώριση αυτή και που θα απαιτούνται από πλευράς κάποιων των κρατών μελών. Τώρα, το κράτος υποδοχής ε, ή το κράτος αποστολέας, αν θα είναι εκείνο το οποίο θα ε, αναγνωρίζει τη δική του νομοθεσία επ' αυτόν, είναι κάτι το οποίο εκρεμεί. Θα πρέπει πραγματικά να δούμε το θέμα της απλούστευσης. Απλούστευση πρέπει να ισχύσει εδώ. Υπάρχουν και άλλα θέματα όπου πραγματικά δεν θα πρέπει να υπάρξουν υπερβολικές προ Αυτά είναι τα πιο σημαντικά νομίζω για να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο συνένεσης. Έτσι πρέπει να προσανατολιστούμε ώστε η οδηγία για τους εργαζόμενους να μπορεί να αποκτήσει σάρκα και οστά με θετικό τρόπο. speaker. Ευχαριστώ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επόμενη παρέμβαση. Παρακαλώ πολύ σύντομη να είστε γιατί έχουμε και ένα άλλο θέμα ακόμα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ναι, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομο, γιατί έχει περάσει και η ώρα. Είναι 6 και. Σε γενικέ γραμμέ ήταν πολύ καλή αντίδραση στην ε, πρόταση από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν βέβαια ζητήματα παγίδα που πρέπει να τα επεξεργαστούμε και δεν μα κάνει εντύπωση. Λίγα σημεία λοιπόν που μπορεί να σα βοηθήσουν στη μελλοντική σα συζήτηση. Πρώτον, όσον αφορά την επαγγελματική κάρτα. Εμείς ε, είμαστε ικανοποιημένοι με την γενική υποστήριξη του θέματος αυτού, όμως θέλουμε να τονίσουμε δύο ζητήματα. Πολύ συζήτηση για την προθεσμία. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε, και αυτή είναι μια προσωπική μου γνώμη, Πότε εκδίδεται η πρώτη επαγγελματική κάρτα στο πλαίσιο τη τρέχουσα επαγγελματική θητεία. Ναι ή όχι. Καλή, καλά είναι να μιλάμε για αρχέ και θεωρίε. Αλλά όταν άρχισε ο Επίτροπο Μπαρνιέ το ζήτημα αυτό, ε, κατόπιν αιτήματο του Κοινοβουλίου, δεν αποκλείω να πει πολύ ωραία, ωραίες οι συζητήσεις, αλλά πότε θα εκδοθεί η πρώτη κάρτα, γιατί έχουμε μια σειρά οδηγιών και έχουμε και τις εφαρμοστικές πράξεις. Απλώς σας ε, ε, διαβιβάζω αυτό το προσωπικό ε, μήνυμα. Όσον αφορά την ανάλυση κόστους και ωφέλου. Πολύ σωστό αλλά μπορούμε να έχουμε μια τέτοιου είδου ανάλυση χωρίς να συζητήσουμε το θέμα του τέλους επαγγελματικής κάρτας. Εγώ δεν βλέπω πώς μπορούμε να προχωρήσουμε δύσκολα τα πράγματα. Η ανάλυση αυτή χωρίς να τεθεί το ζήτημα του κόστου, μου φαίνεται περίπλοκο να γίνει. Επίσης, πολλή υποστήριξη για την ιδέα αυτή του κοινού πλαισίου κατάρτισης, άρθρο 49α, Πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στι τομεακέ οδηγίε. Επίση, θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε μια δεύτερη διάταξη, το 49β, ε, τα τεστ κοινή εκπαίδευση, ε, που δεν ε, ήταν αντικείμενο συζήτηση και πρέπει να συζητηθεί γιατί είναι μια πολύ απλούστερη λύση. Δεύτερο θέμα, άρθρο 59. Ο αριθμός των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, αν έχουμε απορρίθμιση ή όχι. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή τη Επιτροπή σα σε δύο θέματα. Πρώτον, στι αρχέ Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια εξωτερική μελέτη η οποία παρέχει νομική και οικονομική ανάλυση για το όλο θέμα του, ε, του, των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων και των σχετικών δραστηριοτήτων. Ε, έχει νόημα να του ρίξετε μια ματιά, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αρχές Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε. Δεύτερο ε, σημείο, θα το γνωρίζετε από τον τύπο, το, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο, αλλά ο, ο πρόεδρος Παρόσο έλαβε μία επιστολή όσον αφορά ε, την ανάπτυξη ε, από πλευράς κυβερνήσεων. Τι μπορούμε να κάνουμε. Το εξετάζουμε και εξετάζουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δύο ακόμα ζητήματα, ε, οι γλωσσικές δεξιότητες και το τι είναι σημαντικό για μας. Ο έλεγχο των γλωσσικών δεξιοτήτων ε, για του επαγγελματίε της υγείας είναι κοινή λογική, αλλά δεν θέλουμε μια γραφειοκρατία που κανείς δεν ξέρει ποιο κάνει τι. Είναι η αρμόδια αρχή ή είναι ο εργοδότης που πρέπει να το κάνει. Γιατί αν το κάνουν και οι δύο, σύμφωνα με τα διάφορα πρότυπα, είναι ανοησίε και συγγνώμη που το λέω έτσι χοντρά. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση για τις γλωσσικές δεξιότητες, ε, να την προσέξουμε, μην καταλήξουμε με περισσότερη γραφειοκρατία. Πρέπει να βρούμε μια λύση, Αποκινούμε το Κοινοβούλιο. Παρακολούθησα τη συζήτηση για τις Γερμανίδες ε, νοσο... Ε, νοσοκόμες. Έχουμε 8 αποφάσεις του δικαστηρίου από αυτού. 8 λένε ότι οι εθνικές απαιτήσει πρέπει να αρθούν και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει έτσι να προωθήσουμε τη συζήτηση. Να παραπενθεί και πάλι το θέμα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μου φαίνεται περίεργο λοιπόν που ε, θα αρχίσουμε πάλι να αποκλείουμε, να εξαιρούμε τους συμβολιογράφους και μετά θα αρχίσουμε πάλι με επίλυση διαφορών να σας πω την αλήθεια, δεν βλέπω το νόημα. Ίσως καλύτερα να πάμε περισσότερο προς την κατεύθυνση ε, μιας πιο ολοκληρωμένης ε, Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν θα πω σε πολλές πρακτικές λεπτομέρειες για την οδηγία αυτή, λέει η Πρόεδρος. Όμως πρέπει να τονίσω ότι η ακρόαση θα γίνει τέλη Απριλίου, 25 Απριλίου. 25 Απριλίου. Παρακαλώ να είστε παρόντες. Θα έχουμε λίγο χρόνο για τη στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών. Η Μαρία Ιριγκόιεν PRESIDENTA. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους γιατί έμειναν ε, ως αυτήν την ε, προκεχωρημένη ώρα του απογεύματος ε, για να συζητήσουν για ένα ε, ζήτημα το οποίο ήταν αντικείμενο πολύ έντονων συζητήσεων. Είναι το θέμα λοιπόν των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών. Δεν υπάρχει εσωτερική αγορά χωρίς καταναλωτές. Φέτος είναι η 20η επέτειος ε, από την ίδρυση της εσωτερικής αγοράς ε, που θα έπρεπε να ήταν κινητήριος μοχλός ευρωπαϊκής ανάπτυξης και κλειδί για την επίτευξη των στόχων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών συμπεριλαμβανομένης βέβαια της νομοθεσίας ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς η οποία εξελίχθηκε με ταχύτερο τρόπο. Το θετικό αποτέλεσμα της, εσωτερικής, της ενιαίας αγοράς βασίζεται σε μία εξασφαλισμένη και αυξημένη προστασία των καταναλωτών και πρέπει να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό γιατί οι καταναλωτές πολλές φορές στην καθημερινή του ζωή είναι βάλωτοι. Υπήρξαν καταγγελίε από του καταναλωτέ, κυρίω όσον αφορά τι αλλαγέ, τι αγορέ στο διαδίκτυο, τι τηλεπικοινωνίε, μεταφορέ, όπω επίση και τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυξάνονται αυτέ οι καταγγελίε. Οι περισσότερε από τι καταγγελίε αυτέ αναφέρουν ε, τιμολόγηση, συνθήκες ε, πώλησης, ε, καταχρηστικές ρήτρε, προβλήματα διαφήμισης κλπ. Και η κατάσταση αυτή πλήττει ιδιαίτερα τους καταναλωτές που είναι ευάλωτοι ή τέλο πάντων σε μια κατάσταση ευάλωτη και που χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία και μια συγκεκριμένη στρατηγική από πλευρά των αρχών. Αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή νομοθεσία ασχολείται με αυτό το θέμα των ευάλωτων καταναλωτών. Επικεντρώνεται σε ένα μόνο παράγοντα ευάλωτου χαρακτήρα. Και τώρα σε σχέση με την ε, ένα νέο ρυθμό για έναν ευάλωτο καταναλωτή. Έχει ήδη γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο προηγούμενα και υπάρχει ο κίνδυνο να υπάρξει η έννοια του ευάλωτου καταναλωτή που δεν θα έχει την αναγκαία ελαστικότητα να προσαρμόζεται στι ε, ε, διάφορε καταστάσει ευάλωτου χαρακτήρα για ένα τέτοιο στατικού χαρακτήρα ορισμό τα πολιτικά και νομοθετικά μέσα μέχρι αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκή κλίμακα τείνουν στο να επικεντρώνεται σε έναν παράγοντα, τον ευάλωτο χαρακτήρα ή την τροτότητα. Έτσι για πρώτη φορά εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το, την έννοια του ευάλωτου χαρακτήρα των καταναλωτών το 2005 σε σχέση με τις αθέμητες ε, πρακτικές των επιχειρήσεων σε σχέση με το συσχετισμό τους με τους καταναλωτές στην ενιαία εσωτερική αγορά. Με αυτή την εισαγωγή όσον αφορά την επιρροή που θα μπορούσε να ασκηθεί στα, στους καταναλωτές ε, που ε, δεν μπορούν να ασκήσουν ε, τις δικές τους αρμοδιότητες. Αυτό δεν κάλυπτε όμως άλλες πιθανές περιπτώσεις όπως την υγεία τους, την ε, η ηθική τους υπόσταση. Δυστυχώς ε, η οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται σε κάποιους ε, τομείς για τους οποίους υπάρχει ιδιαίτερα ευάλωτος χαρακτήρας και δεν υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση όσον αφορά αυτό το χαρακτήρα, όσον αφορά απλά την αναφορά στο σκεπτικό 34. 34. Υπάρχει και η ανάγκη της εξειδίκευσης όσον αφορά την σύναψη συμβάσεων όταν ο πολιτής ή ε, ο πάροχος ε, δεν ε, υλοποιεί τις υποχρεώσεις του και θα πρέπει αυτό να καθίσταται απόλυτα σαφές σε σχέση με τον καταναλωτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την πρότασή, του, ε, πρότασή της για τους καταναλωτές 2014-2020 θέλησε να βελτιώσει το θέμα της ενημέρωσης των καταναλωτών, παγιώνοντας τα δικαιώματά τους, διευρύνοντας τις δυνατότητες προσφυγής, καθώς επίσης και τι πρέπει να γίνεται σε διασυνοριακό επίπεδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια φιλόδοξη πρόταση που συμπεριλαμβάνει επιπλέον την ε, ένταξη και τον ε, ε, ε, αναγκών των ευάλωτου χαρακτήρα καταναλωτών, καθώς επίσης και τη σημασία που έχει να προαχθεί η κοινωνική τους ένταξη, ώστε να γίνουν αυτόνομοι εμπλεκόμενοι, στην, ε, εμπλεκόμενοι με αυτόνομο χαρακτήρα στην αγορά. Αυτή η δυνατότητα για τους καταναλωτές είναι απόλυτα ελλειπής όσον αφορά τους καταναλωτές με ευάλωτο χαρακτήρα. Η ενημέρωση και πληροφόρηση αυτής δεν υλοποιεί τις υποχρεώσεις αυτές έναντι αυτών των καταναλωτών. Θα πρέπει να λάβουμε την, ε, ε, το χαρακτήρα τον ευάλωτο χαρακτήρα των καταναλωτών, παιδιών, ανήλικων ή άλλων που δεν έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις πληροφορίες που τους διατίθενται και το τι πρέπει να κάνουν. Καθώς επίσης και τα κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ή τα αμόρφωτα ε, άτομα ή ε, με περιορισμένες ε, ικανότητες. Ιδιαίτερα στην περίπτωση διασυνοριακής αγοράς κατανάλωσης για αυτούς όλους τους λόγους θεωρώ ότι είναι αναγκαίο λοιπόν να δημιουργηθεί μια ε, στρατηγική ενίσχυση των ε, δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν στο νομοθετικό τους πλαίσιο συγκεκριμένα εξειδικευμένα μέτρα που θα στοχεύουν στο να εγγυώνται μια επαρκή προστασία που θα ξεπερνά τα στενά πλαίσια απλής πληροφόρησης ή ενημέρωσης ιδιαίτερα σε εκείνα τα επίπεδα όπου το επίπεδο ευάλωτου χαρακτήρα, ο ευάλωτος χαρακτήρα είναι έχει μεγαλύτερες διαστάσεις. Όπου τα μέσα λοιπόν αυτά έχουν αποκαλυφθεί ως μη επαρκή για τα άτομα ευάλωτου χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε σχέση με τους ε, ε, ε είναι αναγκαίο να προστατέψουμε ακριβώς τα άτομα που είναι πιο ευάλωτα παιδιά ε, όσον αφορά τη διαφήμιση προϊόντων ε, με, ε, που περιέχουν λέει χαμηλά λιπαρά ή, έχουν, ή όχι ζάχαρη πρέπει να βελτιωθούν οι επισητιστικές συνήθειες, οι διατροφικές συνήθειες και σε σχέση και με την μη τήρηση της νομοθεσίας, σε σχέση με καθυστέρηση ή ακύρωση όσον αφορά τη, κάποια ταξίδια, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αερογραμμές χαμηλού κόστους, πολλές φορές οδηγεί η ιδιώτες να βρίσκονται σε μια κατάσταση ιδιαίτερα ευάλωτη. Αυτό πολλαπλασιάζεται ε, εν δυνάμει όταν πρόκειται για άτομο με ειδικέ ανάγκες, ε, με αναπηρία. Οι μελέτες έχουν καταδείξει ότι κάποιοι ε, καταναλωτές πληρώνουν τριπλάσια ποσά από άλλους και τα κόμιστρα, οι ναύλοι δεν είναι μέσα σε ένα διάφανο πλαίσιο ώστε να μπορεί το άτομο αυτό να ενημερώνεται με το σωστότερο τρόπο. Και πέρα από το μη περιεχόμενο όσον αφορά τις, ε, τα κοινωνικά δίκτυα πολλές φορές ε, ε, αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά ιδιαίτερους κινδύνους λόγω της διαφήμισης, ιδιαίτερα όσον αφορά και την απελευθέρωση των κυριότερων αγορών δεν οδήγησαν σε μείωση γενική των τιμών αλλά σε μια πρόσθετη δυσκολία για αυτά τα άτομα να επιλέξουν το τι πρέπει να, γίνει, να κάνουν από πλευρά του για να προσαρμοστούν με τον καλύτερο τρόπο ως καταναλωτές. Έτσι τα άτομα που είναι πιο ευάλωτα μπορούν να βρουν δυσκολία ε, για να διαχειριστούν και να ε, χρησιμοποιήσουν τους υφιστάμενους ε, μηχανισμούς. Είτε επειδή δεν τους γνωρίζουν ή επειδή δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν με το σωστότερο τρόπο. Επιπλέον έχουμε και τον ευάλωτο χαρακτήρα της τρίτης ηλικίας, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών για τη σημασία που πρέπει να δίνεται για τα πρότυπα και προδιαγραφές για την ασφάλεια κάποιων προϊόντων θα πρέπει να, να προβλέπεται όχι μόνο η προβλεπόμενη χρήση αλλά και η μη ενδεδειγμένη χρήση. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικέ ανάγκε, με αναπηρίε όσον αφορά τον εναρμονισμό των ενδείξεων και την πρόσβαση στι πληροφορίε με ε, το πιο, τον πιο εύληπτο τρόπο και σχήμα για αυτά τα άτομα. Αυτή η στρατηγική πρέπει να αντανακλάται και για την ημερήσια διάταξη για την ατζέντα της δράσης για τους καταναλωτές 2014-2020. Και ολοκληρώνω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ ότι σε αυτό το στόχο θα πρέπει να εμπλέκονται όχι μόνο οι αρχές, οι κρατικές αρχές, αλλά και οι επιχειρήσεις και οι πάροχοι υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει το πιο διάφανο πλαίσιο συμβατικά που θα δημιουργείται για αυτά τα άτομα στην Ευρώπη. Και οι ενώσεις καταναλωτών που που έχουν ε, σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν για την προστασία αυτών των ανθρώπων. Και παρόλα αυτά επιτρέψτε μου για να ολοκληρώσω να επισημάνω ότι αυτή η εξειδικευμένη προστασία των ευάλωτων καταναλωτών δεν πρέπει να μεταφράζεται στη δημιουργία δύο επιπέδων διαφοροποιημένων μεταξύ του για την προστασία. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τι ε, ενισχυμένε αυτέ ε, δράσει υπέρ των δικαιωμάτων αυτών των ατόμων με μια α το πω έτσι συγκαταβατική αντιμετώπιση. Είναι αναγκαίε αυτέ οι δράσει και για την ανάπτυξη και για την προαγωγή τη ενιαίας εσωτερική αγορά. Ταυτόχρονα μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε την υλοποίηση μια πιο δυναμική ενιαίας εσωτερική αγορά, πιο ασφαλούς και πιο συνεκτική. Θα έχουμε την προθεσμία ε, που θα καταλήξει 24 Απριλίου, θα έχουμε τις τροπολογίες 8 Μαΐου, θα συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες, στις 30 Μαΐου θα ψηφίσουμε προς έγκριση την έκθεση. Θα ψηφίσουμε ψηφιστεί τον ε, Ιούνιο στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Αναμένω τα σχόλιά σας. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Άριας, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα όταν ε, έχουμε την, τον χρόνο που έχει προχωρήσει υπάρχουν, υπάρχουν και κάποιες αλλαγές εδώ εκπροσωπώ τον συνάδελφο Ζουινέν, ο οποίος ως κοιόδης εισηγητής είχε αναλάβει ρόλο σε αυτή την οδηγία και θέλει να βοηθήσει τη συνάδελφό μας κυρία Πέρες αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίες με τον καλύτερο τρόπο, με το πιο επικοδομητικό πνεύμα να την ε, ε, οδηγήσει προς έγκριση. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά της. Η έκθεση λοιπόν για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα, ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Διακομματικά από πλευρά των συντονιστών ε, έχει εγκριθεί, έχει τύχει συνένεση ε, και αυτό το κάνουμε. Όμως ταυτόχρονα πρέπει δυστυχώς να διαπιστώσω ότι τα κυριότερα θέματα δεν έχουν επιληθεί ακόμα και εξ ονόματος του συναδέφου Ζιβάν θέλω να πω ότι έχει την εντύπωση ότι το κυριότερο ζήτημα, δηλαδή για τα άτομα εκείνα τα οποία πρέπει να τύχουν προστασίας, δεν πρέπει αγνοώντας αυτά τα άτομα να αποφασίσουμε να ληφθούν κάποια μέτρα. Και δεν γίνεται κάτι τέτοιο να υιοθετηθεί με αυτόν τον τρόπο. Υπό το πρίσμα του συναδέφου Ζιβάν θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο κάθε καταναλωτής κατά τη διάρκεια του βίου του μπορεί να θεωρείται άτομο με ειδικές ανάγκες που πρέπει να προστατευτεί. Όμως εδώ τίθεται το ερώτημα ποιους συγκεκριμένους κανόνες μπορούμε να θεσπίσουμε. Ένας καταναλωτής όπως εσείς ή εγώ να μπορεί να πρέπει να τύχει ιδιαίτερης ειδική προστασίας θα μπορούσε να δει κανεί και να ξεκινήσει με το Consumer Empowerment. Υπάρχει μια μελέτη του 2011. Καταλήγει στο αποτέλεσμα ότι ε, δεν είναι η ε, αποσαφήνιση εκείνο το οποίο λείπει, αλλά η δυνατότητα τα στοιχεία της πληροφόρησης και ενημέρωσης να γίνουν απόλυτα κατανοητά από πλευράς των καταναλωτών. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να μην κινηθούμε σε μια κατεύθυνση που δεν επιθυμείται εσείς κυρία Πέρες. Βρίσκω ότι η έκθεση σε κάποια σημεία είναι ιδιαίτερα μονοβαρής. Στα σημεία 5 και 9 λέγεται ότι η οδηγία περί καταναλωτών δεν, δεν προβλέπει τίποτα ε, άλλο εκτός από το σημείο 34 για τα άτομα με ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα. Η απαγόρευση, για, παράδειγμα, α, της ε, διαφοροποίησης ή η απαγόρευση σε σχέση με κάποιες ε, τραπεζικές ε, συναλλαγές και εμβάσματα ότι δεν πρέπει να την χάνουν ιδιαίτερη επιβάρυνσης με ξεχωριστό τέλος και σε σχέση με τα δικαιώματα ανάκλησης όσον αφορά μία συναλλαγή, μία αγορά αν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το πρόβλημα είναι για πολλούς καταναλωτές ότι αυτές τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες δεν μπορούν πολλές φορές να τις κατανοήσουν σωστά τότε θα βρωθούμε στο σωστότερο επίπεδο. Αλλά τίθεται για μένα το ερώτημα ποια θα ήταν τα επαρκή ισοδύναμα μέτρα για να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα ως άξονα και πιστεύω ότι και η έκθεσή σας συνεισφέρει υπέρ αυτής της συζήτησης. Για κάποιους τομείς πρέπει κανείς να πει ότι εξαιρούνται από την οδηγία περί δικαιωμάτων καταναλωτών. Μπορούμε να σκεφτούμε λοιπόν κάποιες τροποποιήσεις για το ένα ή άλλο θέμα. Για το σημείο 15 θέλω να πω ότι αναφέρεται ότι η υπερβολική ψηφιοποίηση και για την διαμόρφωση ε, ε, ε, πιο ευνοϊκών τιμών δημιουργεί πρόβλημα για τους καταναλωτές που δεν μπορούν να υποφεληθούν από αυτές τις τιμές σε κάποιες χώρες δεν χρησιμοποιούν ε, τα άτομα της τρίτης γενεάς ε, τέτοιου είδους ε, προσφορές. Πρέπει να υπάρξουν κίνητρα. Η εντύπωσή μου είναι ότι στη Γερμανία το iPad είναι κάτι το οποίο δίνει δυνατότητες με την αλλαγή όσον αφορά τα πλήκτρα για παράδειγμα και όσον αφορά και την γενική μείωση των τιμών ως επιχείρημα θα ήθελα να διαφωνήσω ότι δεν υπήρξε τέτοια μείωση τιμών. Ο ανταγωνισμός όταν σε δίκαιο πλαίσιο διαμορφώνεται όταν σε ένα δίκαιο πλαίσιο ισχύει και διαμορφώνεται, συνεισφέρει από πλευρά του, ώστε η επιλογή των καταναλωτών να είναι μέσα σε ένα ευρύτερο και θετικότερο πλαίσιο και με θετικότερε πιο ευνοϊκέ τιμέ. Εύχομαι να μπορέσουμε να συζητήσουμε και θα είναι ενδιαφέρουσα η περίπτωση αυτή τη εξέταση αυτών των προτάσεων. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Τουρούνεν. Ε, Ευχαριστώ. Θα ξαναμιλήσω στα δανέζικα και γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, είναι έκθεση και πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση να λέμε ότι όχι μόνο συγκεκριμένες ομάδες είναι ευάλωτες, αλλά υπάρχουν και καταστάσεις ευάλωτες, που δημιουργούν αυτό τον ευάλωτο χαρακτήρα, που γίνονται ευάλωτοι οι άνθρωποι. Και οι ειδικοί τομεί ένα τον οποίων είμαστε ευάλωτοι. Τα παιδιά βέβαια είναι πάντα ευάλωτα όσον αφορά τις διαφημίσεις. Όμως, δεν θα πρέπει να αγνοούμε και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία, ε, διανοητικά προβλήματα που είναι και αυτοί οι άνθρωποι ευάλωτοι όσον αφορά τις διαφημίσεις και πωλήσει ε, κατοίκων επίσης. Είναι ευάλωτοι και σε αυτό το σύστημα. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξετάζουμε και καταστάσεις. Πολλοί από εμά είμαστε ευάλωτοι όταν είμαστε σε μια τράπεζα ή όταν ερχόμαστε σε επαφή με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ακόμα και καλά εκπαιδευμένοι άνθρωποι είναι ευάλωτοι. Και εγώ ίδια Πρέπει να παραδεχτώ ότι καμιά φορά βρίσκω δύσκολο να καταλάβω πραγματικά τι δέχομαι στην τράπεζα όταν είμαι σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω είναι σημαντικό να πούμε ότι καμιά φορά ο περίπλοκος χαρακτήρας κάποιων καταστάσεων ε, δυσκολεύει πολύ τα πράγματα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών λέει ότι όσον αφορά τις διάφορες πρακτικές που ακολουθούνται από επιχειρήσεις είναι δύσκολο να πει κανείς ποιος είναι ευάλωτος καταναλωτής και ποιος είναι ο μέσος καταναλωτής. Δύσκολο να προσαρμοστεί αυτός ο χαρακτηρισμός στην πραγματική ζωή. Και είναι σημαντικό αυτό να το συμπεριλάβουμε σε ταμιακή νομοθεσία. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι υπογραμμίζεται. Χρειαζόμαστε επίση μια γενική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των ευάλωτων καταναλωτών και όσον αφορά την τα δικαιώμα, ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά τους και ίσως καμιά φορά για την επιβολή απαγορεύσεων. Απαγόρευση όσον αφορά την έκθεση παιδιών σε κάποια είδη διαφήμισης ή το να αγοράζουν κάποια προϊόντα όπως προϊόντα καπνού και ενοπνευματόδη. Ήδη υπάρχουν τις απαγορεύσεις στην νομοθεσία. Και κάτι τελικό, γιατί δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας, είναι και το εξής. Συμφωνούμε με, το, με τις γενικές γραμμές του κειμένου θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε ίσως κάποιες αυστηρότερες προϋποθέσεις και απαιτήσει. Εγώ η ίδια ενδιαφέρομαι πολύ για τα παιδιά, για τους νέους, όσον αφορά τον τρόπο ζωής και όσον αφορά επιζήμια προϊόντα, όπως είναι τα προϊόντα καπνού και το ενόπνευμα. Είμαι κατάγομαι μια χώρα που είναι πολύ φιλελεύθερη σε αυτού του τομεί και δεν νομίζω ότι ήταν πολύ επιτυχή η πολιτική. Θα πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα το διαδίκτυο και τα iPads όταν τα παιδιά παίζουν παιχνίδια στο διαδίκτυο, οι γονείς καμιά φορά παίρνουν πολύ μεγάλο λογαριασμό διότι μπαίνουν μέσα μια φορά τα παιδιά και αγοράζουν παιχνίδια από το διαδίκτυο. Έξοχη λοιπόν η έκθεση και προσβλέπω και σε περαιτέρω συζήτηση μαζί σα. Ο κ. Σμιθ στα γρήγορα, λέει προέδρο, Ναι, υποθέτω ότι πρέπει να είμαι σύντομο. Είμαι φιλελεύθερο, οπότε τα σχόλιά μου θα είναι από αυτή την οπτική γωνία. Μ' αρέσει η ελευθερία της επιλογής. are... Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι από μόνοι τους μπορούν να λάβουν πολύ σκληρές αποφάσεις και να αποφασίζουν μόνοι τους. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για την έκθεση. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το θέμα και όπως είπε ο κύριος Βάμπ θα διεξαχθούν και διαφέρουσες συζητήσεις. Θα ήθελα όμως να πω ότι η προστασία των καταναλωτών είναι βεβαίως ζωτική σημασίας αλλά αυτό σημαίνει προστασία των καταναλωτών εν γέννη. Όλοι είμαστε ευάλωτοι σε κάποιες καταστάσεις. Εγώ αγόρασα την, ε, επένδυσα στην τράπεζα της Ιρλανδίας, Bank of Ireland εδώ και τρία λεπτά και έχασα μόνο 80% της επένδυσης έκτοτε. Είμαι ευάλωτος καταναλωτής. Ναι, εν αυτή τη ενία ίσως ήμουν ε, ηλίθιος. Αλλά θεώρησα ότι ήταν μια ηθική δέσμευση που είχα απέναντι στην Ιρλανδία. Τέλος πάντων, τέρμα τα αστιάκια θα πρέπει να θεσπίσουμε προστασία, κυρία μου. Σίγουρα αυτό. Εγώ είμαι υπέρ υψηλή προστασία των καταναλωτών στη χώρα μου. Ήμασταν στην πρώτη γραμμή προστασία των καταναλωτών επί πάρα πολλά χρόνια, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σαν, κάποιο, σαν άτομο έχεις δικές σου ευθύνες και αν αφαιρέσει κανείς ευθύνες από το άτομο αυτό θα είναι προβληματικό, τουλάχιστον όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Αμφιβάλλω για κάποιες ε, από τις προτάσεις σας, αλλά θα δούμε. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά, συμφωνώ με την Δανέζα συνάδελφό μου, τα παιδιά είναι βάλωτα και χρειάζονται κάποια προστασία, αλλά έχουν κάποια προστασία τουλάχιστον στη χώρα μου. Έχουν κάποια προστασία. Επίσης λέγω όμως ότι εγώ σαν πατέρας έχω κάποια ευθύνη για το τι κάνει ο γιος μου στο διαδίκτυο πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Τελευταίο όμως σχόλιο που αφορά τους ηλικιωμένου, όλο και περισσότερο γίνομαι ηλικιωμένο. και νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάποιες επιλογές και έχω έναν πεθερό που είναι 92 ετών. Είναι βάλωτος? Δεν το βλέπω. Είναι αρκετά καλός κάνει στο διαδίκτυο ότι τα στέλνει τα τραπεζικά του εμβάσματα. Χρειάζεται κάποια υποστήριξη βέβαια, αλλά τουλάχιστον στη χώρα μου το συζητήσαμε αυτό. Λέμε ότι οι ηλικιωμένοι λίγο πολύ θεωρούνται σαν μη πολίτε και υπάρχουν σοβαρές επικρίσεις επ' αυτού. Θα πρέπει να προσέξουμε και αυτόν τον τομέα. Σα ευχαριστώ όμω πολύ κυρία μου. Θα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση αλλά όπως ξέρετε είμαι φιλελεύθερος, άρα θα έχω κάποιες ε, τροπολογίες σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ για τα ενδιαφέροντα σχόλιά σας, λέει Πρόεδρος. Τελευταίος, ο Αρίας και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οι διερμηνείς ήταν πολύ υπομονετικοί. Θα προσπαθήσω να είμαι το δυνατόν πιο σύντομος, να ευχαριστήσω και να πω ότι από πλευρά ε, προ την εισηγήτρια κατανοώ πολύ καλά ποια είναι η πρόθεση αυτή τη ε, πρόταση που έχουμε στο τραπέζι μπροστά μα. Αυτό που χρειάζεται εδώ είναι πιστεύω να την καθορίσουμε εξειδικευμένα, να την αποσαφηνίσουμε πραγματικά ευάλωτη υπό του όρου που εγώ δίνω περισσότερο χρόνο στα αυτά τα θέματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευάλωτοι είμαστε όλοι, ούτω ή άλλω. Όλοι. Και είμαστε πάμπολοι και υπό αυτή την προπτική αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καθορίσουμε με τον καλύτερο τρόπο στην ορολογία τους όρους αυτής της πρότασης. Και εδώ θέλω να το τονίσω περισσότερο αυτό το θέμα. Η ιδέα είναι πολύ καλή, η πρόθεση είναι πολύ καλή, η πρωτοβουλία είναι πολύ καλή. Εγώ, Μαρία, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να απευθυνθώ σε σένα και να σου προτείνω δύο πράγματα. Το πρώτο, να σου πω ότι στην Ισπανία, η Ισπανία ήταν το μόνο κράτος που καταψήφισε τη νέα οδηγία σε σχέση με τα δικαιώματα καταναλωτών. Και Πιστεύω ότι σε σχέση με αυτή την τοποθέτηση με την Ισπανική κυβέρνηση θα πρέπει να πιστεί ότι πρέπει να αλλάξει η στάση στην ψηφοφορία. Και το δεύτερο, θα ήθελα να υπάρξει βοήθεια για να καθοριστεί καλύτερα αυτή η πρόταση που πιστεύω ότι είναι ήδη καλή. Ευχαριστώ. Lovely. Thank Υπέροχα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την υπομονή σας και ευχαριστώ και τους διερμηνείς να πω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι. Σας παρακαλώ κάντε ό,τι μπορείτε και σας ευχαριστώ για, αυτή την, ε, για αυτό το ενδιαφέρον απόγευμα. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλό σας βράδυ. You wanted to wind up. 30 uh, seconds.